Uh, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Right. Uh, can we um, settle down, please? I'm pleased there's lots of networking going on, but we have some. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε παρακαλώ γιατί έχουμε πολλά και σοβαρά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ας μην καθυστερούμε άλλο λοιπόν. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρώτη από τις δύο πλήρες ημέρες συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να σας πω ότι όπως πάντα αναμεταδίδονται και στο διαδίκτυο οι συνεδριάσεις μας. Οπότε να ζητήσω συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση ε, και να ε, σας πω ότι βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω το νέο μέλος Αρμένα Μπαναχίνο στην Επιτροπή μας, η Βαλτακίνο, που διαδέχεται τον Λουί που έχει γίνει πια αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Μάλτας. Και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αδημονία τη δική σας συμμετοχή και συμβολή. Ο κύριος Μασκά, ο πρωθυπουργός της ε, Μάλτα, επίσης ήταν διακεκριμένο και έγκριτο μέλος της ε, Επιτροπής μας. Οπότε η κυρία Μπέλα ε, έχει μπροστά της προκατόχους πολύ σημαντικούς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το λόγο που μου δίνετε. Ελπίζω και εγώ να ακολουθήσω τα βήματα των προκατόχων ε, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Κυβέρνησης της Μάλτα στην Επιτροπή και σας ευχαριστώ για τα θερμά λόγια και το καλωσόρισμα. Και ο κύριος Μοσκάτα ε, που είναι, ήταν και πρωθυπουργός της, Μάλτα και ο, της Μάλτας και ο κύριος Γκρέχ που έγινε τώρα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ε, σας μεταφέρουν θερμούς χαιρετισμούς. Ωραία. Μπορούμε τώρα να σας ε, ενημερώσουμε και για την ε, επιτυχή επίσκεψη που είχαμε στις αρχές Απριλίου στην Κροατία. Μάλιστα την έκθεση θα τη βρείτε και μεταφρασμένη σε πολλές γλώσσες από την ε, αποστολή αυτή. Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στη διάρκεια της επίσκεψης με τον αντιπρόεδρο τότε κύριο Μίμιτς, που στο μεταξύ έχει διοριστεί υποψήφιος επίτροπος για θέματα καταναλωτή. Και την επόμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, την Τρίτη, Τρίτη 4 Ιουνίου στις 9 το πρωί, 4 Ιουνίου 9.30 το πρωί, θα έχουμε την δημόσια κρόση για την επιβεβαίωση της, ε, του διορισμού του κυρίου Μίμιτς. Θα δούμε κατά πόσο είναι κατάλληλος για τα καθήκοντα του Επιτρόπου Καταναλωτή και ελπίζω να δώσετε όλοι το παρόν σε αυτή την ακρόαση με τον υποψήφιο Επιτροπό Μίμιτς, που επίσης θα αναμεταδοθεί στο ίντερνετ. Τα πρακτικά θα εγκριθούν μέχρι το τέλος συνεδρίες αν δεν υποβληθούν διορθώσεις. Επίσης, ε, αύριο θα έχουμε και ένα από τα καινούργια δελτία, τα ενημερωτικά. Προχωράμε στο πρώτο κυρίως θέμα της ημερήσης διάταξης. Πριν την ε, δημόσια κρόαση, που ενδιαφέρει πολλούς φαντάζομαι, πρόκειται για την ασφάλεια των προϊόντων και την επιτήρηση αγοράς. Προηγουμένως όμως έχουμε άλλα θέματα. Την ενημέρωση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, ε, τριμερού διαλόγου. Η πρώτη αφορά τι δημόσιε προμήθειε. Χθε το βράδυ με τον κύριο Ταραμπέλα δουλεύαμε μέχρι τι 9 το βράδυ. Για να μην νομίζετε ότι όλα είναι ρόδινα και έχουμε και εύκολη ζωή. Μέχρι τις 9 συζητούσα με τον κύριο Ταραμπέλα για τι διαπραγματεύσει τριμέρου διαλόγου. Θα του δώσω τώρα το λόγο για να μα ενημερώσει τι γίνεται με τι δημόσιε προμήθειε. Έχετε το λόγο κύριε Ταραμπέλα. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπω είπατε, όντω θα προσπαθήσω να ενημερώσω την Επιτροπή Ιστορική Αγορά για του δύο τελευταίου τριμερεί διαλόγου. 23 Μαΐου ο πρώτος και εχθές το βράδυ για την τομεακή οδηγία ο δεύτερος. Όπως συζητήσαμε τα τελευταία κομμάτια της γενικής οδηγίας, τα τελευταία κλάστερ και όπως είπα την ε, τομεακή, την ειδική για τους τομείς. Καταρχάς ε, για τη μεταβλητή 43, άρθρο 43 της οδηγίας, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να συμφωνήσουν ε, ως προς μια λύση, γιατί θα μπορούσαν οι αρχές να δώσουν ή μη την άδεια στους ε, αντισυμβαλωμένους να προβάλλουν μία εναλλακτική. Και αυτό ανεξαρτήτως. Όσον αφορά την προειδοποίηση, άρθρο 48 παράγραφος 1 για την ε, κατα... κατακύρωση της ε, σύμβασης, 30 ημέρες προθεσμία προβλέπονται για την κύρωση από την Επιτροπή αντί για 45 πιεστή στο Συμβούλιο. Όσον αφορά την τροποποίηση των συμβάσεων, άρθρο 72, κύριο ζήτημα διαφωνίας για την τροποποίηση των συμβάσεων ήταν παράγραφος 4 για τις ε, επουσιώδεις ή μη τροποποίησης, όπου το Συμβούλιο δεν ήθελε να δεχθεί την πρόταση του Κοινοβουλίου με έναν ε, κανόνα κατοφλίου και είτε ε, εναλλακτικά. Το Συμβούλιο ήθελε σωρευτικά τους δύο αυτούς, ε, τις δύο αυτές αρχές για να εξεταστεί αν είναι ουσιώδης η αλλαγή ή όχι. Έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο δέχθηκε να τροποποιήσει τον κανόνα de minimis για τις υπηρεσίες με 10% τροποποίηση για δε τις, αγοράς, τις αγορές έργων στο 15% όπως είχε προτείνει το Συμβούλιο. Άρα δείξαμε ε, μια κινητικότητα προς το Συμβούλιο, αλλά θέλουμε να επιβεβαιώσουμε και πάλι ότι αυτή οι τροποποιήσεις στην εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη στον ορισμό τους, ώστε να μην χρειάζεται να ξαναρχίσει μια νέα πρόταση δαπανηρή και επαχθής, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει και να δώσει περιθώριο σε καταχρήσεις και ουσιαστικές επιβαρύνσεις, κυρίως οικονομικές, των έργων η Επιτροπή της οποίας θα ήθελα να υπογραμμίσω τον θετικό ρόλο ως συνομοθέτης, που, έχει, που ως συνομοθέτης έχει δραματίσει μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, έκανε μια προσπάθεια να συμβάλλει συμβαστικές λύσεις, να κάνει προτάσεις όπου ήταν δύσκολο ε, η μία πλευρά να υιοθετήσει τις θέσεις της άλλης. Για το άρθρο 82 της τομεακής οδηγίας βλέπουμε το ίδιο ε, προβλέπονται όμως ακόμη πιο ευέλικτοι μηχανισμοί δεδομένης της σημασίας των συμβάσεων. Για το κλάστερ 9 έχουμε δεχθεί την ε, κατάργηση του άρθρου 84 με τον ενίο μηχανισμό ε, εποπτείας και θέλουμε αντίστοιχη προσέγγιση ως προς την εφαρμογή του monitoring, άρθρο 83. και ε, λέμε ότι για το Κοινοβούλιο η ατομική έκθεση του άρθρου 85 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τον υπεργολάβο και τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων για τις ε, διάφορες προτάσεις αναφορά τις εθνικές εκθέσεις, άρθρο 86, υποστηρίζει το Κοινοβούλιο τη φιλοσοφία της Επιτροπής για ετήσιες στατιστικές εκθέσεις, ενώ το Συμβούλιο φρονεί ότι θα πρέπει να προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν αρκεί το TLD για να δοθούν επαρκή στοιχεία. Επίσης, επιμένει το Κοινοβούλιο στην ε, αρχή κατακύρωσης για την επιμελητιακή βοήθεια και όχι στις επιχειρήσεις όπως ήθελε το Συμβούλιο. Επιμένουμε στη ε, χρήση του συστήματος EMI, άρθρο 88, κατά την ανάθεση των συμβάσεων για τις αγορές και αυτά βέβαια είναι όλα τα σημεία τα οποία ε, παρουσιάζουν στα οποία παρουσιάζονται διαφορετικέ ε, ε, απόψεις και θέσεις και για τα οποία οι τεχνικές ομάδες πλέον θα αναλάβουν την επεξεργασία. Εχθές, όπως είπα, είχαμε τα θέματα του τη τομεακή οδηγία για τα άρθρα 4 και 2 αποκλειστικά δικαιώματα, 4ε2 ε, 2 ε, δικαιώματα. Είπαμε ότι η αρχή ανάθεση θα έχει αποκλειστικά δικαιώματα ή ειδικά δικαιώματα, στα οποία για λόγου διαφάνεια θα εφαρμόζεται η οδηγία για τους αποκλεισμούς του άρθρου, των άρθρων 10, 27, 28. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν ως προς την ε, προσέγγιση που θα υιοθετηθεί για την έκθεση στον ανταγωνισμό της αναθέτουσας αρχής. Άρα έχουμε κοινότητα απόψεων ε, και γίνονται δεκτές αυτές τις προτάσεις της Επιτροπής. Επίσης, πιο συγκεκριμένα το Συμβούλιο δέχεται την προσέγγιση του Συμβουλίου που ιδιαίτερα για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με φιλοτελισμό, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες και με επιμελητιακές υπηρεσίες θέλει διαφορετική μεταχείριση. Αποκλείονται επίσης ορισμένα τμήματα δραστηριότητας που εκτίθενται στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή σε μια, που βρίσκεται σε διαδικασία απελευθέρωση σε κάποιο τομέα που είναι ακόμα κατακαιρματισμένη και με διαφορετική γεωμετρία ανάλογα με την χώρα. Άρθρο 45 ε, προσέγγιση διαρθρωμένη προτείνει το Κοινοβούλιο με την απαραίτητη διάρκεια για την απόσβεση της επενδύσεως και την διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων εξουσών αρχών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική τροπολογία για το Κοινοβούλιο, το πράγμα το οποίο όμω δεν δέχεται το Συμβούλιο. Τεχνική συζήτηση και επαναδιατύπωση μπορεί να γίνει, αλλά με διατήρηση των αρχών που σα εξέθεσα εδώ. Και για να ολοκληρώσω, η τάση που καταγράφει ο αρχικό τριμερή διάλογο επιβεβαιώνεται καλές προθέσεις και διαθέσεις εκ μέρους του Κοινοβουλίου, το ξέρατε ήδη, αλλά και εκ μέρους του Συμβουλίου και μια προσπάθεια να ε, συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, διαμεσολαβητής όπου δεν υπάρχουν ακόμα ε, συγκλήσεις απόψεων έρχεται να προτείνει εναλλακτικές θέσεις για τα utilities, για την έκθεση, για τα βασικά αγαθά, κύριε Πρόεδρε, πέραν κάποιων λεπτομεριών που πρέπει να διευθετήσει μια τεχνική ομάδα. Χτες αργά το βράδυ βρήκαμε κάποιες λύσεις κοινέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την έκθεση που μας κάνετε, που δείχνει την σχέση που έχουμε το Συμβούλιο, την εμπλοκή και τώρα φτάνουμε στα τελευταία πολιτικά ζητήματα. Δεδομένης της περιπλοκότητας του ζητήματος, μαζί με τον κύριο Ταραμπέλα κάναμε καλή πρόοδο. Γιατί όχι μόνο ασχοληθήκαμε με τις κλασικές προμήθειες, αλλά και αυτές που αφορούν τις υπηρεσίες κοινή ωφελίας τα Έχετε σχόλια ε, προς τον εισηγητή. Όχι. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα από πλευρά μου. Να... Και καλά νέα και κακά νέα έχουμε. Ε, τα καλά νέα είναι ότι σχεδόν έχουμε φτάσει συμφωνία με το Συμβούλιο και ξέρετε ποια είναι η βάση ε, της συμφωνίας για τα σκάφη ψυχής Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, δεν θα επανέλθω. Ε, ασχοληθήκαμε στις συμφωνίες για τις, με τις συμφωνίες για τις ε, εκτελεστικές και κατεξιδότηση πράξεις. Στάσαμε συμφωνία με το Συμβούλιο, αλλά έκτοτε, δυστυχώς κατά την απόψή μου, η Κομισιόν μας είπε ότι τελικά το Συμβούλιο δεν είναι έτοιμο να δεχτεί την πρόταση αυτή και μπλοκάρουν, μπλοκάρει την τοσχέ, το οποίο πρέπει να υιοθετηθεί με ομοφωνία. Πρέπει να αναθεωρηθεί λοιπόν το Κορεπέρα ακριβώς θα συζητήσει την Παρασκευή για αυτό το θέμα και η σύστασή μου προς την Επιτροπή είναι να περιμένουμε το αποτέλεσμα της συζήτησης του Κορεπέρ την Παρασκευή για να δούμε αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση και μετά θα έρθω σε επαφή με όλους τους κοιόδους εισηγητές για να δω εάν δέχονται το κείμενο αυτό που θα προκύψει από τις προπαρασκευαστικές συζητήσεις ε, προκύπτει ότι μάλλον το κείμενο θα είναι ε, αποδεκτό. Αν ναι, ε, θα προχωρήσουμε. Θα σας δώσω όμως το τελικό κείμενο προς έγκριση. Ε, επομένως θα ψηφίσουμε σήμερα το πρωί. Έχετε ερωτήσεις. Κυρία Ρούλα, βλέπω σηκώνει το χέρι. Τα θέματα των, της επιτροπολογίας και των εκτελεστικών πράξεων προσθέτουν βδομάδες στο διαπραγματευτικό μας πρόγραμμα. Σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε τα επαγγελματικά προσόντα και την αμοιβή αναγνώριση αυτών. Καλό είναι η Κομισιόν και το Συμβούλιο να κάτσουν μαζί μας για να ζητήσουμε, να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να το επιλύσουμε. δεν θα ξαναμιλήσω για εκτελεστικές πράξεις και κατευθυντικές πράξεις, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσουμε, θα ακούμε όλο το πρωί για αυτά. Θέλω να περάσουμε στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά και να καλέσω την Ashley Fox που είναι η συγγήτριά μας να παρουσιάσει το σημείο αυτό. Τον Ashley Fox. Ε, νομίζω ότι είναι καλό καλή συμφωνία, καλά τα όσα έχουμε επιτύχει. Έχουμε 140 τροπολογίες και θα ψηφίσουμε για το σημείο αυτό αύριο. Κύριε Φόξ, Ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και τους κοιόδες ηγητές ε, για τη συνεργασία τους. Ήταν πολύ ζωηρή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και καθόλου εύκολη. Γι' αυτό και θα ήθελα να επενέσω και να συγχαρώ τους συναδέλφους για τη λησαλέα προάσπιση των συμφερόντων και των ενδιαφερόντων τους. Είχαμε γύρω στις 400 τροπολογίες στην έκθεση. Δεν ξέρω <laughs> αν είναι ρεκόρ για, τροπολογ... για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίες. Φαίνεται να είναι. Προσπάθησα πάντως να συμπεριλάβω τις απόψεις όλων των πολιτικών ομάδων στην έκθεση και στις συμβαστικές τροπολογίες. Έχουμε 31 συμβαστικές τροπολογίες επιτάπητος και 17 από αυτές ε, έχουν συμφωνηθεί πλήρως. 14 έχουν απομείνει εκκρεμείς και για μερικές χρειάζονται κάποιες μικροαλλαγές. Σε ορισμένε ε, ίσω ε, χρειαστεί σημαντική αναδιατύπωση και μπορεί να μην κατορθώσουμε καν να καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν πρόκειται φυσικά να αναλύσω λεπτομεριακά και τις 31 ε, συμβαστικές τροπολογίες για να μην ε, μακρηγορήσουμε. Θα αναφερθώ σε ορισμένες. Στην 8. Φυσικά ξέρετε ποια είναι η θέση μου για τις ε, περιπτώσεις επί παραβάση. Ε, είναι η θέση που υποστηρίζει και η Άλντε. Είναι προτεραιότητα και των δύο ομάδων και στα πλαίσια του συνολικού πακέτου συμβιβασμού χαιρόμαστε για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σημειώσει πρόοδο στα θέματα περιπτώσεων ε, επιπαραβάση και ε, αυτό θα τον αναφέρει και η έκθεση. Βέβαια, πολλοί συνάδελφοι δεν συμφωνούν με το welcome, στο χαιρετίζει. Αν πούμε σημειώνει ή επισημαίνει, ίσω καταλήξουμε σε συμφωνία. Πάντω ε, επαναλαμβάνω, η τελική συμβαστική λύση αποτελεί τμήμα του πακέτου. Ε, το, η συμφωνία 8 είναι τμήμα του πακέτου. Τώρα για την 12 ε, θα ήθελα να υποστηρίξουμε την τροπολογία 193 του κ. Κρόιτσμαν που ζητά τη χρήση της τροπολογίας της, του κανονισμού IMI, του Συστήματος Πληροφόρησης εσωτερική αγορά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των Εθνικών Αριθμιστικών Αρχών. Σε ό,τι αφορά την συμβαστική τροπολογία 23, η αντιπρόταση του ΕΛΚ, κατά τη γνώμη μου, ίσως έχει ανεπιθύμητες συνέπειες. Γι' αυτό και υπέβαλα τις δικές μου αντιπροτάσεις που ελπίζω να τις ε, δεχτούν τα κόμματα. Δεν μπορούμε φυσικά να συμφωνήσουμε για οποιαδήποτε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να εμποδίσουμε τα κράτη-μέλη που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση του τομέα των τυχερών παιχνιδιών και σε ό,τι αφορά την τροπολογία 14 είναι πολύ σημαντική γιατί σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση των φορέων τυχερών παιχνιδών με το εθνικό δίκαιο, τονίζει ότι ε, και η εθνική νομοθεσία φυσικά θα πρέπει να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή, την ενωσιακή. Σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τροπολογία 30, ε, έλαβα υπόψη πολλές τροπολογίες ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση το δοτική συμβολή των φορέων τυχερών παιχνιδιών στα κράτη-μέλη στον αθλητισμό. Και χαίρομαι που τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να συμπεριλάβουν αυτή τη συμβολή και να αναγνωρίσουν και κάποια δικαιώματα στοιχημάτων για τα αθλήματα, για τον αθλητισμό, αλλά πιστεύω ότι και αυτό το θέμα θα πρέπει να εμπίπτει στην επικουρικότητα, όπω και άλλε επιτυχίε των διατάξεων για τα τυχερά παιχνίδια. Και εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την επικουρικότητα και στις συμβαστικέ τροπολογίες. Τέλος, ε, έγιναν κάποιες εκκλήσεις ε, να λάβουμε υπόψη κάποιες επικίνδυνες μορφές ε, στοιχημάτων ή τυχερών παιχνιδιών και να τις απογορεύσουμε πλήρως. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υποβάλουμε αξιολογική κρίση για το θέμα αυτό. Καλό θα ήταν να το παραπέμψουμε στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε σε συγκεκριμένε μορφέ τυχερών παιχνιδιών, γιατί δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για την επικίνδυνοτητά του. Και αναφέρω το σημείο αυτό στη συμβαστική τροπολογία 28. Ελπίζω ότι έχουμε σημαντική συμφωνία για πολλά θέματα όπω την επιβολή του ενωσιακού δικαίου, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών αριθμιστικών αρχών, την καταπολέμηση του, συστήμα, των παιχνιδιών και της ε, νομοποίηση ε, παράνομων εξόδων, καθώ και το, το, τα, τα εθνικά μητρώα αυτοαποκλεισμού. Εγώ έκανα σημαντικέ ε, προσπάθειες και με διαλεκτικό πνεύμα προσπάθησα να καταλήξω συμβαστικέ τροπολογίε με όλε τι πολιτικέ ομάδε και πιστεύω ότι ορίμασε η κατάσταση ώστε να δεχτούν όλες οι πολιτικές ομάδες το πακέτο των 31 τροπολογιών συμβαστικών. Και περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την άοκνη προσπάθεια που καταβάλατε στον τομέα αυτό και ε, σας ευχαριστώ για την διαπραγμάτευση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους σκιώδης ηγητές. Ο κύριος Φιέλνερ είναι από τους πιο ενθουσιώδες Εξωτερικού υποστηρικτέ ε, τη έκθεση αυτή τη ίδια πρωτοβουλία για τυχερά παιχνίδια. Θα τον ακούσουμε για αυτόν, αλλά πρώτα κυρία Κλάιντερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον Άσλι Φόξ, που πραγματικά με μεγάλη νυφαλιότητα και με πολύ ζεν συμπεριφορά προσέγγισε τις διαπραγματεύσεις. Γιατί πραγματικά ήταν σφοδρές συζητήσεις και πολύ φορτισμένες συναισθηματικά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει δεδηλωμένη βούληση να καταλήξουμε σε συμβαστικές ε, προτάσεις. Βέβαια, πολλοί επέκριναν ε, τις ε, συμβαστικές τροπολογίες για υπερβολικά επικείς και χαλαρές, όχι αρκετά αυστηρές, με πολλές αδυναμίες και χωλά σημεία, αλλά Νομίζω ότι είναι αυτονόητο όταν προσπαθούμε να δείξουμε διαλλακτικότητα και να κάνουμε υποχωρήσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί υπερβολικά. Βέβαια θα μπορούσαμε να τα είχαμε αφήσει όλα μέχρι την ψηφοφορία, αλλά εγώ προτιμώ την διαλλακτικότητα και την αναζήτηση συμβαστικής και ενιαίας πρότασης. Έγινε μια πολύ στην περιγραφή των διαπραγματεύσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων και πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε αρκετές συμβαστικές προτάσεις. Βέβαια, κάποιες συμβαστικές τροπολογίες ακόμη εκκρεμούν, μερικές για θέματα διατύπωσης και άλλες για πιο σοβαρά. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό ειδικά όταν πρόκειται για απλά θέματα διατύπωσης. Πίστευω ότι προσπαθήσαμε στις συμβαστικές τροπολογίες να συμβάσουμε κάποια αντιφατικές πολιτικές θέσεις. Η Συμβαστική Τροπολογία 8 χαιρετίζει την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά τις υποθέσεις επί παραβάση. Και νομίζω ότι αυτά ήταν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που είχαμε και τις σημαντικότερες προκλήσεις. Και ένα άλλο σημείο στο οποίο σημειώσαμε με σημαντική πρόοδο είναι η συμβαστική τροπολογία 23 και η διατύπωση των παράνομων και αθέμητων δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών. Πιστεύω ότι με συνέχιση των συζητήσεων θα καταλήξουμε και στις πιο δόκιμες ε, τροπολογίες εκεί που έχουν απομείνει κάποιες εκκρεμότητες. Επίσης, το θέμα της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο. Και εκεί υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στη διατύπωση. Θα πρέπει να βρούμε και εκεί την κατάλληλη διατύπωση για να συμφωνήσουμε. Αλλά φυσικά και η δική μου ομάδα είναι υπέρ της συμμόρφωσης ε, των κρατών μελών με το ενωσιακό δίκαιο. Είναι περισσότερο θέμα διατύπωση παρά θέμα αρχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τροπολογία για τις επικίνδυνες μορφές α, τυχερών παιχνιδιών, πιστεύω ότι και εκεί θα βρούμε τελικά μια συμφωνία, παραπέμποντας στο Συμβούλιο, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθεί ένας κοινό ορισμός για την ταξινόμηση των επικίνδυνων μορφών τυχερών παιχνιδιών. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ να παραπέμψουμε το θέμα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Να μην λάβουμε εμεί θέση, να μην χαρακτηρίσουμε συγκεκριμένα τυχερά παιχνίδια ως επικίνδυνα. Ε, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα σημεία, πολύ λεπτά και σημαντικά και για τη δική μας πολιτική ομάδα. Τώρα σε ό,τι αφορά άλλα σημεία στην συμβαστική τροπολογία 14 που αφορά και πάλι τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο. Επί της αρχής, επαναλαμβάνω, συμφωνούμε. Είμαστε υπέρ της τήρησης του ενωσιακού δικαίου, αλλά θα θέλαμε κάποια αναδιατύπωση που, που να αντανακλά καλύτερα τη δική μας ε, ερμηνεία περί συμμόρφωσης. Πιστεύω ότι με με αρκετή προσπάθεια και συνεργάσιμο πνεύμα θα σημειώσουμε πρόοδο και θα οριστικοποιήσουμε και τις υπόλοιπες συμβαστικές τροπολογίες. Παρέμεινα κάποιες ακρεμότητες για ε, το ευαίσθητο θέμα της, του χαρακτηρισμού των διαδικασιών καταγραφής και των ορίων που θεσπίζονται. Αλλά περιμένω στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων και ελπίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες ε, θα δείξουν πνεύμα συνεργασίας για την αναζήτηση συμβαστικών λύσεων. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά έχουμε κάποια ευελιξία και με τις προφορικές τροπολογίες. Κυρία Σαλντεμόζη. Ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Φόξ και τους ε, συναδέλφους για την προσπάθειά τους. Όντως είχαμε πολλές συναντήσεις ε, και συζητήσεις, αλλά Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε μάχη για τις πολιτικές μας απόψεις, αλλά φυσικά ταυτόχρονα έχουμε και συνεργάσιμο και διαλλακτικό πνεύμα και θέλουμε να καταλήξουμε συμβαστικέ συμβαστικές τροπολογίες για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση στο διαδίκτυο. Έχουν μείνει βέβαια κρεμή κάποια θέματα στην συμβαστική τροπολογία 6, 6α, στην 8, την 14, την 23, την 28, αλλά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση τελικά. Πολλές συζητήσεις γίνονται για το τι είδου ε, τυχερά παιχνίδια θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία από τις εκκρεμότητες είναι πώς θα συζητήσουμε και πώς θα ερμηνεύσουμε το ενωσιακό δίκαιο, την κοινοτική νομοθεσία. Και άσχετα από την έκβαση της συζήτησης, είναι σημαντικό να πούμε ότι για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι σημαντική η αρχή της επικουρικότητας. Δεν θέλουμε, τουλάχιστον προς το παρόν, μια πραγματική εσωτερική αγορά για τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, σε απευθεία σύνδεση, όπου ε, κανείς έχει κατάσταση σε, κέντρα σε μια χώρα και μπορεί πάντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει υπηρεσίες. Θα έχουμε βέβαια συμβαστικές τροπολογίες για να ε, πούμε ότι πρέπει να συμμορφώνεται μια χώρα με το κοινοτικό δίκαιο, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά το θέμα είναι ποιο είναι αυτό το κοινοτικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο και πώς το ερμηνεύουμε. Πάντως ε, υπάρχει ορατή πρόοδος και προσβλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων και φυσικά στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσω γερμανικά γιατί αλλιώς θα ξαφνιαστούν οι γερμανόφωνοι δημοσιογράφοι και άλλοι να ακούσουν να μιλάω αγγλικά. Είναι πολύ καλή δουλειά και θα ήθελα να παρακαλέσω, Κρίστη, Έχουμε ένα απλό πρόβλημα σχετικά. Έχουμε την αρχή της επικουρικότητας, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε. Δεν μπορεί κανείς να παραβιάσει την αρχή της επικουρικότητας, αυτό είναι σαφές. Όταν λοιπόν μιλούμε για ευρωπαϊκό δίκαιο, αυτό που λέμε είναι ότι σε ένα κράτος μέλος, εάν ξεκινήσει μια διαδικασία απολύσεων, τότε τηρούνται οι κανόνες που έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτός είναι άλλωστε και ο ορισμός του ευρωπαϊκού δικαίου. Όπου έχω μονοπόλιο, και το δέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν υπάρχει προσφυγή κατά του μονοπωλίου, παραμένουν τα πράγματα όσο έχουν, ενώ όταν προκύπτει μια διαδικασία απολύσεων, τότε τηρούνται οι κανόνες της νομολογίας που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε αυτό συμφωνούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφωνίες εδώ, διότι αυτό είναι και το νόημα των προτάσεών μας. Και έτσι 23 29 τροπολογίες αυτό εννοούν, ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν εάν βλέποντας σε παραδείγματι μία ε, ένα σχεδιασμό από πλευρά Φερρυπίν της γερμανικής εθνικής κατηγορίας, του, γερμανικού πρωτοθλήματος, εάν υπάρχει η πρόθεση για εισαγωγή τελών συμμετοχής, αποφασίζει το κράτος μέλος, εάν πρόκειται για δημόσιο αγαθό και αν θα το δεχθεί ή όχι. Δεν μπορεί να του το επιβάλλει κανεί δηλαδή. Και έτσι έχουμε και το συμβασμό μεταξύ διαφορετικών τοποθετήσεων. Εδώ έχετε δίκαιο, κυρία Σάλτε Μόζε, ότι δεν πρέπει να είναι υπερβολική η επιτρεπόμενη διαφήμιση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε υπερβολικές διαφημίσει, διότι ε, θα πρέπει και να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Και σε αυτό θα πρέπει να, να δώσουμε προσοχή. Αυτή πρέπει να είναι μια γενική γραμμή και με τις ε, προτάσει αυτέ, να μην περιοριστούμε μόνο σε αυτά που έχουμε πει η κυρία Μόζε και εγώ, αλλά προχωρήσουμε ένα παραπέρα και να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα, ώστε θεματοφύλακα των συνθήκων, να ε, προτείνει στα κρατη σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι συνθήκε ε, κάποιες διαφορετικές λύσεις. Αλλά εφόσον αυτό είναι ουσιώδες ε, πρόβλημα. Από την άλλη θα πρέπει να δεχθούμε ότι η Ευρώπη έχει και διαφορετικές νοοτροπίες και παραδόσεις σε κάθε χώρα και έτσι όταν υπάρχει διαδικασία διοδότησης θα πρέπει να λέμε ότι επιτρέπουμε να ε, λειτουργήσει αυτή η διαδικασία της αδειοδότησης με βάση τις αρχές της δημοκρατίας. Εάν υπάρχει μονοπόλιο, τότε με βάση το μονοπόλιο που έχει κανείς ορίσει στο κράτος του ή με βάση όποιους κανόνες έχει προβλέψει το ιστορικό δίκαιο για την αδειοδότηση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα, έχουμε, δηλαδή, ότι θα επιβάλλουμε για όλους ή πιο αυστηρούς ή πιο χαλαρούς κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να αφήσουμε ένα ευρύ περιθώριο και θέλω να έχουμε εγώ καλύτερη πλειοψηφία για την αρχική μου πρόταση πρόθεση για την έκθεση αυτή, να προχωρήσουμε με μια γερή πλειοψηφία πίσω μα και να στήσουμε από την Επιτροπή αυτή τη στάση ώστε με το φύλακα συνθήκων να κρατήσει. Και θα ήθελα επίση να προσθέσω, εάν υπάρχει θέμα απάτη δηλαδή... Ε, στη σήματος παιχνιδιών, εάν υπάρχει ζήτημα διαφθοράς σε, σε ε, σε αθλητές, τότε βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα γιατί το διαδικτυακό παιχνίδι δεν γνωρίζει σύνορα, και έτσι εάν υπάρχει ζήτημα αδειοδότησης θα πρέπει και να γνωρίζει ο καταναλωτής μια ένδειξη ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι εφόσον εμπλακεί σε αυτό είναι ε, ρυθμιζόμενο, έχει περάσει από τη διαδικασία της αδειοδότησης και ε, τηρείται κάποια εποπτεία πάνω σε αυτό. Και έτσι μπορεί να ξέρω ότι είναι πιο ασφαλής. Ευχαριστώ. κυρία Ρούλα. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ζητώντα συγγνώμη ταυτόχρονα, διότι ίσως δεν ήμουν δραστήρια ως και ηγετρία όσο θα περίμενε ίσως. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι η τρίτη έκθεση μέσα σε πέντε χρόνια που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ίδιο θέμα και διερωτώ με αν πράγματι χρειάζονται για το ίδιο θέμα τόσε πολλέ ε, εκθέσει. Εγώ προσωπικώ με την κυρία Μόζε και την έκθεση της, ε, και του κυρίου Κρότσμαν ε, νομίζω ότι είχαν λυθεί τα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει τόσο πολλά περισσότερα πράγματα, μια επιπλέον έκθεση. Ε, εξού και είμαι επιφυλακτική και γι' αυτό συνέβαλα πολύ λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Ο Πρόεδρος. Νομίζω για να είμαστε δίκαιοι προς την Επιτροπή και τον κύριο Φόξ, ότι μια ανακοίνωση επιτροπή ήταν εκεί, η οποία ε, οδήγησε στην ανάθεση του κύριο Φόξ εκθέσεω, η οποία ανακοίνωση Επιτροπή προκύπτει ω φυσικό αποτέλεσμα της εκθέσεω Σαλδεμόζε και Κρόιτσμαν. Είμαι βέβαιο ότι στην τρέχουσα θητεία δεν θα το ξαναδούμε το θέμα, αλλά ασφαλώ με το νέο κοινοβούλιο και νέα ομάδα και φρέσκη ομάδα, ίσω να του ξαναπροσχολήσετε. Δεν ξέρω αν ο κύριο Φόξ, η κυρία Σάλντε Μόζα ή ο κύριος πάνε έχουν όρεξη να ξανασχοληθούν με το θέμα. Ο κύριο Σαλντίνη, ο κύριος Φιέλνερ, Κονφεράτη, Σαμπέλα. Αλλά παρακαλώ να ε, επιταχύνουμε λίγο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Όσο πιο πολύ μυρίσει μάλιστα ο κύριο Κοφεράτη για το διαδικτυακό παιχνίδι, α έχει υπόψη ότι θα μιλήσει λιγότερο για τη δική του έκθεση. Κύριε Σαλβίνη, εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Είναι σημαντικό ο καταναλωτής να είναι πρώτος πριν την αγορά, γιατί ο καταναλωτής είναι και πολίτης. Ουσιαστικά τα τυχερά παιχνίδια ε, για πολλά κράτη είναι ένας τρόπος να βγάζουν λεφτά. Στην Ιταλία ειδικά ε, είναι μια αρρώστια. Ε, εμείς θα πρέπει να εστιάζουμε καταρχήν στα δικαιώματα του πολιτική και μετά στην αγορά. Ε, ως Λέγκα του Βορρά, σε ευχαριστώ πολύ για την ευαισθησία που δείξατε στα αιτήματά μας. Ε, περιέργως πώς, εμείς που είμαστε πίσω σε όλα ως Ιταλία, σε όλα τα θέματα, εδώ στη σχετική νομοθεσία είμαστε μπροστά. Θέλουμε λοιπόν να γίνουν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες, οι παραδόσεις των επιμέρους κρατών μελών. Η Ευρώπη τουλάχιστον σε αυτό τουλάχιστον τον τομέα ας ασχοληθεί και ας παρέμβει το λιγότερο δυνατό. Να κρατήσουμε ό,τι καλό υπάρχει στα κράτη-μέλη. Να μην αφαιρέσουμε όλα τα θετικά. Να, δεύτερον, να περιορίσουμε την παραπλανητική διαφήμιση, ε, να περιορίσουμε τις, ε, τα ξένα site, κυρίως από τρίτες χώρες, ε, παράνομα κτλ, κυρίως από την Ασία κτλ. για τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και στην χώρα μου και ειδικά στην πόλη μου πέσουμε κυρίως στο ίντερνετ Ε, και τα τυχερά παιχνίδια offline ε, δημιουργούν όχι μόνο οικονομικό πρόβλημα, αλλά και κοινωνικό, υγειονομικό θα έλεγα, γιατί οποιοδήποτε ας πούμε καφέ έχει και μία μηχανή, ένα κουλοχέρι, ξέρω, για να παίζει οποιοδήποτε. Επίσης, ε, οικονομικές κυρώσεις να επιβάλλουμε ε, σε ορισμένες χώρες όπως λέμε μάλλον, όπως η Ελλάδα επειδή δεν ανοίγουν λέει την αγορά τους στα τυχερά παιχνίδια. Αυτό είναι παλαβομάρα, διότι δεν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυτό το πρόβλημα τώρα ότι πρέπει να ανοίξει την αγορά στα τυχερά παιχνίδια, έχει να κάνω άλλα προβλήματα ας πούμε, ας αφήσουμε τα κράτη να κάνουν τη δουλειά τους. Πρώτα είναι τα δικαιώματα των πολιτών και μετά είναι η αγορά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υπομονή που δείξατε ε, καθώς τίνατε σε όλα τα αιτήματα ευήκονους. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλοί ομιλητές, παρακαλώ ε, ο καθένας για δύο λεπτά, όχι παραπάνω. Ποιος Φίλνερ. Κανένας δεν είναι ικανοποιημένος ε, με την κατάσταση, ούτε τα κρατημέλη, ούτε η operator, ούτε τα μονοπόλια. Και ας δούμε το κείμενο. Τι απάντηση δίνει στα προβλήματα. Η απάντηση είναι επικουρικότητα. Δεν χρειάζεται δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα θα έλεγα. Το μήνυμα είναι ότι με βάση την αρχή της επικουρικότητας τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν και να αποφασίσουν. Δηλαδή τα ίδια κράτη-μέλη είτε δεν θέλανε, είτε δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στο... στα τυχερά παιχνίδια αυτά. μας τους λέμε ασχοληθείτε τώρα. Ε, το πιο προβληματικό σημείο είναι το 8 για τις παρεμβάσεις. Εμείς ζητήσαμε κατά, κατά επανάληψη να υπάρξει πρόοδο στις παρεμβάσεις. Το κάνουμε από το 2007. Φυσικά Καλό είναι το ότι η Κομισιόν είπε ότι επιτέλους θέλει να κάνει κάτω. Και η κυρία Σαντελμόζε ε, έχει δίκιο που λέει ότι έχουμε νομική αβεβαιότητα. Και η απάντηση ποια είναι. Είτε να νομοθετήσουμε ή να ξεκαθαρίσει την κατάσταση το δικαστήριο. Ορισμένοι από εμά εδώ λένε δεν θέλουμε να τα ξεκαθαρίσει τα θέματα αυτά η νομοθεσία. Άρα τι σημαίνει, είναι σαν να λέμε ότι θα πρέπει να παρεύει το δικαστήριο. Επίσης, συμβασμοί 14 και 23. Δεν τους καταλαβαίνω. Είμαστε Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε αμοιβαία αναγνώριση. Αλλά αυτό είναι η αντίστροφη αμοιβαία αναγνώριση. Ε, όχι ότι αν είσαι νόμιμο σε μια χώρα, είσαι νόμιμος σε όλες. Είναι ότι αν είσαι παράνομος σε μία, είσαι παράνομος σε όλες. Επίσης, για την αναφορά στην ενωσιακή νομοθεσία. Μαλώσαμε για αυτό το θέμα, για να φύγει αυτή η αναφορά. Ειλικρινά σας λέω, το να λέμε ότι... Α, όταν λέμε ότι ας ενισχύσουμε τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη τα οποία δεν κάναν τίποτα και το να λέμε ότι δεν θέλουμε ενωσιακή νομοθεσία πουθενά είναι κρίμα, είναι χαμένη ευκαιρία, ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Γιατί ε, πολεμάμε για να κρατήσουμε το status quo. Ενώ η πραγματικότητα μας ξεπερνάει. Ο κόσμος θα παίζει τυχερά παιχνίδια online, θα έχουμε χάσει την ευκαιρία να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Τι να σας πω, εγώ έτσι το βλέπω. Σήμερα τουλάχιστον το πράγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για το συνεχές ενδιαφέρον και το ζήλο σας για τα θέματα αυτά. Ίσως στο επόμενο, στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία θα έχετε την ευκαιρία να αναλάβετε το θέμα και ως συγγετής. Ο κύριος Κοφεράτη, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δέχομαι αυτή την ιδέα των ε, επικοινωνούν δοχείων συγκοινωνούν των συγγνώμη δοχείων σε ό,τι αφορά το χρονομιλία. Ό,τι κερδίζουμε από εδώ το δίνουμε αλλού. Λοιπόν, τι θέλω να πω, κάτι γενικό. Κινδυνεύουμε να χάσουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Ε, αυτή η διάταξη, αυτό το νομοθέτημα, εν πάση περιπτώσει, είναι η συνέχεια άλλων. Τι θα ήταν ένα βήμα προ τα εμπρό, να φτάσουμε σε μια ενωσιακή νομοθεσία. Γιατί αν περιοριστούμε από ότι μου φαίνεται ότι προκύπτει από τους συμβασμούς ε, και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό για τη δουλειά που έκανε ο εισηγητή και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Αν περιοριστούμε όμω, όπω λένε οι συμβασμοί, στο να ασχοληθούμε με τη ρύθμιση των εθνικών συστημάτων και δεν έχουμε ένα σημείο ενοποιητικό, α πούμε, με ευρωπαϊκή προοπτική, θα χάσουμε μια ευκαιρία που δεν θα την ξαναβρούμε σύντομα. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα αυτό είναι. Δεν έχει επιληθεί ακόμα και ήθελα να το υπογραμμίσω. Κυρία Ζαβέλα, συγγνώμη που σας τριμώχνω την πρώτη φορά που θα λάβετε το λόγο στην ε, Επιτροπή, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε. Και συγχαίρω και τον εισηγητή για την πολύ ισορροπημένη του προσέγγιση, γιατί λαμβάνει υπόψη ε, την ανάγκη διαφύλαξη των κανόνων εσωτερική αγορά αφενό και την ε, υποχρέωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή να του επιβάλλει να ζητήσει την εφαρμογή τους ε, χωρίς να ξεχνά όμως και τις ευαισθησίες που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Έχω κάποιες επιφυλάξεις για ορισμένες τροπολογίες που προσπαθούν να λιώσουν την ισορροπία που με τόσο κόπο ε, επιτύχαμε. Οι συμβαστικέ τροπολογίες ε, αναφέρουν το γεγονός ότι παρά, παρόλο που τα τυχερά παιχνίδια είναι στο τομές. τα θέματα ε, της ελευθερίας αγοράς ε, ισχύουν και για αυτόν τον κλάδο και οποιασδήποτε παραβέσει θα πρέπει να κρίνονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και συμφωνούμε με την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις εκκρεμείς υποθέσεις επί παραβάση κατά των κρατών πελών που δεν συμμορφώνονται με τη συνθήκη. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εφαρμόζουν εθνικέ νομοθεσίε που αντιβαίνουν στην ενωσιακή νομοθεσία, γιατί κάτι τέτοιο επιτείνει την ε, έλλειψη ασφάλεια δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά ω προ την παρθενική μου ομιλία για το θέμα αυτό στην Επιτροπή σα. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Φόξ, για τα καταληκτικά σχόλια. Α μην ξεχνούμε και την αυριανή ψηφοφορία. Έχετε το λόγο κύριε Φόξ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον ε, Αλέξανδρο από τη Γραμματεία, τη Λίζη από το, την ομάδα και τη Μελίσα από το γραφείο για, την, για τις επανειλημμένες προσπάθειες ε, διατύπωσης και αναδιατύπωσης των συμβαστικών τροπολογιών. Και παρακαλώ στείλτε τις, τα τελικά σας σχόλια από των συμβαστικών τροπολογιών στο γραφείο μου μέχρι τις 12 το μεσημέρι για να δούμε σε πόσα σημεία έχουμε ριστικοποιήσει τη συμφωνία μας. Κύριε Φιέλνερ, ε, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και στην ομάδα σας. Αν ήταν ε, εκείνο και ο δισηγητής, θα, ήταν πολύ πιο εύκολο και το δικό μου έργο. Πάντως, ευχαριστώ και πάλι τους και ο μας για το συνεργάσιμο πνεύμα τους και θα επανέλθω αύριο στην ψηφοφορία για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τον ηγετικό ρόλο που ασκήσατε στο θέμα αυτό. Εκτιμούμε ιδιαίτερα στη θέση σας και όπως είπε η κυρία Ρούλε, το θέμα δεν είναι καθόλου πρωτοφανές, είναι πολύ παλιό, αλλά τουλάχιστον είμαστε από τις ίδιες επιτροπές που το κρατούν στην επικαιρότητα. Και μάλιστα έχουμε και ένα πολύ καλό ενημερωτικό σημείωμα της βιβλιοθήκης για το θέμα αυτό. Όποιοι ενδιαφέρεστε, ε, παρακαλώ ψάξτε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Δίνει μια πολύ καλή ανακεφαλαίωση του περίπλοκου αυτού θέματος. Έχουμε εδώ την κυρία Χόγκαν ως εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ε, δεν ε, ήθελε να λάβει το λόγο, αλλά παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα τεκτενόμενα. Περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση του κυρίου Κοφεράτη προς την Επιτροπή Βιομηχανίας Ενέργειας και Έρευνας. Ε, για την έκθεσή τους ότι αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CARS 2020 ε, για μια βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία. Πολύ σημαντική έκθεση και παρακαλώ όσους αποχωρούν να μην κάνουν φασαρία. Ο κύριος Καφεράτη έχει συντάξει μια γνωμοδότηση για το θέμα αυτό, θα μας την παρουσιάσει, μετά θα ακούσουμε τους συγκητές, τον κύριο Μπορισόφ, Χατζημαρκάκη, Ρούιλε, Ανθέλη, Είμαι και εγώ σκιώδης, ο κύριος Χέντερ απουσιάζει. Κύριε Κοφεράτη, εσείς πρώτα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, προκαταρτικά θέλω να κάνω δύο σχόλια πριν περάσω σε μια γρήγορη παρουσίαση της ε, ουσίας της πρότασης. Επικεντρώθηκα για προφανείς λόγους ε, σε θέματα που αφορούν την πρόταση ανακοίνωσης και που αγγίζουν πιο πολύ τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή μας, δηλαδή τους κανόνες εσωτερικής αγοράς και θέματα καταναλωτών. Το δεύτερο προκαταρτικό σχόλιο. Στο κείμενο θα βρείτε ένα κατάλογο, μια παρήθμιση των προβλημάτων, που δεν είναι εξαντλητικός όμως. Για λόγους χώρου καθαρά, δεν έβαλα μέσα προς το παρόν στο κείμενο που σας παρουσίασα κάποια σημεία τα οποία θα θεωρούσα χρήσιμο να τα εντάξουμε εκ των υστέρων μέσω των τροπολογιών. Και θα προσπαθήσω να σας πω ποια είναι αυτά τα σημεία που μπορούμε εκ των υστέρων να επανέλθουμε. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια πρόταση της Κομισιόν που θεωρώ ότι συνολικά είναι πολύ λογική. Έχει στοιχεία καινοτομία που μπορούμε να δεχτούμε περίπου 100%. Θέλει να εμπλουτίσει, θέλουμε να εμπλουτίσουμε μάλλον και να βελτιώσουμε όπου γίνεται την πρόταση που μας κάνει η Κομισιόν. Το πρώτο θέμα είναι να εξασφαλίσουμε, μια και εμείς ασχολούμαστε με την προστασία των καταναλωτών, ε, να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια στον τομέα των αυτοκινήτων. Όχι μόνο κατά διάρκεια της παραγωγής, αλλά και για τη δευτερογενή αγορά δηλαδή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ε, σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν ακριβείς ορισμοί σε ό,τι αφορά την αξία των αυτοκινήτων και τους τρόπους αγοράς ή πώλησης. Και αυτό είναι ζημία και για τον καταναλωτή από τη μία και προφανώς αποτελεί και στρέβλωση του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Δεύτερο και πολύ σημαντικό, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε πάντα σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές και την προστασία τους, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά την αλυσίδα πληροφόρησης για τα καύσιμα. Συχνά οι πληροφορίες που δίδονται δεν είναι αληθείς. Το αποτέλεσμα είναι ζημιά για τους καταναλωτές. Και από την άλλη, με, αυτές τις, ε, με αυτή την παραπληροφόρηση κρύβουμε τις ε, πραγματικές επιπτώσεις στο, επιπλα, ε, στο επι, περιβάλλον των καυσίμων που διατίθενται στην αγορά. Και προφανώς αυτός που το κάνει, αυτός που λέει ψέματα, το κάνει για να υποφεληθεί, αλλά και για να προωθήσει αυτοκίνητα που δεν πρέπει και η εγγνώση του ή η εναγνία του κάνει κακό και στο περιβάλλον. Επομένω, η σωστή πληροφόρηση, η διαφάνεια για τη σύνθεση των καυσίμων, για τι επιπτώσει του, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Επίση, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε επενδύσεις στην προηγουμένη τεχνολογία, γιατί το αυτοκίνητο είναι ένας όριμος τομέας με τρομερές όμως ικανότητες καινοτομίας αν δρούμε σε κάθε συνιστόσα του αυτοκινήτου. Σε κάθε εξάρτημα, σε κάθε στοιχείο του. Ε, υπάρχουν πιο ασφαλή αυτοκίνητα. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα αυτοκίνητα πιο ασφαλή, να καταναλώνουν λιγότερο, να έχουν θετική σχέση με το περιβάλλον στο οποίο κινούνται. Αν η έρευνα και η τεχνολογία στραφεί προς αυτήν την κατεύθυνση, θα το πετύχουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το προφίλ ενός αυτοκινήτου. Ένα αυτοκίνητο, αν είναι ωραίο, ε, φυσικά είναι, πάει καλύτερα στην ε, αγορά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα του προϊόντος. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως. Και εκεί πρέπει να δοθούν οι περισσότερες ε, επενδύσεις. Όχι μόνο το design, αλλά και την έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, που προωθούν και προάγουν την ασφάλεια και την άνεση. Επίσης, κάτι άλλο που τονίζει με ανησυχία η Κομισιόν πολύ σωστά είναι ότι πολλοί παραγωγοί επικεντρώνονται στις εξαγωγές. Γιατί η εσωτερική αγορά είναι, είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Υπάρχει μια πτώση, μια ύφεση. Εδώ, κρατάει εδώ και χρόνια αυτή η ύφεση. Και ευτυχώς σταμάτησε λιγάκι αυτή η ύφεση τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά έχουμε σαφώς μια πτώση της αγοράς αυτοκινήτου ε, σε, σε όλες τις χώρες σε διαφορετικούς βαθμούς. Και αυτή, αυτή η ύφεση, αυτή η πτώση είναι σημαντική. Επομένως, το θέμα είναι όχι μόνο πώς θα ενθαρρύνουμε τις εξαγωγές, αλλά πώς θα ξαναενισχύσουμε την εσωτερική ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να πρώτον να έχουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις των μακροοικονομικών πολιτικών, αλλά να δώσουμε και κίνητρα για την ανταλλαγή των παλιών αυτοκινήτων που σήμερα κυκλοφορούν ε, προάγοντας ε, αγορά, την αγορά αυτοκινήτων καινούριων που σέβονται αυτά που είπα πριν. Δηλαδή, θετική σχέση με το περιβάλλον και ασφαλή αυτοκίνητα. Μια πολιτική κινήτρων όμως, για να υπάρχει, θα πρέπει να συντονίζεται. Γιατί αν κάθε χώρα κάνει τα δικά της, μπορεί ενδεχομένως ε, οι προσπάθειές της να έχουν θετικά αποτελέσματα για τους δικούς τους πολίτες, αλλά αλλοιώνει το μηχανισμός σχέσεων και δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του τομέα. Δηλαδή θα πρέπει να αποφύγουμε τα κίνητρα αυτά, τα οποία είναι σίγουρα ένα πλεονέκτημα για τους καταναλωτές, αθέλητα, και βεβαίως θα ήταν ακόμα πιο σοβαρό αν αυτό γινόταν από πρόθεση για κερδοσκοπικούς σκοπούς, να οδηγήσει λοιπόν αυτή η ιστορία σε μια στρέβλωση, σε μια αλλίωση του ανταγωνισμού. Τελευταίο, όχι για την, ε, το λιγότερο σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι το θέμα της α, διαχείρισης των αδιαρθρώσεων. Ξέρετε ότι ο τομέας αντιμετωπίζει σοβαρότατες αλλαγές και θα αντιμετωπίσει. Αν ο τομέας αυτός στραφεί προς την παγκόσμια αγορά, αν όμως ε, παράλληλα ε, προωθήσει και την ασφάλεια κτλ, ε, θα τα πάει καλύτερα. Ο τομέας αυτός, το τομέα αυτό ε, δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες άτομα. Λογικό είναι να το στηρίξουμε αυτό το τομέα και με σχετική νομοθεσία. Επίσης, ε, να έχουμε υπόψη μας και την προστασία των εργαζομένων. Ε, να έχουμε κοινέ διατάξεις, ε, συγκλίνουσες, όχι διαφορετικές. ούτω ώστε να αποφύγουμε και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Σε ό,τι αφορά τώρα στοιχεία που δεν έχει ενσωματώσει η πρόταση, θέλω να αναφέρω επιγραμματικά τα στοιχεία αυτά, γιατί πιστεύω ότι μέσω των τροπολογιών μπορούμε να τα εντάξουμε αυτά τα στοιχεία στο κείμενο. Έχουμε ένα πρόβλημα με το σύστημα ετικετοθεσίας των ε, καυσίμων. Θυμάστε αυτά που είπα πριν. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα καύσιμα, να έχουμε σωστές πληροφορίες και πρέπει να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε από την ετικέτα τους. Ποια καύσιμα σέβονται τους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, και έχουν θετική επίπτωση στο περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να εναρμονίσουμε τα διάφορα συστήματα χρηματοδότησης αγοράς αυτοκινήτων. Προηγουμένως μιλούσα για κίνητρα η αγορά ενός αγαθού όπως το αυτοκίνητο συχνά υποβοηθείται από τις τράπεζες μέσω διαφόρων δανείων που δίνουν οι τράπεζες που είναι τελείως διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Εντάξει, δεν θα έχουμε το ίδιο σύστημα παντού, ε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία έτσι ενοποίησης, ομοιομορφίας και το μηχανισμό χρηματοδότησης αγοράς του αυτοκινήτου. Αυτό πρέπει να ενταχθεί στα κίνητρα. Και κάτι άλλο. Σημαντικό είναι το θέμα των επενδύσεων. Το είπα πριν. Είναι σημαντικό για το μέλλον του κλάδου. Το να χρησιμοποιηθούν προηγμένες τεχνολογίες. Θα πρέπει να συνδέσουμε την βιομηχανική πολιτική με, με τον ορίζοντα 2000 και τη σχετική χρηματοδότηση που προβλέπεται. 2020, συγγνώμη, και της, ε, τη χρηματοδότηση που προβλέπετε. Και θα πρέπει ε, να έχει θετική επίπτωση σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και βεβαίως να μην ξεχνάμε και αυτό το πολύ σημαντικό βιομηχανικό τομέα. Μην πω ότι είναι συνώνυμο με την ταυτότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τελευταίο που θέλω να πω είναι η οδική ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι μία από τα στοιχεία των αυτοκίνητων του μέλλοντος και οι κανόνες που διέπουν αυτή την ασφάλεια θα πρέπει κατά την άποψή μου να ενισχυθούν και να εναρμονιστούν. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 14η Ιουνίου. Έχουμε χρόνο λοιπόν για να ξανασυζητήσουμε. Είμαι στη διάθεσή σα. Φυσικά να λάβω υπόψη όλες τις απόψεις των σκιωδών και αυτές που θα εκφραστούν στη συζήτηση που θα ακούσω τη σημερινή, αλλά και τις υπόλοιπες που θα μου αποσταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ευχαριστώ για την πολύ καλή παρουσίασή σας και τις, προτάσεις Και τώρα, 10 λεπτά για ανταλλαγή απόψεων. Μια και έχουν προβλέψει τις ε, ψηφοφορίες στις 10 και 4, ο κύριος Μπόρισοφ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα δράσεως, γιατί αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Πρέπει να βελτιωθούν ε, οι ικανότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια από τις πιο μεγάλες βιομηχανίες. Με εκατομμύρια θέσεις εργασίας άμεσα εξαρτώμενες. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση του κυρίου Κοφεράτη, τον ευχαριστούμε πολύ, ιδιαίτερα για τις παραπλανητικές πληροφορίες και τη βασχετική παρατήρηση και ευχαριστούμε και για την παρατήρηση ότι χρειάζεται και διαδικασία αποτελεσματικής οδήγησης. Θα θέλαμε ωστόσο να βελτιώσουμε κάποιες ιδέες του κύριου Κοφεράτη και ιδιαίτερο στο θέμα της έρευνας και της καινοτομίας που θα θέλαμε να υποστηρίξουμε περισσότερο. Έχουμε μεγάλο επίπεδο δαπανών με 28 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 που απαιτείται να διατηρηθεί υψηλό προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Πρέπει να διευκολυνθεί λοιπόν αυτό. Και επίση, ως νομοθέτης, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να εξασφαλιστεί ένα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο για την πρόθεση της καινοτομία και την ε, οδική ασφάλεια βεβαίως θα περιλαμβάνει αυτό. Αυτή τη στιγμή στα θέματα της ασφάλειας είναι πρωτοπόροι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της Ευρώπης, αλλά πρέπει να διατηρήσουν αυτή την πρωτοπορία. Και αυτό θα αποτελέσει και την προσθεμένη αξία τη αυτοκινητοβιομηχανίας μα και στι ξένε αγορέ. Η αγοριστική δύναμη επίση του Ευρωπαίου πολίτη πρέπει να ενισχυθεί και να ενισχυθεί η δυνατότητα του Ευρωπαίου καταναλωτή να αγοράζει καθαρά και πιο ασφαλή αυτοκίνητα. Μια αγοραστική δύναμη που έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλέ χώρε και χρειάζεται υποστήριξη και με φορολογικά μέτρα και κίνητρα ώστε να δοθεί νέα στην κατανάλωση για τις εξαγωγές, που είναι πολύ σημαντική πηγή εισοδήματο και δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε καλή παρουσία στις ξένες αγορές και πρέπει να τη διατηρήσουμε, ενισχύοντας και τις δυνατότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πολλά άλλα πράγματα μπορούμε να πούμε, κυρίε και κύριοι. Εναλλακτικά καύσιμα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τεχνολογίες του μέλλοντος, όλα αυτά τα οποία μπορώ με τροπολογίες να υποστηρίξω στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς ευχαριστώ τον κύριο Κομφεράτη. Καταρχάς Νομίζω ότι θα χρειαστεί κάποιε τροπολογίε για να βελτιώσουμε το κείμενο. Και δεύτερον, πρέπει να επισημάνω ότι δεν μιλάμε για αμεληταία ποσά. Μιλάμε για 700 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, 12 εκατομμύρια θέσει εργασία, 180 εργοστάσια, ε, εγκαταστάσεις παραγωγής ανά την Ευρώπη. Πρόκειται για μια ε, για ένα τεράστια σημασία κλάδο της βιομηχανίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και με ιδιαίτερη προσοχή αλλά και με, πολιτικό, με σαφή πολιτική στόχευση να προχωρήσουμε και σε αυτό μου φαίνεται ότι είναι πολύ γενικόλογη η παρατήρηση για τα αναλλακτικά καύσιμα στο σημείο 2 και στο 7. Εγώ θα θέλαμε να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Χρόνια και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχουν γίνει σύνοδοι έχουν γίνει πρωτοβουλίε, έχουν, γίνει, έχουν διατυπωθεί ιδέε και προτάσει, αλλά αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Πέρσι 2.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα απολύθηκαν στη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, στη Γερμανία, και αυτό είναι ψίχουλα. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή ξέρετε που αποτυγχάνει ε, όλη αυτή η προσπάθεια απο, αποτυχάνει στο μέγεθο τη ε, πρίζα, τη δυνατότητα δηλαδή φόρτωση ενό αυτοκινήτου που αγόρασα στη Γερμανία όταν θα πάω στη Γαλλία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη εσωτερική αγορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε την απαρχίδα τη οικονομία και τη παραγωγή μα. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε πάνω σε μια πρίζα, σε ένα ρευματοδότη, ρευματολήπτη, τότε τι να σα πω και επιπλέον πρέπει να, περιοριστούμε, να περιορίσουμε αυτά τα, τα γενικόλεγα μπλα μπλα, τα, και στο συγγνώμη που χρησιμοποιώ την έκφραση. Έχω κάνει εγώ συνόδους κορυφή στο Βερολίνο για τα ηλεκτρικά ε, αυτοκίνητα, όπου είχαμε περισσότερους ομιλητές ε, στο βήμα, ε, από ό,τι κοινό μέσα στην αίθουσα. Είχαμε υπουργού, είχαμε ειδικού, είχαμε εκπρόσωπου βιομηχανία και πολύ λίγο κοινό. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, κύριε Κοφεράτη, για να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ανταλλαγή όπου υπάρχουν ζητήματα, όπου μπορούμε να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη, παραδείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περάσουν ε, τα δημόσια οχήματα που χρησιμοποιούν με τα full pack στο ε, ηλεκτρικό σύστημα. Αυτό είναι το ένα. Επίσης, όταν έχουμε να κάνουμε με ανταλλακτικά και με, ε, όχι, και με τμήματα ε, που έχουν να κάνουν με την ισοστάθμιση και τη ρύθμιση του αυτοκινήτου. Εδώ έχουμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ε, εμπόδια στην αγορά, προσκόμματα στην εσωτερική αγορά. Ο κύριος Ζώνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας το επιβεβαιώσει. Η πώληση ανταλλακτικών και άλλων εξαρτημάτων ε, έχει καταστεί αδύνατη ουσιαστικά από το ένα κράτο στο άλλο. Και στη Γαλλία και την Ιταλία ιδιαίτερω εντοπίζεται το πρόβλημα αυτό, γιατί οι εθνικέ διατάξει είναι τέτοιε, απεριόριστα εισάγονται, οι οποίε περιορίζουν ε, αυτή την, ανταλλαγή, αυτή την πώληση μέσα στην αγορά των ανταλλακτικών. Οι Μαζεράτη, η φίατ ε, έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποκλείσουν την διάθεση στην αγορά εναλλακτικών ανταλλακτικών. Λοιπόν, εάν αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε να διαμορφώσουμε, κυρίε και κύριοι, εάν η εσωτερική αγορά με διάφορα ε, λεπτομερεί ρυθμίσει μπορεί και εθνικέ ε, νομοθεσίε μπορεί να ε, καταστρέφεται από τα κράτη-μέλη, ε, νομίζω ότι πλέον δεν έχουμε εσωτερική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρόπο αποφασιστικό αυτέ τι διατάξει σε επίπεδο Γαλλία και Ιταλία ιδιαίτερω όπω είπα. Ασφαλώ και νομικά υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά ό,τι και να κάνουμε με τα νομικίστικα ε, δεν ε, βγάζουμε άκρη. Γι' αυτό παρακαλώ και ο πρόεδρο μα να με μεριμνήσει ειδικά για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή τη Εσωτερική Αγορά να ανασκουμποθεί και να αναλάβει αποφασιστική δράση Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε. Ναι και δεν έχουμε χρόνο, πρόεδρε, ας μην πω τίποτα. Θα ήθελα κι εγώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, γιατί είμαι και σκιώδης ηγητής, όπως είπα. Καταρχήν, είχα την τιμή να, να λαμβάνω μέρος στο στην πρώτη ομάδα υψηλού επίπεδου για το ΚΑΡΣΑ, που συστήθηκε το 2005. Και ο Φιλίπ Ζαν τον οποίο καλωσορίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν τότε εκεί και ήμουν ο μόνος ευρωβουλευτής που συμμετείχε σε αυτήν την ομάδα υψηλού μαζί με τον κύριο Βαν Λάγκε. Και ομολογώ ότι λυπάμαι για την απόφαση της διάσκεψης των προέδρων ε, των πολιτικών ομάδων να αποκλείσει τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών στην ε, χάραξη αυτών και κατάρτιση αυτών των σημαντικών εγγράφων εργασία. Τώρα η ομάδα εργασία ε, αποτελείται από εννέα εκπροσώπου των κρατών μελών και αυτά επιτρόπου. Δηλαδή, οι εταίροι μα στη συναπόφαση λαμβάνουν ενεργό μέρο στη συζήτηση μαζί με πολλού ενδιαφερομένου και εκπροσώπου αυτοκινητοβιομηχανία ε, και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Νομίζω ότι είναι κρίμα να μην συμμετέχουν οι ευρωβουλευτέ σε αυτό, σε αυτή την προσπάθεια. Και παρακαλώ να το ε, αναφέρεται και στις πολιτικές ομάδε ομάδες για να, γίνουν κάποια διαβήματα. Και άλλο συνάδελφος συμμετείχε ε, στο, στη πρωτοβουλία για το ΚΑΡΣ 21 πριν αποκλειστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι σε αυτό το περίπλοκο κλάδο θα πρέπει να καταλάβουμε τη δυναμική και να μελετήσουμε ε, τις δυνάμεις που αναπτύσσονται εκεί. Και μάλιστα είμαι μηχανικός, 20 χρόνια εργάστηκα στην αυτοκινητοβιομηχανία Έχω αρκετές γνώσεις για το θέμα. Θα είμαι σύντομος, γιατί θα πρέπει να περάσουμε και στην ψηφοφορία σε λίγο. Αλλά θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Χατζημαρκάκη για τα θέματα της εσωτερικής αγοράς. Και ο κύριος Κοφεράτη μας παρουσίασε το θέμα πολύ σωστά υπό το πρίσμα του καταναλωτή. Το θέμα της έγκρισης τύπου, για το οποίο είμαστε ε, αρμόδιοι, και το πώς λειτουργεί, πώς συνδυάζεται με το θέμα των ανταλλακτικών και μάλιστα ο κύριος Χατζημαρκάκης ε, αυτή τη στιγμή μιλάει με το διπλανό του. Συμφωνώ μαζί του πάντως. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλούς φιλόδοξους νέους στόχους ότι αφορά τη διεθνή νομοθεσία που ε, αποκτά όλο και ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια και των ε, διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τις Ηνωμένες Τώρα, σε ό,τι αφορά τη, διεθνή νομοθεσία, θα ήθελα να πω ότι πήγαμε στη Γενέβη, στα Ηνωμένα Έθνη, για να παρακολουθήσουμε τις συζητήσεις ακριβώς για τον κανονισμό που αφορά τα, την αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαστε η μόνη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μόνη επιτροπή που ε, ενδιαφέρεται και παρακολουθεί τις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα αυτά και χαίρομαι και για το ενδιαφέρον που έδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεσή μας. Επίσης, να σας επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή μιλά συγκεκριμένα για τις εφαρμοστικές διατάξεις πολλών κανονισμών, περίπλοκων κανονισμών για τα οχήματα και φυσικά θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων αυτών των εφαρμοστικών ε, νομοθετημάτων και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό και τις οικονομικές επιπτώσεις των εφαρμοστικών διατάξεων και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ότι οι κατασκευαστές μικρών αυτοχημάτων, οι μικροί κατασκευαστές μάλλον, να έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση στην αγορά και με επιτυχία παρακολουθήσαμε το άνοιγμα των αγορών στον τομέα αυτό. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει και τις διατάξεις εποπτείας της ε, αγοράς ό,τι αφορά την ε, έγκριση τύπου οχημάτων. Μάλιστα τώρα θα εξετάσουμε και τις νέες προτάσεις για την εποπτεία της αγοράς και θα πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις το θέμα του αυτού με τα οχήματα και την έγκριση τύπου. Πολλέ πτυχέ εσωτερική αγορά θα πρέπει να προσθεθούν στη γνωμοδότηση. Βέβαια, ο κύριο ε, Κοφεράτη περιορίζεται από τις από τους κανόνες που ισχύουν για την έκταση των γνωμοδοτήσεων, το μήκος τους. Πάντως χαίρομαι για την γνωμοδότηση αυτή και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει και μία μελέτη για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ένα θέμα που επισήμανε και ο κύριος Κοφέρα στην γνωμοδότησή του. Άλλωστε έχουμε και τη γνωμοδότηση για το καθεστώς δοκιμών των οχημάτων. Εκεί ε, θα ρίναμε ρητά τα κράτη-μέλη ώστε Στι αιτήσει ε, διαδικασίε, στου αιτήσιου ελέγχου, να λαμβάνεται υπόψη και χιλιομετρικέ αποστάσει που διανύουν τα αυτοκίνητα. Και ιδιαίτερα για τα μεταχειρισμένα να γίνουν κάποιε προσαρμογέ για να μην βγαίνουν χαμένοι σε τελική ανάλυση οι καταναλωτέ. Πάντω, ε, προσβλέπω σε πολύ αγαστή συνεργασία με τον κύριο Κοφεράτη για την γνωμοδότηση. Δεν ξέρω, Φίλιπ, ε, θέλει πολύ σύντομα να λάβει το λόγο ή αργότερα αργότερα. Πολύ ωραία και ευχαριστώ πάντως που ήρθατε. Κύριε Κοφεράτη, θέλετε το λόγο για κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ουσιαστικά επιχειρήματα που ακούστηκαν από τους συναδέλφους. Ε, θα τα λάβω υπόψη μου. Φυσικά κάποια από αυτά τα σημεία θα προκαλέσουν πολύ έντονες συζητήσεις προφανώς, κυρίως αυτό που αφορά το, μέσο, το μέλλον, είναι καινοτομία, αλλαγή του προϊόντος, φερειπίν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ευχαριστώ φυσικά τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Θα τις χρησιμοποιήσω γράφοντας τις δικές μου τροπολογίες. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, επίσης Πρόεδρε, για το πώς συντάσσονται αυτά τα κείμενα. Ε, χρειάζεται να εμπλέκεται άμεσα το Κοινοβούλιο. Ε, για κάποια κείμενα έχει γίνει αυτό. Έχουν εμπλακεί οι ευρωβουλευτές. Εδώ τώρα μιλάμε για το αυτοκίνητο, για την πιο σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας τον πλούτο που παράγεται από τα αυτοκίνητα. Όταν αποφασίζουμε λοιπόν οπουδήποτε θέματα για αυτοκίνητα, νομίζω ότι είναι αναγκαία η παρουσία μας. Καλό θα ήταν και για την Κομισιόν αυτό. Καλό θα ήταν να ξέρει εκ των προτέρων ποια είναι η άποψη των Ευρωβουλευτών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τη δική μου πολιτική ομάδα, λοιπόν, ε, θα υποστηρίξω την θέση που υποστηρίξατε κι εσείς ό,τι αφορά την εμπλοκή του Κοινοβουλίου στις εργασίες. Πολύ ωραία. Σα παρακαλώ λίγο ησυχία για να κάνουμε τα... τις Έχουμε και αύριο βέβαια ψηφοφορίε, σα το υπενθυμίζω. Απλώ ε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα πριν από την ακρόαση. Ένα θέμα ουσία έχουμε να ψηφίσουμε. Αντώνιο Κορέα κάμπο σχέδιο γνωμοδότηση για την έρευνη λειτουργία τη Ιστορικής αγορά ενέργειας. Κύριε Κάμπος, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι. Ψηφοφορία λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες. Ε, αν, όχι, αν δεν έχετε κάρτες ε, θα ψηφίσουμε δυνατά σας βέβαια, αλλά καλώς. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 1. Η 1 έχει αποσυρθεί. Η συμβαστική 1 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται προφανώς. 7. Πιατικά, έναν. σημειώνουμε. Ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 του εισηγητή εγκρίνεται 2 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 13 του εισηγητή αρχή ψηφορία υπέρ, κατά, πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται. 14. Κορέα Δεκάμπος. Υπέρ, κατά. Ας επαληθεύσουμε βέβαια. 14. Πέρας ψηφορίας εγκρίνεται. Η 15 υπέρ η φιλελεύθερη. Ας επαληθεύσουμε τη 15. Πέρας Απορρίπτεται. Σας, σας, ψηφί, σας υπολογίσαμε. Ως προσθήκη εγκρίνεται 17 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ. Ας αρχίσουμε την ηλεκτρονική επαλήθευση. 23. Πέρας Εγκρίνεται 21 ψήφι υπέρ, 15 κατά. Συμβιβαστική 3 σε τμήματα όπως έχει στήσει το ΕΛΚΑ. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τέσσερα παρακαλώ. Συμβαστική τέσσερα υπέρ, κατά εγκρίνεται. Η 31 υπέρ. Ας επαληθεύσουμε. 31, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. 32 υπέρ, κατά, εγκρίνεται η 33 με προφορική τροπολογία Μάμφης. Κατά. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Ας επαληθεύσουμε. 34 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 σε τμήματα από την Αλντέ έχει ζητηθεί. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Ε, και αυτό εγκρίνεται. Τριάντα 38. Άρχεται η ψηφοφορία για την 38. Right. The vote is closed. And that's rejected. Πέρας, απορρίπτεται. Και έτσι ψηφίζουμε το σχέδιο γνωματοδότησης, τελική ψηφοφορία, μια ονομαστική. Άρχεται. It's closed. Πέρας. 34 υπέρ και μία κατά. Α, 35 υπέρ, διορθώνω. Λέει ο μιλητής. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και στην Επιτροπή Βιομηχανίας για τον συντάκτη. Μία ψηφοφορία τώρα, μόνο μία, για την ε, έκβαση του τριμερούς διαλόγου για τον Ενωσιακό Τελωνιακό Κώδικα. Θέλετε να πείτε τίποτα, όχι, κύριε Λουγκρίπ. ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Τελωνιακός κώδικας αναδιατύπωση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας, 33 υπέρ. Μία αποχή. Ευχαριστούμε κυρία Ντεγκρυπ, Grip, Και έτσι πάει στην Ολομέλεια το θέμα. Βλέπω και την παρουσία της Επιτροπής εδώ. Κύριο Ζελίνσκι και η ομάδα του αξίζουν συγχαρητηρίων για τη συνεργασία τους μαζί μας και δεν ξέρω αν είναι κανείς και από το Συμβούλιο εδώ, αλλά πάντως και αυτούς πάντα τους ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν έτσι την ψηφοφορία. Μίλης μονεστό, όμως να φέρετε και αύριο στις 12 τις κάρτες σας για την έκθεση Fox και άλλων και άλλες και πάντως σας ενημερώνω ότι η ψηφοφορία για τα σκάφια αναψυχής αναβάλλεται μέχρι να δούμε την έκβαση των σχετικών διαπραγματεύσεων της Παρασκευής. Και πάμε τώρα στην ακρόαση. Όποιος δεν ενδιαφέρεται να μείνει στην αίθουσα παρακαλώ να αποχωρήσει ησύχως. Μέχρι τις 12.30 έχουμε μια πολύ σημαντική ακρόαση. Ησυχία παρακαλώ για τους επισκέπτες μας και καλωσορίζω ιδιαίτερος όλους όσοι ενδεχομένως μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Παρακαλώ αγαπητοί συναδελφοί, ησυχία. So uh, ορίζω όποιον έχει συνδεθεί από το διαδίκτυο για να παρακολουθήσει την ακρόασή μας. Στις επόμενες δύο ώρες ε, καλωσορίζω φυσικά όλους όσοι έχουν επιδείξει την, ε, αυτό το ενδιαφέρον, όσοι θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και μέσω από τον ιστότοπο ε, υπάρχει δυνατότητα της υποβολής σχολείων και βέβαια οι συγητές περιμένουν να τα ακούσουν. Καλώς ήρθατε τους λοιπόν για να προχωρήσουμε. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι όλοι οι συνάδελφοι, οι παριστάμενοι, θα λάβουν αντίγραφο των τοποθετήσεων των ε, βιογραφικών σημειωμάτων των ομιλητών. Είναι πολύ σημαντική η ειδική. κυρία Γκόιενς που βλέπω εδώ και τακτικά έρχεται είναι γνωστή μας. Παλιά γνωστή, αλλά και άλλοι, Βίσνερ Μπουρκε και άλλοι είναι πολλά, πολύ γνωστοί συνάδελφοι. Τους καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι. Είχαμε ξανασυναντηθεί στη συζήτηση για τις προδιαγραφές, αν δεν με τα πρότυπα. Ε, πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναπούμε. Καλωσορίζω την κυρία Μανιου. Α, όχι, δεν είναι εδώ η κυρία Μανιου. Σήμερα. Την ομάδα της Επιτροπής, εν πάση περιπτώσει. Από τις δύο γενικές ευθύνσεις που ασχολούνται εδώ, βλέπω γνωστά πρόσωπα και θα δώσω το λόγο για κάποιες εναρκτήρες παρατηρήσεις στην κυρία Σάλτε Μόζε πρώτα νομίζω και την κυρία Πιέτη μετά και μετά ξεκινάμε την ε, ακρόαση για την ασφάλεια των προϊόντων. Κυρία Σάλτεμος, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω όλους τους ειδικού που είναι εδώ σήμερα Μελέτησα προσεκτικά το τι μπορώ να πω σήμερα, αλλά μια και δεν έχουμε καθόλου περιθώριο χρονικό στην ακρόασή μας, δεν θα υπησέλθω στις λεπτομέρειες των προτάσεων της Επιτροπής. Έχουμε την ευκαιρία αργότερα. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλή ε, ισορροπημένη λύση και πρόταση νομοθετική για, τις, ε, για την ικανοποίηση των αναγκών βέβαια των καταναλωτών και πολιτών, αλλά και για να επιτρέψουμε στη βιομηχανία να λειτουργήσει έτσι, ώστε να έχουμε μια ε, απρόσκοπτα λειτουργούσα ε, εσωτερική αγορά. Έχουμε όμως και εκπροσώπους από την έχουμε όμω προσκαλέσει και εκπροσώπου από τι ΗΠΑ σήμερα, γιατί θέλαμε όχι βέβαια να ευθυγραμμιστούμε, αλλά πάντω να δούμε αν μπορούμε να συντονίσουμε τι νομοθετικέ μα ρυθμίσει. Δεν μπόρεσαν όμω να έρθουν ήθελα να σας ενημερώσω. Πάντως περιμένω να ακούσω τις παρουσιάσεις σας και να συμμετάσχω στις συζητήσει μετά. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, την ώρα που τελειώνατε την ομιλία σας, κατεβάσαμε τα φώτα, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για την εκτίμηση που τρέφουμε στα όσα είπατε. Απλώς προετοιμαζόμαστε για, την, για τις παρουσιάσεις μετά από τις οθόνες. Και θέλω να συγχαρώ την κυρία Σουάλντε Μότσερ για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα για την έκθεση πρωτοβουλία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Όπω ξέρετε, μία από τις πρωτοβουλίε τη Επιτροπή μας είναι η επεξεργασία πολιτικών προτάσεων πριν από την κατάθεση των ε, θέσεων ε, και προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω να πω ότι η κυρία Σουαλντεμόζα στην υπόθεση αυτή έχει κάνει πάρα πολύ προπαρασκευαστικό έργο και τη συγχαίρουμε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρακτική και πιστεύω ότι και άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου μας θα πρέπει να την ακολουθήσουν ώστε να δώσουν ουσία στην διαδικασία τη νομοθετική. Και περιμένουμε να δούμε να αντικατοπτρίζονται αυτέ τι προτάσει και στι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Πιέτικα είναι τώρα για την ε, ποιοπτία τη αγορά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και εγώ. Ε, για λόγους χρόνου θα είμαι σύντομη. Ξεκινώ ζητώντα συγγνώμη που θα χρειαστεί να αποχωρήσω γιατί είμαι σκιώδη συγγήτρια σε τριμερή διάλογο και διαπραγματεύσει για τι καταχρήσει αγορές. Ε, πάντως ε, θα επανέλθω για το τελευταίο τμήμα της συζητήσεως όπου θα μιλήσουμε κυρίως για την εποπτεία στην ε, ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχολεί και για τον καταναλωτή βεβαίως, για την πτυχή της ασφάλειας, αλλά και για λόγους ευθύνης στην αστική ευθύνη στην εσωτερική αγορά και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλε αυτέ τι διατάξει χωρί ε, περιττή γραφειοκρατική επιβάρυνση. Ωστόσο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό και για την ε, Ευρώπη 2020. Η καινοτομία, η ε, παραγωγή, τα νέα και ασφαλή προϊόντα στην Ευρώπη πώς μπορούμε να τα αναπτύξουμε, πώς μπορούμε να έχουμε νομοθεσία για την ε, ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και πώς μπορούμε να μεριμνήσουμε ώστε να έχουμε την εποπτεία της στήρησης των ρυθμίσεων αυτών, των διατάξεων αυτών. και μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να βρουν πιο ευνοϊκή ε, αντιμετώπιση ε, εκείνοι οι οποίοι ε, με μεγαλύτερη χαλαρότητα αντιμετωπίζουν τους κανόνες σε σχέση με αυτούς οι οποίοι προσαρμόζουν την παραγωγή τους σε αυτούς. Ήταν πολύ καλή ιδέα της κυρίας Σαλτεμόζε να έχουμε εκπροσώπου για να αντιληφθούμε ποιε είναι οι διατάξει και πώ εφαρμόζονται οι διατάξει από την Αμερικανική πλευρά και να προχωρήσουμε στη συνέχεια και σε συντονισμένο ενδεχομένω. Τα σχόλια μου ήταν αυτά λοιπόν και περιμένω να ακούσω τι προτάσει μέσα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ασφαλώ δημόσια ακρόαση και που θα αποτελέσουν μια πολύ καλή βάση για τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τι δύο για τη δουλειά που κάνουν στο θέμα αυτό. Θα ξεκινήσουμε ε, το πρώτο τμήμα της ακρόασης ε, μέχρι τις 11.30. Θα ασχοληθούμε με τις πτυχές ε, της ασφάλειας των προϊόντων, το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας προϊόντων και της εξορρόπησης των αναγκών των ενδιαφερομένων, δηλαδή που συμμετέχουν στην, στο σχεδιασμό, παρασκευή, εμπορευματοποίηση και πώληση αυτών των προϊόντων στους καταναλωτές. Θα δώσω ένα πεντάλεπτο στο κάθε καλεσμένο μας και μάλιστα θα ενεργοποιήσουμε το χρονόμετρο για να μην αφαιρεθείτε. Και μάλιστα δεν ήρθε δυστυχώς ο εμπειρογνώμονας ακόμη από την Αμερικανική Πρεσβεία που κάλεσε η κυρία Σαλντεμόζε. Βλέπω ότι ε, τα φώτα ξαναδυνάμωσαν. Φαντάζομαι θα χαμηλώσουν σε λίγο. Έχουμε τη Μόνικο Γιένς, που είναι Γενική Διευθύντρια της BOIC, του Ευρωπαϊκού Κινήματος Καταναλωτών. Είναι γνωστή στην Επιτροπή μας. Ε, είναι πάντα ευπρόσδεκτη στην Επιτροπή. Έχουμε τον Ζαν Φιλιμποφόρ, που είναι εμπειρογνώμονα σε θέματα ευθύνη για τα προϊόντα και ασφάλεια προϊόντων, σύμβουλο πολλών ε, επιχειρήσεων και ειδικό σε θέματα ασφάλεια προϊόντων. Η Εμιλή Προυσέ, ε, πρωτοστατεί στο θέμα αυτό εκ μέρους της Eurocommerce, ε, Ένωσης ε, Ελληνεμπόρων και φυσικά ε, έχει άμεσες επαφές με τους πελάτες και επίσης έχουμε και έναν πρόεδρο της Ένωσης Επιπλοποιών που θα μας δώσει τη δική του εμπειρία από την εφαρμογή των διατάξεων. Πόρατα το λόγο έχει η κυρία Γκόγενς για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε θερμά και για την πρόσκληση. Φυσικά το θέμα της ασφάλειας, των της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών είναι ένα τεράστιο ζήτημα της πολιτικής των καταναλωτών και ύψιστη προτεραιότητα για μας. Έχω μόνο ένα πεντάλεπτο από ό,τι κατάλαβα. Είναι αδύνατο βέβαια να είμαστε εξαντλητικοί σε ένα τόσο περίπλοκο πακέτο. Αλλά σας έχουμε στείλει και ένα ενδελεχές έγγραφο ε, με τις θέσεις μας που καταρτήσαμε από κοινού με την ΑΝΕΚ ε, την Αδελφού Ένωση. Οπότε έχετε εκεί πολύ πιο λεπτομεριακά σχόλια. Εδώ θα επικεντρωθώ σε 4-5 μείζωνα ζητήματα. Καταρχήν, ω προ το πακέτο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί διαπιστώνουμε κάποιε ευπρόσδεκτε βελτιώσει, αλλά έχουμε και κάποιε επιφυλάξει και ανησυχίε. Η πρώτη μα ε, ανησυχία είναι ότι η τρέχουσα νομοθεσία ε, είναι νομοθεσία ονόσημο, ορόσημο, γιατί θεωρείται ω δίκτυο ασφαλεία. Και ε, το GPSD, αυτός ο κανονισμός για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, ε, αναλαμβάνει κάποια δράση για την προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια των καταναλωτών. Βέβαια, διαπιστώσαμε στην τελευταία πρόταση μια αλλαγή του ύφου. Και δεν υπάρχει πια η εντύπωση αυτή, ότι αυτή η οριζόντια νομοθεσία συνιστά και ένα δίκτυο ασφαλείας και η τήρηση των τομεακών κανόνων θεωρείται πια αεπαρκής για την θέση εμπορία ενός προϊόντος, κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Σε μερικά σημεία πιστεύουμε ότι δεν επαρκεί η τομεακή νομοθεσία για να καλύψει όλα τα θέματα ασφάλεια του προϊόντο. Δεύτερη επιφύλαξη. Έχει εξαφανιστεί η αρχή τη προφύλαξη, κάτι που κρούει για μα τον κόδωνα του κινδύνου αν θεωρηθεί αυτονόητο, προτιμούμε παρόλα αυτά να αναφέρεται ρητά στο κείμενο, γιατί το θέμα της αρχής προφύλαξης ή της πρόληψης ε, είναι σημαντική για τις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υπόνοια ή μερική απόδειξη για την ε, ύπαρξη κινδύνου, καλό θα είναι να αναλαμβάνετε δράση για να εξασφαλιστεί η προστασία και ασφάλεια των καταναλωτών. Πάντως, ε, αυτό που καλωσορίζουμε στο κείμενο είναι ότι ο κανονισμό προβλέπει πιο αποτελεσματικά εφαρμοστικά μέτρα που θα είναι και δεσμευτικά και μόνιμα. Ενώ στο ισχύον σύστημα ε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό τη νέα πρόταση που ευελπιστούμε ε, θα παραμείνει αλόβητο καθ' όλη τη διάρκεια τη νομοθετική διαδικασία. Χαιρετίζουμε και τι διατάξει του κανονισμού που αφορούν τη βελτίωση τη συχνηλασιμότητας των προϊόντων. Ιδιαίτερα το γεγονό ότι το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστού ή του εισαγωγέ θα πρέπει να αναφέρεται, να, να φαίνεται στο προϊόν. Βέβαια το θέμα του, της, ε, της, ε, της, ε, της αναφοράς προέλευσης μάλλον ε, δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές παρά εξασφαλίζει κάποια σαφήνεια. Φυσικά θα πρέπει να αποφεύγονται παραπλανητικές πληροφορίες για τους καταναλωτές και το σήμα Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αφαιρείται από το πακέτο ή την, το προϊόν γιατί παραπλανεί τους καταναλωτές και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις για την ασφάλεια του προϊόντος και δεν εξασφαλίζει την ε, σωστή πληροφορία για την ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να θεωρείται ως τεχνικό έγγραφο για τις αρχές εποπτείας, αλλά όχι ως εργαλείο για τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή αυτό το ευρωπαϊκό σήμα. Και τέλος, σημαντικό όμως θέμα, για να τηρήσω το πεντάλεπτο, όπως ανέφερε και η κυρία Σχαλντεμόζερ, είναι σημαντικό να μην περιοριζόμαστε στα όρια, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λάβουμε υπόψη και την παγκόσμια αγορά, τη διεθνή αγορά και από αυτήν την άποψη μας προβληματίζουν οι σχέσεις ελεύθερων συναλλαγών και διαπραγματεύσεις για την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί φοβόμαστε ότι κάποιοι κανόνες ασφάλειας τροφίμων θα τεθούν σε κίνδυνο εξαιτίας των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ακριβώς επειδή δεν έχουμε πρόσβαση ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών στη διαπραγματευτική εντολή στο κείμενο, ε, στηριζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσει και να μεριμνήσει ώστε το θέμα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων και του καταναλωτή να μην αφαιρεθεί από τις εμπορικέ διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ασφαλώς θα διατυπωθούν ερωτήσεις μετά. Θα υπενθυμίσω μόνο στους συναδέλφους ότι θα έχουμε χρόνο αργότερα για την υποβολή ερωτήσεων προς τους ε, ομιλητές μας, για τις παρατηρήσεις τους. Και τώρα, ο κύριος Μονφόρ, με διαφάνειες. Θα ξανακατεβάσουμε λοιπόν τα φώτα. Έχετε πέντε λεπτά κύριε Μονφόρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η δική μου προσέγγιση είναι το πώς μπορεί να αξιολογήσει την διάθεση στην αγορά προϊόντων ασφαλών ένας νομικός. Και θα προσπαθήσω να δώσω τη συμβουλή που θα έδινα ως δικηγόρος ε, στον παραγωγό, στον κατασκευαστή. Όπως ξέρετε αντιμετωπίζουν πολύ περίπλοκες νομοθεσίες και πολλά περίπλοκα νομοθετήματα οι ε, κατασκευαστές, η παραγωγή. Πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιους όρους μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια των ε, προϊόντων. Για το καλό βέβαια του καταναλωτή και της ιστορικής αγοράς. Χρειάζεται μια σαφής και αναλογική υποχρέωση για ενημέρωση. Καταρχάς, τη ευκρίνηση του νομικού πλαισίου. Το πλαίσιο που έχουμε με την Γενική Οδηγία, τη GPSD, και τις άλλες διατάξεις που ισχύουν παραδείγματι στο πακέτο για, τις, ε, για τα αγαθά, ε, για τα προϊόντα όπως ε, τα νομοθετήματα 768 και 765 ε, αποτελούν μια περίπλοκη, ένα περίπλοκο πλαίσιο, ακόμα και για νομικούς όπως εγώ. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο λοιπόν να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η σαφήνεια του κανονισμού και ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της προτινόμενης ε, εναρμόνισης και της εναρμονισμένης ε, αγοράς. Εάν δείτε, Υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν αποκλειστεί από την CPSR όπως ε, τρόφιμα, υπάρχουν άλλα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί και ως εκ τούτου καλύπτονται πλήρως από την CPSR και κάποια άλλα που ανήκουν σε τομείς ρυθμιζόμενους και δεν έχουν εξαιρεθεί και ως εκ τούτου υπάρχονται στην CPSR και τελικά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι ισχύει. Το άρθρο 2.4 με τις ε, παρεκκλήσεις στα κεφάλαια 2 και 4 δεν είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ε, διατάξεις επαρκής για την ε, προστασία της υγείας και ασφάλειας με εναρμονισμένες ε, διατάξεις. Δηλαδή εξαιρούνται τα καλλιτικά και τα παιχνίδια ουσιαστικά τα οποία, για τα οποία έχουν υιοθετηθεί με βάση τη διάταξη 768 ειδικέ διατάξεις ή 768 καλύτερα ειδικέ διατάξεις. Υπάρχουν άλλες ρήτρε, υπάρχουν τομείς διαφορετικοί οι οποίοι ενδεχομένως υπάγονται στις προϋποθέσεις για την υγεία και την ασφάλεια. Ε, είναι σαφή η κατάσταση λοιπόν και εγώ θα πρότεινα είτε να εφαρμοστεί το CPSR ως μοναδικό νομοθέτημα το οποίο θα προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, του, δρα... του ε, φορέα παραγωγής ε, και μόνο, είτε τότε θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε με εναρμονισμένη νομοθεσία σε ρυθμιζόμενου τομεί. καλλιτικά δηλαδή, θα μπορεί κανεί να κοιτάξει ποιο είναι ο κανονισμό για τα καλλιτικά που εφαρμόζεται και θα εφαρμόζεται μόνο αυτός ο κανονισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πιστεύω θα πρέπει να σα απασχολήσει ε, και προσωπικώ θεωρώ ότι το CPSR θα πρέπει να παραμείνει ω μόνο νομοθέτημα που θα ισχύει για όλους τους τομείς και, την, και θα έβγαζα την οδηγία για τα παιχνίδια και τα καλλιτικά με τις διατάξει που έχουν εισαχθεί τώρα στο CPSR και οι στο CPSR. Η αναλογικότητα τώρα των ε, προϋποθέσεων και θα επικεντρωθώ σε ορισμένες μόνο από αυτές. Καταρχάς μια προσέγγιση στηριζημένη στην διακινδύνευση. Ε, είναι πολύ σημαντικό εδώ να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ της στήρησης των προδιαγραφών και της ασφάλειας. Το GBST ήταν, ε, αφορούσε την ασφάλεια, ενώ το νέο CPSR εισάγει ορολογία που προέρχεται από το πακέτο για, τις, ε, για τα προϊόντα που έχει να κάνει με συμμόρφωση, compliance. Και εδώ ακριβώς έχουμε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών ζητημάτων και δύσκολες αποφάσεις για τον παραγωγό, τον κατασκευαστή και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η GPSD η οδηγία αφορά περισσότερο την ασφάλεια και όχι την συμμόρφωση δύο διαφορετικές, δηλαδή αντιλήψεις νομικές. Επίσης προς την ισότιμη κατανομή των ευθυνών. Θα έλεγα ότι οι διατάξεις όπως έχουν καθιστούν πολύ δύσκολο ιδιαίτερα το ρόλο των, ε, του διανομέα στο να εξασφαλίσει την επαλήθευση της ασφάλειας. Δηλαδή θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον παραγωγό, τον Ευρωπαίο παραγωγό, εισαγωγέα κτλ να βεβαιωθεί ότι είναι ασφαλή τα προϊόντα, να ε, παληθευτεί αν έχει την υποχρέωση να το πράξει αυτό και το καθεξής. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη εισήγηση και ενδεχομένως να απαλλάσσεται ο κατασκευαστής από την ευθύνη σε περίπτωση που έχει πια περάσει όλη τη διαδικασία και έχει έχουν ενημερωθεί οι κρατικές αρχές στο να προσαρμόσει ένα προϊόν στις ε, προδιαγραφές. Μάλλον έχει εξαντληθεί ο χρόνος μου, αλλά πάρα πολύ στο με ένα τελευταίο σχόλιο, προσωπικού χαρακτήρα μάλλον. Εγώ θα πρότεινα οι εμπλεκόμενοι στην αγορά να κοινοποιούν όχι απαραίτητα σε εθνικό επίπεδο τα μη ασφαλή προϊόντα, αλλά ίσως θα πρέπει να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλη εμπειρία, γνώση, πείρα και όταν έχουμε να κάνουμε με παγκόσμιο χαρακτήρα δυνατότητες ε, προσφυγής, Κινέζους, Αμερικανούς, Βραζιλιάνους, Ευρωπαίους, καλό θα είναι να μην μπορεί κανείς να, ή να μην χρειάζεται κανείς να επιλέξει το σωστό κράτος μέλος και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα εφόσον ε, υπάρχει ζήτημα να ενημερωθεί από τις επιχειρήσεις για προϊόντα των οποίων η ασφάλεια ίσως αμφισβητείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ που μας είπατε όλα αυτά τα σημεία. Υπάρχει ένα θέμα για την αρχή της ε, προφύλαξης ε, που το ανέφερε η προηγούμενη ομιλήτρια. Ε, υπάρχουν αντίγραφα των διαφανειών για τους συναδέλφους, θέλω να το πω αυτό. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην κυρία Πχουζέ από το Eurocommerce. Θα μιλήσει από τη δική της κοπιά για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε τους ίδιους ε, σκοπούς, ότι πρέπει να διαθέτουμε δηλαδή στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να πλουστεύσουμε τα συστήματα, την ε, πραγματογνωμοσία, την κάλυψη των προϊόντων και κυρίως ε, την ευθύνη που έχει ο κάθε δημόσιος και ιδιωτικός φορέας με σαφή και ισορροπημένο τρόπο. Θα ήθελα καταρχήν λοιπόν να τονίσω κάποια στοιχεία. Μιλάμε ε, για χιλιάδες προϊόντα που έχει ένα κατάστημα, το οποίο προέρχεται από πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές, από μεγάλες εταιρείες, μικρές εταιρείες. Επίσης, καμιά φορά έχουμε και τα δικά μας προϊόντα στο μαγαζί, δηλαδή τα, που τα έχουν κάνουν ε, λιανέμποροι, για ειδικέ εξειδικευμένες ανάγκες των καταναλωτών. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι κατασκευαστέ έχουν την ευθύνη για τα δικά του προϊόντα, οι διανομείς έχουν την ευθύνη για προϊόντα από τους εισαγωγείς, οι Ευρωπαίου κατασκευαστές και μερικέ φορές ε, έχουμε και την ε, ευθύνη ω εισαγωγή. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο ευθυνών ανάλογα με την νομοθετική κάλυψη των προϊόντων. Τρόφιμα, μη τρόφιμα, εναρμονισμένα, μη εναρμονισμένα θα επικεντρωθούμε λοιπόν στις υποχρεώσεις των διανομέων σήμερα. Ε, θα δείτε τις διαφάνειες και τις κοινέ ε, προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε για προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα. Αυτή τη στιγμή σιωθετηθεί το πακέτο. Τι σημαίνει όμως αυτό συγκεκριμένα. Έχουμε ήδη την εμπειρία αυτών των κανόνων για τη νέα οδηγία για τα παιχνίδια, η οποία θα τεθεί σε ισχύ και επίσης έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Να σα εξηγήσω τι εννοώ. Αν πάρετε ένα παιχνίδι το οποίο οι διανομή θα πρέπει να ελέγχουν ότι το προϊόν έχει κάποια σήματα, ε, το ΕΚ, το όνομα του παραγωγού, την διεύθυνσή του. Επίση, ε, και για τα μη αρμονισμένα προϊόντα ίδιες υποχρεώσει υπάρχουν. Αυτή η υποχρέωση όμω ε, ερμηνεύεται τελείως διαφορετικά στην Ευρώπη και από τις αρχές επιτήρησης αγοράς. Θα θέλαμε να πρέπει να ελέγχονται η, καταρχάς και τα σήματα και η αληθοφάνεια αυτών. Δεν θα πρέπει να επαληθεύεται η, τα όσα λέει η, το σήμα. Επίσης χρειαζόμαστε τεχνικές πληροφορίες, αλλά Συχνά αυτή η τεκμηρίωση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα όταν ζητάμε από τους ε, εμπορικούς μας εταίρους. Υπάρχουν θέματα εδώ επιτεπτικότητας, αντιγραφής κτλ. Φαντάζεστε η Apple ας πούμε, να δώσει ε, στο καφού όλες τις τεχνικές ε, πληροφορίες και προδιαγραφές των προϊόντων. Αποκλείεται. Αν κάνουμε μια ανάλυση και να δούμε την επάρκεια των σημάτων, αυτό το κόστος κάποιος πρέπει να το φέρει, κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Πώς θα γίνει αποτελεσματική αλυσίδα προσφοράς προϊόντων. Στην ευρωπαϊκή αγορά οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν τη βασική ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων. Γιατί είναι αυτοί που έχουν όλη την πραγματογνωμοσύνη, όλη τη γνώση για το προϊόν. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβε την ανάγκη για ισορροπημένους ορισμούς ε, δεν θα πρέπει να έχουμε τεχνικές, ε, τεχνική τεκμηρίωση για όλα τα προϊόντα, αλλά θα πρέπει να έχουμε στοιχεία για την ε, γρήγορη ανείχνευση του προϊόντος. Οι διανομής είναι στοιχεία κλειδιά που ελέγχουν την παρουσία του προϊόντος ε, και μειώνουν και τον κίνδυνο ε, διαφορετικής ερμηνείας. Επίσης, θα πρέπει να έχουν τα τεχνικά στοιχεία ε, και να είναι θεματοφύλακες όλων των, της τεκμηρίωσης που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας αγοράς. Υποστηρίζουμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ θα πρέπει να εμπλακούν και οι επιχειρήσεις να δώσουν την πραγματογνωμοσύνη τους, να εξηγήσουν τις ανησυχίες τους. Αυτή τη στιγμή ένα προϊόν μας λένε ε, διανεμηθεί κάπου, γιατί θα πρέπει να ελεγχθεί, ας πούμε στην Ισπανία, γιατί θα πρέπει να ελεγχθεί και στις υπόλοιπε χώρες. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην, στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Θα πρέπει η πληροφορία να είναι ε, ψηφιακή, να, δίδεται και στα αγγλικά. Επίσης, δεν θα πρέπει οι πληροφορίες στα τελωνία να είναι οι μόνες πληροφορίε για την ανιχνεσιμότητα. Θα πρέπει να προωθήσουμε την αναλογικότητα, μεγαλύτερη συνέπεια και να απλουστεύσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την καλύτερη εφαρμογή μέσω του μηχανισμού ασφάλειας. Uh, και τέλο για τον πρώτο γύρο, ο κύριο Μάρκο Βίσνερ, που είναι πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Επίπλων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση στην δημόσια αυτή ακρόαση. Και ο πρόεδρος ΕΦΕΚΤ τη Ευρωπαϊκής ε, Βιομηχανίας Επίπλων απασχολεί 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους και αντιπροσωπεύει 150.000 επιχειρήσει, Βέβαια, εγώ εκπροσωπώ τον αυστριακό κλάδο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Είναι καθημερινή μα μέρημνα και είμαστε υπεύθυνοι για κάθε λάθο που λαμβάνει η χώρα και είμαστε υπεύθυνοι να αναλάβουμε τα μέτρα για να αποφύγουμε τραυματισμούς εξαιτία αδυναμιών στην ασφάλεια. Οπότε μα επηρεάζει άμεσα η πρόταση αυτή και θέλουμε αυστηρά να τηρήσουμε τις διατάξεις της. Να είμαι σαφή λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Επιπλών ε, χαιρετίζει θερμά την πρόταση, γιατί είναι μια καινοτόμα πρόταση για την προστασία του καταναλωτή και επιπλέον είναι ένα πρακτικό εργαλείο για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να τονίσω ότι χαιρετίζουμε ιδιαίτερα στο θέμα της ταυτοποίησης και της ε, αναφοράς της προέλευσης. Και να σας εξηγήσω γιατί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στους καταναλωτές. Οι καιροί έχουν αλλάξει και η συμπεριφορά των καταναλωτών επίσης έχει αλλάξει. Οι καταναλωτές ε, δεψούν για περισσότερες πληροφορίες και ο κλάδος, η βιομηχανία θέλει να δίνει τέτοιες πληροφορίες. Η παραγωγή θα πρέπει να είναι πιο διαφανής ε, σε ό,τι αφορά τον τόπο παραγωγής και οι καταναλωτές ε, έχουν δικαίωμα να κάνουν ε, κατατοπισμένη και τεκμηριωμένη την επιλογή τους. Θα πρέπει να γνωρίζουν και τον παραγωγό και τον εισαγωγέα. Δεν θα πρέπει να αποκρύβονται πληροφορίες από τον καταναλωτή και η αναφορά της προέλευσης χορηγεί επιπλέον γνώση στον καταναλωτή. Ο καταναλωτή θα πρέπει να γνωρίσει και την προέλευση δηλαδή του προϊόντος, τον, τον τόπο παραγωγή και να ενημερώνεται καλύτερα για, τα, για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές στον τόπο προέλευσης. Θα πρέπει έτσι να μπορεί ελεύθερα και τεκμηριωμένα να κάνει τις επιλογές του. ό,τι αφορά τη βιομηχανία ειδών επίπλωσης. Εμείς έχουμε τα παράπονα όλο και περισσότερων παραγωγών κατασκευαστών επίπλων ότι εξαναγκάζονται να αφαιρέσουν τις ετικέτες τους ε, με πληροφορίες για τα έπιπλα. Και αυτό για να αποφευθεί οποιαδήποτε ε, ταυτοποίηση για τον καταναλωτή. Κατά τη γνώμη μας, περισσότερη ενημέρωση σημαίνει και περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων. Γιατί ο εντοπισμός της χώρας προέλευσης ε, διευκολύνει το έργο των, ε, των ε, αρχών ελέγχου για την ειχνηλασιμότητα ενός προϊόντος, εφόσον η ταυτοποίηση, η εντοπισμός είναι δύσκολος μερικές φορές. Βέβαια έτσι αυξάνεται και η ευθύνη του παραγωγού, του κατασκευαστή. Γιατί ο καταναλωτής θα ζητήσει να λογοδοτήσουν οι οικονομικοί τελεστές για τη συμμόρφωσή τους ε, με την ασφάλεια των προϊόντων. Και μάλιστα σε εμά στην βιομηχανία επιπλέον ο παραγωγό είναι υπεύθυνο για όλα τα μέτρα που αφορούν την ασφάλεια του προϊόντο. Ε, Δοκιμέ, ε, πιστοποίηση, αποσύρσει προϊόντων και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν ε, η βιομηχανία επίπλων να είναι σίγουρη ότι όλοι οι παραγωγοί φέρουν την ίδια ευθύνη. Δεν ζητούμε λοιπόν αύξηση του προστατευτισμού σε καμία περίπτωση. Εμείς απλώς θέλουμε ίσες ε, και θεμητές συνθήκες ανταγωνισμού. Κάθε παραγωγός και κατασκευαστής θα πρέπει να φέρει το ίδιο μερίδιο της ευθύνης. Ε, κερδισμένος ε, από την ε, ίση αυτή ευθύνη, τη δίκαιη κατανομή της ευθύνης, θα είναι ο καταναλωτής. Επίσης, μας ενδιαφέρει η χνηλασιμότητα των προϊόντων και πιστεύουμε ότι η αναφορά της προέλευσης θα ωφελήσει και τον καταναλωτή και την ευρωπαϊκή μεμηχανία. Ε, ζητούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της μια ισχυρή βιομηχανική βάση που είναι απαραίτητη για μια ευημερούσα και αθώς οικονομικά Ευρώπη. Και φυσικά θέλουμε μέτρα που θα προωθήσουν και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανία μας. Η βιομηχανία επίπλο λοιπόν θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η υιοθέτηση μιας καλής άρτιας πρότασης που φυσικά επιδέχεται βελτιώσει, αλλά κατά τη γνώμη μα είναι θετική αυτή τη στιγμή και με τη μορφή που έχει και για του παραγωγού και για του καταναλωτέ. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ όλου. για τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που μα εκθέσατε. Τώρα να ακούσουμε τα σχόλια και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Τώρα στους ομιλητές. Θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και μετά θα έχετε το περιθώριο να απαντήσετε. Η κυρία Σχάλντε Μόζε πρώτα. Ο κύριος Μπαλτασάρη θέλει επίσης να μιλήσει. Έχει αναλάβει το έργο του Σκιώδου Συγητή εκ μέρους του, κυρίου, ε, εκ του Ο κύριος Φόξ όμως είναι εδώ και άλλοι. Η κυρία Σφάλτε μαζί πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες σας και την παρουσίασή τους τόσο σύντομα. Ε, θα ήθελα πολύ βέβαια να τις συζητήσουμε και έχω μια ερώτηση προς όλους. Μονίκ, είπες εσύ ότι είναι πολύ σημαντική η αρχή της πρόληψης στην νομοθεσία και ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να έχουμε την αρχή της πρόληψης και έναν ορισμό του σοβαρού κινδύνου, της σοβαρής διακινδύνευσης. Αυτό θα μας θα σε κάλυπτε για τον κύριο Μόντφορτ. Μονφό. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε και τη συμμόρφωση και την ασφάλεια ταυτόχρονα μέσα στην νομοθεσία σαν προσέγγιση. Θέλετε να μας κάνετε μια πιο διεξοδική παρουσίαση των θεσεών σας για την ε, e-commerce. Δεν είμαι βέβαια αν κατάλαβα τι εννοείτε. Μιλάτε για χαλάρωση των υποχρεώσεων από τη νέα νομοθεσία ως προς το ρόλο του διανομέα. Διότι αν συμβαίνει αυτό δεν θα συμφωνήσω. Εάν όμως υπάρχει θέμα διευκρίνησης των ε, υποχρεώσεων του, του κατασκευαστή, τότε να το συζητήσουμε. Πάντω για μα ήταν σαφέ όταν ήρθε η ώρα με το NLF ε, στο η προηγούμενη θητεία, μάλιστα είχα ασχοληθεί εγώ και με την απόφαση 768. Είχαμε πει ξεκάθαρα ότι πρέπει να επιβληθούν σε όλου του παράγοντε που εμπλέκονται στην αγορά οι υποχρεώσει. Αν μπορούμε να βρούμε δηλαδή τον κατασκευαστή τόσο το καλύτερο, εάν όχι, ο διανομέα έχει φέρει εκείνο την ευθύνη αφού εκείνος φέρνει το προϊόν στην αγορά. Ας το αναπτύξετε όμως λίγο. Και μια τελευταία για τα έπιπλα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είπατε όντως ότι δεν έχετε καμία πρόταση για αλλαγή, για τροποποίηση. Και για την Business Europe συμφωνεί και η Business Europe σε αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ κύριε Μπαλτασάρε. Εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμώ τις παρεμβάσεις των εμπειρογνωμόνων. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Η Κομισιόν παρουσίασε ένα πακέτο που ανταποκρίνεται στο αίτημα να έχουμε ένα πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για όλα τα προϊόντα. Και μιλάμε εδώ για τα καταναλωτικά προϊόντα και για τα μη καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή η διάκριση δεν είναι σαφής. Δεν μας διευκολύνει. Και μια και την ξαναβρίσκουμε αυτή τη διάκριση στο νέο πακέτο, ανάμεσα σε καταναλωτικά και μη καταναλωτικά προϊόντα. Διερωτώ λοιπόν, μπορούμε πραγματικά να, να κάνουμε αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε καταναλωτικά και μη καταναλωτικά προϊόντα. Πώς θα διακρίνετε τα προϊόντα για να καταλάβουμε λιγάκι ε, πιο καλά αυτή τη διάκριση. Επιπλέον. Σε αυτή την οδηγία αναφέρονται μία σειρά από προϊόντα εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν αποκλείονται και μία σειρά από προϊόντα που δεν εμπίπτουν εκεί. Δεν θα είχε νόημα ε, να έχουμε ένα κατανονισμό για όλα τα προϊόντα εκτός από αυτά που συμπεριλαμβάνονται σε άλλες πράξεις εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη διχοτομία πώς την αντιλαμβάνονται οι εμπειρογνώμονες αυτή η διχοτομία που υπάρχει στην, στην πρόταση που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή. Οι εμπειρογνώμονες πώς την αντιλαμβάνονται, τι άποψη έχουν. Ευχαριστώ. Άκουσα και τον κύριο Μπαλτασάρ και την κυρία Σόλτε Μόζε και συμφωνώ και με τις δύο. Θα ήθελα να θέσω μάλιστα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτές. Ε, ε εξεπλάγει και με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση ε, των ε, λεγόμενων καταναλωτικών προϊόντων. Τι άποψη έχουν οι εμπειρογνώμονες. Πιστεύω ότι είναι καλό αυτό που πρότεινε η Επιτροπή ή θα δημιουργήσουν, θα δημιουργήσουν αυτές οι αλλαγές α, περαιτέρω προβλήματα. Ο, το γεγονός δηλαδή ότι περιορίζεται ο ορισμός ας πούμε των κανονικών προϊόντων. Επίσης οι εξαιρέσεις δεν είναι σαφείς, δεν ρυθμίζονται με σαφήνεια. Υπάρχει υπερβολική έτσι νεφελώδης κατάσταση και πολλοί περιορισμοί. Ποιε είναι οι απόψει των εμπειρογνωμόνων. Επίση υπάρχει η προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο. Επηρεάζει όλο το πακέτο. Αυτή η προσέγγιση όμω δεν έχει προσδιοριστεί πουθενά. Ο κίνδυνο δεν έχει προσδιοριστεί πουθενά και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Σαλντεμόζ εδώ. Το πρόβλημα της ασφάλειας τότε και της προσέγγισης που να βασίζεται στον κίνδυνο, αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα δούμε από κοινού. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο σαφή ορισμό αυτής της έννοιας, της προσέγγισης που να βασίζεται στο ρίσκο, στον κίνδυνο. Επίσης, συμφωνώ με την κυρία Σαλντεμόζε ότι τελικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν εδώ. Οι παραγωγοί φυσικά έχουν ευθύνη, αλλά φυσικά και οι εισαγωγεί έχουν ευθύνη και οι μεμονωμένοι ναι λιανέμποροι. Ο καθένα έχει την ευθύνη του. Κανένα άλλο τρόπο δεν υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Όλοι πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του. Ο κύριο Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει, αν μου επιτρέπετε. Καταρχά, για την ένδειξη τη προέλευση στο άρθρο 7. Οι εμπειρογνώμονέ μα μπορούν να μα σχολιάσουν την πιθανή επίπτωση στι επιπτώσει αυτού του άρθρου από την μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν ε, ξέρω ότι δεν έχει αποτιμηθεί το κόστος στις επιχειρήσεις και στις κυβερνήσεις. Φυσικά αυτό το κόστος κάποιος θα το πληρώσει. Πολύ πιθανώς ο καταναλωτής, φαντάζομαι. Ποιες είναι οι απόψεις για αυτό το σημείο. Δεύτερον, στο άρθρο 15 και το σύστημα ανιχνευσιμότητας. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα, αντιμετωπιστούν, καθοριστούν οι ομάδες προϊόντων ή τα προϊόντα μέσω καταξιοδότηση πράξεων. Σας αρέσει αυτό. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εμείς περνάμε την ε, νομοθεσία και η Κομισιόν κάνει ό,τι θέλει, ό,τι της καπνίσει. σε ποιο βαθμό χρειαζόμαστε δημόσια διαβούλευση και μελέτη αντικτύπου για αυτές τις ε, πράξη. πράξεις. Γιατί η Κομισιόν έχει την τάση, αυτή τη στιγμή συζητούμε κάποιες εξουσίες, ε, να κάνει μετά το δικό της. Ποια είναι τα σχόλιά σας αυτό. Ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι και εγώ πότε θα μιλήσουμε για τις εφαρμοστικές πράξεις. Κύριε Σαλβίνη. Grazie Presidente, vorrei capire una volta Το σήμα προέλευσης έχει ένα κόστος. Το κόστος αυτό είναι ε, αποδεκτό ότι, ή είναι υπερβολικό. Δεν θέλω να μπλέξουμε τον, τον καταναλωτή. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε ποιου θα υποστηρίξουμε εδώ, του πολίτε ή τι επιχειρήσει. Κυρίω αυτέ που παράγουν χωρί να σεβαστούν κανένα πρότυπο ασφάλεια, ε, ε, προστασία του περιβάλλοντο, προστασία των ε, εργαζομένων. Αλλιώ κοροϊδευόμαστε. Αυτό που ονομάζεται επίση ελεύθερη αγορά στην Ινδία, στην Ιαπωνία, στι Ηνωμένε Πολιτείε συνδέεται με την προστασία τη τοπική παραγωγή. Εδώ τα, τα αισθάνομαι αμήχανα, αμήχανοι. Ορισμένοι διερωτώνται γιατί αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός. Αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ευρώπη δεν μπόρεσε να προσφέρει στους καταναλωτές τη τη σιγουριά ότι αγοράζουν αυτό. Ότι αυτό που αγοράζεις παρασκευάζεται εκεί. Εάν δεν μπορεί να δώσει αυτή τη σιγουριά στου καταναλωτέ, η Ευρώπη δεν ε, χρησιμεύει σε τίποτα. Ε, προστατεύουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, ε, τους ε, Ευρωπαίους εργαζόμενους ή εκείνους που μετεγκαθίστανται στο Μπαγκλαντές, στο Πακιστάν και πληρώνουν τον κόσμο 3 ευρώ τη μέρα. Και μετά λένε «Α, δεν θα πρέπει να μπερδεύουν οι ετικέτες». Γιατί αν εμείς προχωρήσουμε με αυτό το ρυθμό, τότε οι υποστηριχτές ενός άλλου τύπου Ευρώπης θα πολλαπλασιαστούν. Πρέπει η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι πολίτες να ξέρουν τι αγοράζουν, τι τρώνε, τι παπούτσια αγοράζουν, τι κλωστοφαντουργικά αγοράζουν, τι αγρο... αγροτικά προϊόντα και τι τρόφιμα αγοράζουν. Αν δεν τα ξέρουμε αυτά, η Ευρώπη αυτή δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Ακούσαμε όλους τους κοιόδες εισηγητές Έχω την κυρία Κοφεράτη και την κυρία Ρόιτεμπεργκ. Εκτό από αυτού θέλουν και άλλοι να πάρουν τον λόγο. Ο κύριο Κοφεράτη. Πώς... Συνεχεία κυρία Ρόιτεμπεργκ. επειδή δεν μίλησα για την, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, νομίζω ότι η κυρία από την Κομισιόν μπορεί να μιλήσει. Ε, ναι, εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Και υπάρχει και εκπρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Δεν ξέρω αν θα, έχετε, θα έχουμε το χρόνο να σας ακούσουμε και το απόγευμα, αλλά σίγουρα θα καθίσετε κι άλλο, όχι μόνο σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Σκοφεράτη. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα προς την κυρία Μονίκ Γκογιάν. Για να είναι πλήρης η προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να έχει στη θέση του όλα τα στοιχεία που αφορούν το προϊόν που, που αποφασίζει να αγοράσει και να το χρησιμοποιήσει. Όλα όσα ε, χρειάζονται ούτω ώστε να γνωρίζει την προέλευση του, του προϊόντος, τους τρόπους με τους οποίους παρασκευάστηκε. Όλα αυτά είναι στοιχεία της ικανότητας των καταναλωτών να επιλέξουν και βεβαίως αυξάνουν και το επίπεδο ασφάλειας. Όμως εδώ υπησέρχονται και άλλα στοιχεία. Αν ξέρω, ας πούμε, ότι ένα ένδυμα παρασκευάζεται από παιδιά, για λόγους ηθικούς και διοντολογικούς, ε, να το αγοράσω. Επομένως, η ανιχνευσιμότητα ενός προϊόντος θα πρέπει να θεωρηθεί ως βασικό εργαλείο για να εξασφαλίσουμε αυτή τη γνώση ε, του καταναλωτή, του ατόμου που αγοράζει αυτό το προϊόν. Η ανιχνεσιμότητα θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαρκώς από κάθε καταναλωτή. Και θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες ε, που είναι σχετικές. Γιατί υπάρχουν πραγματικές τραγωδίες που συμβαίνουν γύρω από αυτά. Παραδείγματο χάρη το δράμα του Μπαγκλαντέ, όπου πέθαναν πάνω από χίλια άτομα στο, στην πρόσφατη στα, τραγωδία. Αλλά δεν είναι η μόνη. Γιατί υπάρχει μία αλυσίδα παραγωγής που λειτουργεί με τελείω τρευλέ ιδέε. Ότι θα πρέπει να παράγει δηλαδή με το χαμηλότερο δυνατό κόστο, ακόμα και αν θέσει σε κίνδυνο την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, ακόμα και τη ζωή του μερικέ φορέ. Αυτό δεν θα με επικεντρωθώ βασικά σε αυτό. Το ανέφερα μόνο και μόνο επειδή σε αυτή την περίπτωση και για λόγου ηθικούς μπορούμε να αρνηθούμε να αγοράσουμε, να χρησιμοποιήσουμε ένα προϊόν επειδή δεν γνωρίζουμε που παρασκευάστηκε αυτό το προϊόν. Η ανιχνευσιμότητα όμως είναι ένα πλεονέκτημα όχι μόνο για τον καταναλωτή αλλά και για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν καταφανείς, ε, παρα, καταφανή παραδείγματα ε, στρεβλού ανταγωνισμού. Συχνά αυτοί που σέβονται τους κανόνες ε, είναι τα θύματα. Είναι αυτοί που τιμωρούνται, που πλήττονται. Θέλω να το καταλάβω. Εγώ σας είπα την ε, γνώμη μου συντομία. Η ανιχνευσιμότητα είναι το βασικό εργαλείο για τον καταναλωτή για να αποφασίσει. Εγώ θέλω να ξέρω πού παράγεται το νερό που πίνω. Γιατί να μην έχω τη δυνατότητα να το μάθω αυτό. Και για ποιο λόγο υπάρχουν ε, αντιρρήσεις ε, ως προς αυτό. Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι ζημία για, τους επιχειρη... τις επιχειρήσεις. Σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Αλλά μιλάω για τις επιχειρήσεις βέβαια που σέβονται τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτο. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι η συγγήτρια ε, για το πακέτο των 8 οδηγιών που αφορούν τη θέση εμπορία προϊόντων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εφαρμογή του πακέτου για την ασφάλεια προϊόντων. Και μιλήσαμε για τα κριτήρια της εποπτείας της αγοράς. Στη διάρκεια όμως του, τριμέρου τριμερούς διαλόγου φαίνεται ότι ε, αποφασίσαμε ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην οριζόντια οδηγία για την ασφάλεια των ε, προϊόντων. Έχω κάποιες επιφυλάξεις ε, γι' αυτό. Φοβούμαι ότι θα μειωθεί το επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων αν υπαχθεί το θέμα της εποπτείας μόνο στην οριζόντια οδηγία. Έχω και ένα άλλο σχόλιο. για το τι θα καλύπτεται από αυτό το νέο κανονισμό ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις όπως ε, τα φάρμακα υπάρχει σαφήνεια, αλλά για ορισμένα προϊόντα δεν υπάρχει τέτοια σαφήνεια. Ίσως θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποια ελάχιστα κριτήρια που θα, εφαρμόζουν, θα εφαρμόζονται και θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα. Έτσι, θα έχουμε πολύ πιο ακριβή νομοθεσία για τα φάρμακα σίγουρα, αλλά κάποιες αρχές περί χνηλασιμότητας ή ε, περί υποχρεώσεων των ε, κατασκευαστών και των διανομέων είναι γενικά και θα πρέπει να ισχύουν στην Ευρώπη για όλα τα προϊόντα. Αυτό ισχύει στις Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα. Αν θέλει κανείς να εξαγάγει προς τις Ηνωμένε Πολιτείες, εκεί οι κανόνε είναι σαφεί και θα πρέπει να του ε, τηρούν οι εισαγωγείς όσοι θέλουν να εξάγουν προς, την, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ε, πιστεύετε ότι μια οριζόντια οδηγία και με γενικές εξαιρέσεις είναι η κατάλληλη προσέγγιση για τέτοιου είδους νομοθεσία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, μερικά από τα θέματα που θίξατε θα καλυφθούν στο δεύτερο τμήμα τη δημόσια ακρόαση που αφορά την εποπτεία τη αγορά. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο σήμα ΕΚ και κατά πόσο θα πρέπει να καταργηθεί. Ε, μερικές φορές ε, οι καταναλωτές δεν το καταλαβαίνουν, είπε η Μόνικα Γκρένς, και μάλιστα συνάδει στη σύγχυση παρά στην ε, σωστή ενημέρωση του σε ένα τέτοιο σήμα. Και ίσω και παραπλανητικό αποτέλεσμα μερικέ φορέ. Θα ήθελα να το εξηγήσει αυτό η κυρία Γκόεν. Θα δώσω τώρα το λόγο στου καλεσμένου μα με την αντίστροφη σειρά, ξεκινώντα από τον κύριο Βάισνερ, μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Προυζέ, τον κύριο Μονφόρ και στο τέλο την κυρία Γκόεν. Ένα δίλεπτο παρακαλώ στον καθένα. Ελπίζω να καλύψετε τις ερωτήσεις στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα για να περάσουμε και στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Ο κύριος Βάισνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, τα γερμανικά, αν μου επιτρέπετε. Ε, για την ερώτηση της κυρίας Σαλτεμόζε, νομίζω ότι δεν έχουμε προτάσει να διατυπώσουμε επί της ε, ουσίας, φυσικά, στις λεπτομέρειες. Ναι, στα ε, μεταχειρισμένα προϊόντα και σε άλλα προϊόντα τα οποία, στα οποία χρειάζεται και ο ορισμός ακόμη να επανεξεταστεί αλλά δεν μπορούσα σήμερα να έρθω με μια μεγάλη με ένα μακροσκελή κατάλογο ε, δεδομένου ότι είχαμε και σχετικά βραχυπρόθεσμα αυτή την πρόσκληση δεχθεί ε, δεν μπορούσα να επεκταθώ πολύ γι' αυτό θέλησα να επικεντρωθώ στα πέντε μου λεπτά στις βασικές αρχές η βιομηχανία επίπλων λοιπόν με όλες αυτές τις περιπτώσεις ε, ευθύνης από προϊόντα, αντικειμενικής ευθύνης από προϊόντα, ε, πιστεύει ότι οι προτάσεις και οι γενικές αρχές καλύπτει τις δικές μας ε, ανησυχίες και μελήματα. Απλώς θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει να υπάρξουν διαφορές ως προς τις ευθύνες. Δηλαδή να μην, έχουμε, να μην καταλήξουμε σε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες θα είναι η μία εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, ε, υπάγονται στην περιφερειακή ενδεχομένω ή πάντως εθνική νόμοθεσία για την αντικειμενική ευθύνη και θα έχουν ε, την υποχρέωση για μια σειρά από δοκιμές, δοκιμασίες να υποβάλουν τα προϊόντα τους, επαληθεύσεις και να παίρνουν την πιστοποίηση και τη διαχείριση ποιότητα που απαιτείται από την εσωτερική νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτή την ε, ασφάλεια στα προϊόντα του και να μπορούν να την προβάλλουν. Και από την άλλη, άλλε επιχειρήσει είτε είναι εισαγωγή, είτε είναι μικρότερε επιχειρήσει ε, των οποίων τα προϊόντα έχουν παραχθεί πιο ρηπού στον κόσμο και για τα οποία ο καταναλωτή δεν είναι σε θέση προκαταβολικά να γνωρίζει εάν ε, την ώρα πάει να κάτσει σε μια καρέκλα και πέσει και χτυπήσει, έχει τη δυνατότητα να κάνει την αγωγή του και να ζητήσει αποζημίωση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να υπάρχει μια αντίστοιχη πρόβλεψη για την διασφάλιση της ποιότητας, για την αποφυγή των κινδύνων. Εμείς μικροί επιχείρησιόντες, έχουμε 30.000 ευρώ το χρόνο για την πιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, για να είμαστε σε θέση, εάν ποτέ κάτι συμβεί ομιγέννητο, να λέμε, ορίστε εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε για να διασφαλίσουμε το του επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας. Βεβαίως έχουμε λοιπόν προτάσεις. Οι προτάσεις μας όμως αυτές δεν έχουν να κάνουν με τις γενικές προτάσεις, με τις γενικές αρχές της ε, νομοθετικής προτάσεως. Και βεβαίως η Συνομοσπονδία θα υποβάλει, φαντάζομαι, λεπτομερέστερες ιδέες για τα παρεπόμενα έξοδα ή δαπάνες που επανέρχονται κατά καιρούς συζήτηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την δήλωση, την ιδέα. θα σας πω το εξής. Εγώ φοράω ένα πουκάμισο όταν το βάζω το πρωί, ξέρω, το έχουν φτιάξει στη Μαλαισία, το έχουν φτιάξει μια μεξικανική επιχείρηση, η οποία όμως έχει ε, το σχεδιασμό στη Γερμανία και άρα μπορώ με αυτά τα κριτήρια να ξέρω εάν είναι καλό να φορέσω το πουκάμισο αυτό ή όχι αν σήμερα ω καταναλωτή άκουγα ότι να, ένα προϊόν, το, το πουκάμισό που είναι φτιαγμένο στον Μπαγκλαντέ, τότε ίσω πέρα από τα όσα έχουμε ακούσει, να έλεγα, ίσω ίσως τελικά να υπάρχει πρόβλημα ω προ την ασφάλεια. Και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να είμαστε αρκετά συνεπεί για να μην αφήνουμε περιθώρια να ε, αποφεύγει κανεί την υποχρέωση για ενημέρωση, για χορήγηση των πληροφοριών σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής, από το πρώτο στάδιο μέχρι τον ε, καταναλωτή, μέχρι το λιανοπολιτή συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ κυρία Προυζέ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω και εγώ τη μητρική μου γλώσσα, τα γαλλικά, για να είμαι και σαφέστερη. Ε, φαίνεται ότι δεν είμαι και πολύ σαφής προηγουμένως και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν ζητούν οι έμποροι υποβάθμιση της ευθύνης, μικρότερη ευθύνη. Το αντίθετο. Σίγουρα ε, έχουμε τις διακρίσεις ε, ε, κατασκευαστής εισαγωγές και μετά διανομές. Με βάση τη δική μας εμπειρία και το νέο νομικό πλαίσιο το γνωρίζουμε μέσω της νέας οδηγίας, της Γενικής Οδηγίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων. Η εμπειρία μας μας έχει δείξει ότι τα κράτη-μέλη, ακόμη και στο εσωτερικό σε μερικές φορές, θετούν διαφορετικές ερμηνείες. Και η Επιτροπή, καλό θα ήταν να ακούσει και αυτή αυτόν τον προβληματισμό, γιατί μερικές φορές ε, θα πρέπει να μιλούμε και για την ασάφεια που υπάρχει. Θέλουμε να είναι σαφείς οι υποχρεώσεις μας. Αν πρέπει να τηρούμε πέντε όρους, να μπορούμε να τους ε, εφαρμόζουμε και να, να εξακριβώνεται η τήρηση αυτών των πέντε όρων. Είναι σαφές λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει να είναι ξεκάθαρες υποχρεώσεις. Και εμείς ως διανομής ε, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες ε, για το προϊόν. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή η τεκμηρίωση εξαντλητική για το κάθε προϊόν ε, περιλαμβάνει κάποια στοιχεία καινοτομία, ε, κάποιες αναφορές ελέγχου. Είναι εμπιστευτικέ πληροφορίε και χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα προϊόν. Δεν τι δίνει ο παραγωγό στο διανομέα. Υπάρχει θέμα εμπιστευτικότητα, υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Μερικέ φορέ υπάρχει και θέμα θέμα του ανταγωνισμού. Οπότε δεν μπορούν οι διανομείς ε, που διαθέτουν σε εμπορία διαφορετικά προϊόντα να ε, γνωρίζουν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες ε, των διαφόρων ανταγωνιστικών προϊόντων. Δεν τις δίνουν οι κατασκευαστές ή οι παραγωγοί. Γι' αυτό ζητήσαμε μια εξισορρόπηση των ευθυνών, ώστε ο καθένας να αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί. Επίσης, άκουσα ότι με το πακέτο αυτό θα πρέπει να μειώνεται η ευθύνη στην Ευρώπη λογοδοσία. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχαμε σε ένα σεμινάριο για την ανάλυση κινδύνων και αύριο θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση κινδύνου για κάθε προϊόν που τίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά ως παραγωγή και για τα μη εναρμονισμένα προϊόντα. Ανάλυση κινδύνου προϋποθέτει τεράστια έξοδα γιατί καλύπτει το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη φάση πριν την θέση εμπορία πρέπει να καθορίζονται όλοι οι πιθανοί δυνητικοί κίνδυνοι προϊόντος με βάση τη σύνθεσή του με την κατάρτιση κάποιων σενάριων. Είναι μια εξαιρετικά επαχθής διαδικασία αυτή η ανάλυση κινδύνου. Βέβαια, πρόκειται για μια νέα υποχρέωση που, κατά τη γνώμη μου, αυξάνει το επίπεδο ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση δεν το μειώνει. Σε ό,τι αφορά την προέλευση. Τεράστια συζήτηση για το θέμα τη προέλευση. Επαναλαμβάνω. Εμείς ε, δεν μιλούμε εδώ για την προέλευση των προϊόντων, αλλά για το πακέτο ασφάλειας των προϊόντων. Και ε, σίγουρα οι τελωνιακοί κανόνες ε, και το κατά πόσο θα συνάδουν στην αδιαλέπιση της δεν είναι βέβαιο. Εγώ πιστεύω ότι η προέλευση αφορά τους κανόνες δασμολόγησης. Και μόνο τα εισαγόμενα προϊόντα θα έχουν το made in. Αλλά για το ίδιο προϊόν μπορεί να παράγεται στο ίδιο εργοστάσιο ή να έχει δύο διαφορετικές προελεύσεις. Ανάλογα με τη μεταποίηση. Αυτό μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή η ανάφορα της ε, προέλευσης και να παραπλανήσει και τις ε, αρμόδιες αρχές. Αυτό λένε οι έμποροι. Το θέμα δεν είναι αν θα πρέπει να ενημερώνουμε τον καταναλωτή για την προέλευση των προϊόντων. Αυτό είναι άλλη, άλλο Ευαγγέλιο, άλλη συζήτηση. Αλλά σίγουρα για την ασφάλεια η αναφορά της προέλευσης δεν είναι ε, εργαλείο ιχνηλασιμότητας. Έχουμε άλλα πολύ πιο χρήσιμα εργαλεία ιχνηλασιμότητας. Τώρα, για τις κατεξουδιώτες πράξεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με διαβούλευση, προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, με τους επαγγελματίες. Και διεκδικούμε συμμετοχή στο EMSF. Πάμε, αλλά ο χρόνος έχει λήξει και ήμασταν υπερβολικά γενναιόδοροι. Θα ήθελα να σα δώσουμε και άλλο χρόνο, αλλά δυστυχώ τέθηκα τόσε πολλέ ερωτήσει. Ο κύριο ε, Μονφόρ. Όντω, πολλέ και εύστοχε ερωτήσει για την συμμόρφωση και την ασφάλεια. Ερώτηση που τέθηκε από πολλού. Ε, το θέμα τη ε, συμμόρφωση προέρχεται από την οδηγία για τα αγωθά. Αφορά την απέτηση ετικετοθεσία, σήμα κτλ. Και ε, νομίζω ότι ο κανονισμό ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων είναι πολύ καλό και αναφέρει ότι αν δεν υπάρχει συμμόρφωση ή τεκμήριο, θα πρέπει να υπάρχει τεκμήριο ε, για την ασφάλεια και θα πρέπει να εξακριβωθεί. Δεν λέω ότι είναι κακό το κείμενο του κανονισμού. Απλώ ε, σα ακούω τον κόδωνα του κινδύνου ε, για την περιπλοκή αυτών των διατάξεων που μια τέτοια περιπλοκή ίσως δημιουργήσει σύγχυση όσους καλούνται να το εφαρμόσουν να δημιουργήσει πρόβλημα ασφάλεια σε ένα προϊόν που δεν είχε αρχικά θέμα ασφάλεια, μόνο εξαιτία του θέματο συμμόρφωση. Να μην μπερδέψουμε την αγορά. Καλύτερα να έχουμε έναν απλό συγκριτικό κανόνα παρά να περιπλέκουμε τον κανονισμό με τέτοιου είδου προβλήματα όπω αυτό τη ε, συμμόρφωση. Ό,τι αφορά την αρχή τη προφύλαξη. Εγώ δεν θεωρώ ότι μια άμεση ε, μνήμα της αρχής προφύλαξης στο κείμενο θα βελτιώσει κάτι. Γιατί ε, ε στο στον, στην εκτίμηση του κινδύνου που θα πρέπει να κάνουν οι εταιρείε εμπεριέχεται αυτή η αρχή της προφύλαξης. Αναφέραμε το παράδειγμα της καρέκλας που πέφτει κάποιος από μια καρέκλα και τραυματίζεται και θα πρέπει να ξέρουμε γιατί συνέβη κάτι τέτοιο, γιατί δημιουργήθηκε αυτό το ατύχημα και μπορούμε να έχουμε διαφορετική αξιολόγηση ανάλογα με την πιθανότητα δημιουργία τέτοιου ατυχήματο. Και εκεί ισχύει η αρχή τη προφύλαξη. Αν οι αρχέ γνωρίζουν ότι κάτι συνέβη, κάτι υπήρχε σε αυτή την καρέκλα, το αυτοκίνητο λοιπά το προϊόν, μπορούν να είναι σίγουρες ότι ε, ο κίνδυνος έχει υπερκεραστεί αν ε, φροντίζεται για την ασφάλεια των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και την αρχή της προφύλαξης. Παραλαμβάνω, η αρχή της προφύλαξης είναι εγγενής, ε, εμπεριέχεται έμεσα στον κανονισμό αυτό. Δεν χρειάζεται να αναφέρεται ρητά γιατί ίσως δημιουργήσει παρερμηνίες. Τώρα, ε, τα καταναλωτικά προϊόντα σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Τα βιομηχανικά προϊόντα καλύπτονται από το πακέτο υποπτία τη αγορά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήδη αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Τώρα, ίσως θα πρέπει να, γίνει, να καταργηθεί η διάκριση μεταξύ εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων προϊόντων. Θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι προδιαγραφέ για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα απλοποιήσει την νομοθεσία. Αυτή η διάκριση μεταξύ εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων δεν είναι σωστή. Αυτά και ευχαριστώ. Και τελικά η Μόνικ Γκόιενς. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σαφή ω προ την προοπτική του καταναλωτή για την ε, επισήμανση προέλευση. Σήμανση πρόελευση, δεν θα συμφωνήσω ε, οι περισσότερες πληροφορίες δίνουν πιο πολύ διαφάνεια μόνο όταν είναι εύστοχες οι πληροφορίες, δεν έχουν νόημα. Και η σήμανση προέλευσης ε, δεν έχει νόημα αν είναι περίπλοκη και συγχαίει την εικόνα για τον καταναλωτή. Δεν είναι αυτό ευφύη νομοθεσία γιατί θα φέρει περισσότερο κόστος για τη βιομηχανία και καμία προσθεμένη αξία για τον καταναλωτή. Από τη δική μα την προοπτική το ίδιο. Είναι σαφές αυτό. Για τα, ε, όχι για τα τρόφιμα βέβαια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε στον τομέα εκτός τροφίμων, γιατί στα τρόφιμα γίνεται ο αγώνας βέβαια να ξέρουμε που προέρχονται, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά συστατικά κομμάτια, εξαρτήματα, τμήματα στα προϊόντα που παράγονται ανά τον κόσμο, που είναι αδύνατον ουσιαστικά να δώσουμε στοιχεία ε, καθοριστικά ε, σαφή για την προέλευση ενό ε, βιομηχανικού προϊόντος και επίση αν το περιλάβατε στο κείμενο θα πρέπει να προβλέψετε και τι σχετικέ αρχέ, οι οποίε θα εποπτεύουν την τήρηση. Αυτή τη στιγμή ακόμα και για τα ζητήματα τη ασφάλεια τροφίμων έχετε περιορισμού στον προπολογισμό για τι αντίστοιχε αρχέ. Ε, γιατί λοιπόν να προβλέψετε και άλλα καθήκοντα σε αρχέ, που έχουν προτεραιότητε που ακόμη δεν έχουν μπορέσει να υλοποιήσουν. για την αρχή προφύλαξη ε, νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει στο κείμενο. Γιατί να φύγει, αφού υπήρχε στο αρχικό κείμενο, έχει πολύ μεγάλη ασία, αξία για την προστασία του καταναλωτή αλλά και για τι εταιρείε. Ένα χρήσιμο εργαλείο όπω και για τι ε, δημόσιε αρχέ οι οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση, ακόμη και αν υπάρχει χαμηλό επίπεδο στατιστικών για ατυχήματα, να παρέμβουν, γιατί το ότι δεν υπάρχουν στατιστικές δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Μπορεί να, έχει προβλέψει, να μην έχει προκύψει ατύχημα, αλλά πολύ μακροπρόθεσμα να προκύπτει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Άρα λοιπόν πρέπει να το προβλέψουμε στο κείμενο ως ένα πυλώνα πάνω στον οποίο θα μπορούν οι δημόσιες αρχές να στηρίξουν τη δράση τους για την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ τους ειδικού μας και του συναδέλφους που μίλησαν. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα περισσότερα θέματα. Αν μα περισσέψει ο χρόνο φυσικά μπορείτε να συμμετάσχετε και στο επόμενο τμήμα της συζητήσεω ε, που θα ακούσουμε και περνάω αμέσω σε αυτό για την ε, εποπτεία στην αγορά το, έχει το θέμα αυτό η κυρία Πιετικά, έναν η οποία όμως χρειάστηκε να αποχωρήσει για μια κατεπίγουσα υποχρέωσή της ε, στην οικονομική επιτροπή. Θα χρειαστεί να αποχωρήσει μια κατεπίγουσα υποχρέωση στην ε, Επιτροπή των ε, Οικονομικών. Θα ακούσουμε τους ειδικού μας. Κύριο Στίβεν Ράσελ, γνωστός γνώριμ, παλιός γνώριμος από την ΆΝΕΚ ομάδα καταναλωτών που αναλαμβάνει το συντονισμό των δραστηριοτήτων των σχετικών με την τυποποίηση, με τα πρότυπα. Ο κύριος Φανμπούρεν θα έλεγα ότι κάνει έρευνα αγοράς, είναι ερευνητής αγορών, αν και δεν ξέρω αν ισχύει αυτός ο όρος, για την ε, προστασία ε, των, καταναλωτών ή, εν πάση περιπτώσει, εμπορικές προδιαγραφές στον τόπο, στο χώρο ε, πλην τροφίμων, εκτός τροφίμων, τον καλωσορίζουμε, ο κύριος Κούμπερχ Φαντεμπράχ από την ε, Business Europe, εμπειρογνώμονας της Philips, ο κύριος Σλάιερ, η κυρία Σλάιερ, Αλεξάνδρα Σλάιερ, από την Ένωση Μηχανουργικών Βιομηχανιών, και θα δούμε αν ε, μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη συμφωνία που προκύπτει εκεί. Και η κυρία Βόικτ, Γενικός, Γενική Διευθύντρια, Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την Ενέργεια και το Περιβάλλον. Να δούμε αν έχει να μας πει και εκείνη κάτι. Έχετε πέντε λεπτά έκαστος. Ο Στίβεν Ράσιλ πρώτος. Και έχετε και τις διαφανίες σας, οποίες θα προβάλλουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να τα καταφέρω με το μηχάνημα. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ θέλουν ασφαλή προϊόντα και οι επιχειρήσει θέλουν ε, δίκαιο ανταγωνισμό. Απλά πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει πραγματική εποπτεία τη αγορά και εφαρμογή των ε, νομοθετημάτων. Υπάρχει πρόβλημα. Το, γι' αυτό τον Απρίλιο του 2009 ε, δημοσιεύθηκε μια έκκληση προ τα θεσμικά όργανα, ώστε να υπάρξει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για την εποπτεία τη αγορά. Ε, υποτίθεται ότι με αυτές τις θέσεις προσπαθούμε ακριβώς να ανταποκριθούμε σε αυτή την έκκληση. Θα περιοριστώ λοιπόν σε κάποια γενικά σχόλια σήμερα ε, ακριβώς για αυτό το θέμα. Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι η εποπτεία της αγοράς θα τους ε, προστατεύσει από την αγορά μη ασφαλών προϊόντων. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Σημαίνει αυτό το, αυτή η έννοια σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικά, διαφορετικές χώρες. Ε, η εποπτεία της αγοράς είναι ευθύνη των κρατών μελών. Και απλώς πρέπει να, εφαρμοστούν οι, πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία και τα κοινά πρότυπα. Ε, επομένως, στα πιο ασθενή μέλη ε, έχει σημασία κατά πόσον εποπτεύεται η, αγορά. δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά νομοθετικά εργαλεία μέχρι το 2008 που να ασχολούνται με την ε, εποπτεία της αγοράς και οι υποχρεώσει των κρατών μελών είναι να αποσύρουν τα επικίνδυνα προϊόντα από την αγορά, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε μία συνεπή προσέγγιση σε όλες τις χώρες για την εποπτεία της αγοράς. Ούτε οι πόροι που υπάρχουν σε, σε διάφορα κράτη-μέλη, τα θέματα, α, οι δεσμεύσεις αυτές δεν είναι αυτές που κερδίζουν από αυτές που κερδίζουν ψήφι. Το Οκτώβριο 2009 έγινε μια μελέτη που έδειξε ότι τα περισσότερα κρατημέλη δεν δίνουν περισσότερου πόρου παρά το γεγονό ότι υιοθετήθηκε ο κανονισμό 765. Αν θέλουμε ένα παράδειγμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αρχέ τη εποπτεία αγορά, είναι η εφαρμογή της απόφασης ε, της Κομισιόν για την ασφάλεια των αναπτύρων. Είναι ένα ε, γνωστό παράδειγμα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Με βάση την Κομισιόν ε, έχουμε 40 θανάτους και 900 ατυχήματα στην Ευρώπη από αναπτύρες και τα θύματα είναι παιδιά. υποτίθεται ότι υπάρχει το νομοθέτημα, η απόφαση μάλλον, και έπρεπε μέχρι το, το 2008 να είχαν αποσυρθεί οι επικίνδυνοι αναπτήρες. Παρ' όλα αυτά, το 76% των αναπτύρων, όπως ε, ελέγχθηκαν από την ProSafe, το Φεβρουάριο του 2010 δεν είχαν αποσυρθεί το 76% των μη συμμορφούμενων αναπτήρων δεν έχουν αποσυρθεί. Τώρα, ε, η νέα νομοθεσία θέλει να καλύψει τα κενά του 765, αλλά πηγαίνει αρκετά μακριά. Μερικές, υπό κάποιες έννοιες πηγαίνει πολύ μακριά. Οι πόροι που υπάρχουν τώρα στις αρχές εποπτείας της αγοράς ε, δεν είναι επαρκείς ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την καθαρότητα της αγοράς από επικίνδυνα προϊόντα όπως ε, οι μη συμμορφούμενοι αναπτήρες. Ε, επεκτείνεται όμως και στην ασφάλεια των προϊόντων, στην, προστασία, στην ασφάλεια των εργαζομένων, στην προστασία του περιβάλλοντος. Καλά όλα αυτά, αλλά από πού θα προκύψουν τα χρήματα, οι απαραίτητοι πόροι που χρειαζόμαστε και πώς. Ε, υποτίθεται ότι τα τέλη θα είναι επαρκή για το σύστημα, αλλά λέει, λέει ΑΝΕΚ. Επίσης είμαστε ε, απογοητευμένοι που η αρχή της προφύλαξης δεν, αντι, δεν αντικατοπτρίζεται στο MSR, ε, γιατί είναι πυλώνας της προστασίας στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Χρειαζόμαστε μία αναφορά στο MSR και στο CPSR. Ε, η σήμαση της προέλευσης. Ακόμα κάτι που πρέπει να εφαρμόσουν οι αρμόδιες αρχές. Και βεβαίως μην, ξέρετε, μην ξεχνάτε ότι μπορεί να φαλκιδευτεί όπως οποιοδήποτε άλλο σήμα. Επίσης, ε, το MSR δεν ε, επιτηρεί την ε, ψηφιακή αγορά και τις ε, πωλήσει στο ίντερνετ. Ε, χρειαζόμαστε επίσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια βάση δεδομένων για τα ατυχήματα για λόγους ασφάλειας. Τα κράτη-μέλη το μόνο που ενδιαφέρονται όμω είναι να μάθουν πόσο θα κοστίσει αυτό. Μην το βλέπετε ω κόστο, να το βλέπετε ω επένδυση στην ασφάλεια. Θα ανακτήσουμε αυτέ τι δαπάνε ε, γιατί θα μειωθούν τα, τα έξοδα από ατυχήματα κτλ. Νομίζουμε ότι μόνο με 7,5 εκατομμύρια ευρώ μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη βάση δεδομένων για τα ατυχήματα. Και πιστεύουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή στην εκνομοδότησή τη για τον κανονισμό υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Η Ευρώπη μπορεί να έχει την καλύτερη νομοθεσία, μπορεί να έχουμε τα καλύτερα πρότυπα, πρόεδρε. Αλλά χωρί εφαρμογή, τι νόημα έχουν αυτά, είναι άχρηστα. Και ω καταναλωτέ δεν θα πρέπει να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Σάιμον ο συνήθως ε, πολύ οξυδερκής ε, και με στέση παρατηρήσεις Τώρα, τι γνώμη έχουν οι αρχές εποπτείες αγοράς ε, μετά την σχετικά ζωφερή ανάλυση της ΕΝΕΚ για το μέλλον και πώς, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί. Κύριε Βανμπύρεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια αναδρομή στο νέο πακέτο για την εποπτεία το, της αγοράς υπό το πρίσμα των οργανώσεων εποπτείας αγοράς. Τι θα συμβεί λοιπόν μετά την εισαγωγή του πακέτου. Καταρχήν να δώσω θερμά συγχαρητήρια στις δύο Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΣΑΝΚΟ και Επιχειρήσεων γιατί είχαν το θάρρος να καταλήξουν σε μια πολύ καλή νομοθετική πρόταση συγχωνεύοντας τις δύο προηγούμενες. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, συνδύασαν πάρα πολλά σημεία. Εγώ θα περιοριστώ σε τέσσερα από αυτά. Στο νέο πακέτο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδύασε τον έλεγχο στα σύνορα, την εποπτεία στις αγορά, στην αγορά, την εποπτεία, την πιστοποίηση και τα αιτήσια σχέδια των κρατών μελών. Πολύ σημαντικά αυτά τα σημεία και δίνει σε εποπτικές αρχές ε, πολλές νέες δυνατότητες σε αυτό το νέο πακέτο. Θα αναφερθώ σε τρεις ή τέσσερις από αυτές τις νέες δυνατότητες. Φυσικά, πολύ σημαντικό για μας είναι η εισαγωγή του, της υποχρεωτικής βάσης δεδομένων για τα προϊόντα πλήν των τροφίμων, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στο έργο μας. Γιατί είδατε τι έγινε στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τη στιγμή που ελέγχονται τα προϊόντα και θεωρείται ότι συμμορφώνονται, δεν χρειάζεται και οι Ολλανδικές αρχές να ελέγξουν τα προϊόντα. Ε, ο δεσμευτικός χαρακτήρας, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της βάσης είναι πολύ καλό στοιχείο. Επίσης, ε, τα εργαστήρια αναφοράς θα βοηθήσουν πολύ τις εποπτικές αρχές της αγοράς, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές τέτοιες εποπτικέ αρχές που δεν έχουν όμως ε, εργαστήρια αναφοράς για τα προϊόντα πλην των τροφίμων. Κάτι που δημιούργησε σφοδρές συζητήσει για τα αποτελέσματα, τα πορίσματα ε, τέτοιων εργαστήριων. Σίγουρα αν έχουμε εργαστήρια αναφοράς θα, θα βοηθήσουν σε περίπτωση αντιδικίας ή διαφωνίας μεταξύ εποπτικών αρχών. Επίση, ε, θέμα κατανομής. Ο νέο κανονισμό μα δίνει την ε, δυνατότητα επιβολής ε, τελών για τα μη εναρμονισμένα προϊόντα, τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί τέτοιες συνεισφορές χρειάζονται και 70% των προϊόντων που ε, συνδέουμε στο λιμάνι του Ρότερνταμ δεν, είναι, δεν τηρούν τις διατάξεις. Οπότε θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικές οι αρχές αν μπορούν να απαιτήσουν την καταβολή τελών από τους εισαγωγείς τέτοιων προϊόντων. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στη σύσταση δύο ομάδων, του IMP για την εποπτεία της αγοράς και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Εποπτείας Αγοράς, του EMSF. Και οι δύο ομάδες δίνουν την ευκαιρία σε εμά, τις εποπτικές αρχές, αλλά και στα κράτη-μέλη, τη δυνατότητα να συζητούν τα αιτήσια αμοιβαία του σχέδια, τη στρατηγική τους για την εποπτεία αγορά και να συνδυάσουν τις δράσεις τους. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εποπτής Αγοράς συζητάται μόνο στην ομάδα εργασίας των εποπτικών αρχών που δίνει μόνο ένα φόρουμ ε, για τις εποπτικές αρχές. Τώρα έχουμε δύο τέτοιες ομάδες εργασίας, δύο τέτοια φόρουμ και έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε και για τα εναρμονισμένα προϊόντα. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα για το πώς ε, λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Χθες είχαμε μια συνεδρίαση για τη σήμαση σε προϊόντα ενέργειας. Πόσα κράτη-μέλη λοιπόν ε, ε, έχουν ήδη εφαρμόσει αυτή την οδηγία για την σήμαση των προϊόντων ενέργειας. Πέντε Έξι, 7 το πολύ. Καμία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Δεν λειτουργούν λοιπόν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ούτε γίνεται καμία συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για το ποιο θα επενδύσει τι και ποιο θα ελέγξει τι. Εμεί θα ελέγξουμε και τα γερμανικά προϊόντα ή θα επικεντρωθούμε μόνο στα ολλανδικά προϊόντα. Και δεν χρησιμοποιείται καθόλου η δάση δεδομένων. Οπότε ε, οι οργανώσεις εποπτικών, εποπτής αγοράς δεν μπορούν να αξιοποιήσουν ε, τις διάφορες εμπειρίες, ούτε να τις ανταλλάξουν. Επίσης, ε, έχουμε ανεξάρτητες διαδικασίες δοκιμασίας των προϊόντων και οι δοκιμές, οι έλεγχοι είναι πολύ δαπανηροί. Εμείς κάνουμε τέτοιους ελέγχους στα δικά μας εργαστήρια και 2.500 ευρώ πετούνται για να ελεγχθούν μόνο 50 δείγματα ένα ελάχιστο τμήμα δηλαδή των προϊόντων στην αγορά. Και επίσης, στην ομάδα για την ε, σήμανση της ενέργειας δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων. Τι βελτιώσει λοιπόν θα πρέπει να γίνουν από την ομάδα αυτή. Τι βελτιώσει μάλλον μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο νέο της πακέτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει τέτοιους ελέγχους, αλλά θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προσέξει τη διατύπωση του άρθρου που είναι πολύ γενικό και όριστο προς το παρόν. Και σίγουρα η δεσμευτική έλεγχη ε, και για τα προϊόντα τροφίμων ε, χρειάζονται γιατί έτσι ευθυγραμμίζονται οι έλεγχοι για τα προϊόντα αυτά με, τα, με τους ελέγχους για τα τρόφιμα. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν ε, και ποιος θα πληρώσει την, ε, τους ελέγχους αυτούς. Επίσης, ε, η διοργάνωση κοινών δράσεων. Να γίνεται όχι μόνο για τα μη εναρμονισμένα, αλλά και για τα εναρμονισμένα προϊόντα. Και η χρήση του IS, ICSMS θα πρέπει να γίνεται από όλα τα κράτη-μέλη για να το φροντίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, οι αρχέ υποπτήρες αγορών θα πρέπει να είναι και πολύ δημιουργικέ ω προ την επιβολή κυρώσεων. Χθε έμαθα από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι εκτός ότι επέβαλαν πρόστιμο σε έναν παραγωγό και εισαγωγέ για μη ε, ε, συμβατά προϊόντα, θα πρέπει ο εισαγωγέ να πληρώσει και τον την περιβαλλοντική ζημία με αποτέλεσμα να είναι πολύ υψηλό και υπέροχο αυτό το πρόστιμο. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Και θα έχουμε και θέματα να απαντήσουμε μετά. Ας ακούσουμε από πλευράς των παραγωγών. κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους οργανωτές που μας προσκάλεσαν να συζητήσουμε εδώ την Business Europe. Ε, θα ήθελα να πω ότι εν γέννη μας ε, φαίνεται καλή αυτή η πρόταση. Θέλουμε να έχουμε ε, καλά προϊόντα στην αγορά με εμπιστοσύνη του καταναλωτή και με ε, ασφάλεια. Άρα πρέπει να ενισχυθεί η εποπτεία της αγοράς. Η απλούστευση βεβαίως είναι σημαντική, θα οδηγήσει σε ανάπτυξη, θα έχουμε χαμηλότερο κόστος για την συμμόρφωση και ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών. Και όταν είναι χαμηλό το κόστος θα έχουμε και καλύτερη συμμόρφωση. Άρα θα προτείναμε περισσότερη απλούστευση και όχι τροπολογίες που θα περιέπλεκαν τις διατάξεις. Δεν θα χρησιμεύσει τίποτα να περιπλεκούν οι διατάξεις. Έχουμε καταθέσει προτάσεις μας στο έγγραφό μας, θα αναφερθώ σε κάποια βασικά ζητήματα και καταρχάς το πεδίο εφαρμογής η εποπτεία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για τα προϊόντα και όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά ζητούμε σαφείς ορισμούς, γιατί πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ του κινδύνου στην ασφάλεια και των άλλων ε, μη σχετικών ζητήματων, αλλά θα πρέπει επίσης να έχουμε και μια διαβάθμιση του κινδύνου, σαφή, και το, τη διάκριση τη μη συμμόρφωση του προϊόντος του ίδιου από την τυπική μη συμμόρφωση, γιατί χωρίς να είναι αυτή ασήμαντη είναι διαφορετική κατηγορία μη συμμόρφωση. Και επίσης δυστυχώς η αξιολόγηση κινδυνού όπως την έχουμε τώρα δεν είναι ικανοποιητική πρακτική. Καταλήγουν δηλαδή διαφορετικά κράτη σε διαφορετικά αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα το οποίο ακούστηκε και νωρίτερα ε, σε έναν βαθμό. Ένα μοντέλο ε, αναπτήρα που, βρέθηκε, που ασφαλές στην Ελλάδα, κρίθηκε μη ασφαλές στις κάτω χώρες, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος άδικο, είναι καλό να κοιτάξουμε να καταλήγουμε σε κοινέ ερμηνείε, γιατί το αντίθετο οδηγεί σε προβλήματα και στην αγορά και βεβαίω προ την ασφάλεια του καταναλωτή και ω προ την δραστηριότητα του παραγωγού. ή δε εγκάρσια συνεργασία, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, και αξιολόγηση των εκτιμήσεων συμμόρφωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μας βοηθήσει πολύ. Ε, ένα φόρουμ που θα βοηθούσε στην εμπλοκή των ε, φορέων της αγοράς, θα βοηθούσε πολύ στην διευκρίνηση των θεμάτων το θέμα της ανάληψης δράσης από τις αρχές, σε περίπτωση όπου υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης, αλλά αποδεικνύεται ότι ένα προϊόν δεν συμμορφούνται τελικά, ανοίγει πόρτες σε αυθαίρετες εκτιμήσεις και μέτρα δυσανάλογα βαριά. Πρέπει φυσικά να έχουν οι αρχές την ευχέρεια να αξιολογήσουν αυτόνομα το κίνδυνο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ε, αιτιολογούν τον λόγο για τον οποίο παρεμβαίνουν και ε, παρεκτιμούν ένα προϊόν. Και επίσης θα θέλαμε καλύτερες διαδικασίες αποκατάστασης, γιατί με μόνη την αγωγή στα δικαστήρια που κρατάει χρόνια και που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις. Θέλουμε, χαμηλότερες, ε, θέλουμε πιο ταχύες διαδικασίες και πιο απλές αλλά και φθηνές. Η εποπτεία στην αγορά λοιπόν δεν έχει επαρκή σπόρους και θέλουμε να εκφραστεί η πολιτική βούληση για τη χρηματοδότησή της, αποτελεσματική και ουσιαστική οργάνωση, ε, εξοπλισμός αλλά και αρμόδιες αρχές γνωστές που να ώστε να ξέρουμε ποιος εφαρμόζει τον νόμο. στις ε, κυρώσεις και πρόστιμα δεν θα πρέπει οι αρχές ε, σε περίπτωση που αυτά είναι πολύ ψηλά να τα δουν ως κίνητρο για να αναλάβουν δράση μόνο και μόνο για να έχουν μεγαλύτερο όφελος. Και θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο αποδέκτη του αν λόγω Θα πρέπει τα πρόστιμα να είναι αποθαρρυντικά, αποτρεπτικά και αναλογικά και να αφορούν ουσιαστικά προβλήματα συμμόρφωσης και όχι κάποιο τυπικό σφάλμα στην τεκμηρίωση. Και αυτά δεν πρέπει να μπαίνουν στον ίδιο τον κανονισμό, αλλά στα παραρτήματα. Αποτελεσματικότητα επίσης, παλήθευση από εργαστήρια, όλα αυτά θα πρέπει να υποστούν ε, τη δικασία της πιστοποίησης. Καθώς είναι πολλά τα εισαγόμενα προϊόντα και τα προβλήματα συμμόρφωσης που σχετίζονται με αυτά θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι στα σύνορα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει καθυστερήσεις αδικαιολόγητε στα σύνορα και επιβάρυνση αυτών των προϊόντων. Οι προτάσεις για καλύτερη συμμόρφωση δεν μας βρίσκουν σύμφωνος και εάν η υποχρεωτική επαλήθευση διευρυνθεί ο καλοπροαίρετος προμηθευτής θα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση και θα πρέπει να πληρώνουμε τον τρίτο επαληθευτή της συμμόρφωσης χωρίς να γίνονται πιο ασφαλή τα προϊόντα. Οι προϋποθέσεις για επαλήθευση της συμμόρφωσης και η παροχή των πληροφοριών θα πρέπει να διαμορφωθεί με εμπλοκή και διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ευχαριστούμε πολύ. Um, Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Σλάιφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην ακρόαση σας. Εγώ εκπροσωπώ την, τις ε, εταιρείες μηχανικών και μηχανολογίες. Τα περισσότερα μας προϊόντα εμπίπτουν στεναρμονισμένα. αρμονισμένα η εποπτεία των αγορών για μας, για τους κατασκευαστές μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο υπό το πρίσμα των ασφαλών προϊόντων, αλλά και υπό το πρίσμα της ανάγκης συμμόρφωσης ε, και με, τι με, τα περιβαλλοντικά με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, γιατί εκεί ανακύπτει και ζήτημα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Γι' αυτό και η εποπτεία της αγοράς για μας είναι όλο και πιο σημαντική. Και χαιρετίζουμε κάθε πρωτοβουλία που θέλει να καταστήσει πιο αποτελεσματική και αποδοτική την εποπτεία της αγοράς. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ των στόχων του νέου πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη ακούσαμε ότι σας ενδιαφέρουν οι επιφυλάξεις και οι ανησυχίες μας. Έχουμε πολλές και διάφορες στο έγγραφο μας. Εγώ θα επικεντρωθώ στις πιο σημαντικές, που είναι η ιδέα της συμμόρφωσης και του κινδύνου. Η νέα πρόταση κανονισμού, κατά τη γνώμη μας, παραμελεί και διαφορεί για την ανάγκη του ελέγχου της συμμόρφωσης προϊόντων, ε, προτιμώντας ε, την ε, αξιολόγηση του κινδύνου. Δεν ξέρουμε α, πώς, α, θα πώς είναι δυνατόν να γίνονται ανεξάρτητοι έλεγχοι αξιολόγησης του κινδύνου. Δηλαδή, οι εποπτικές αρχές να αποφασίζουν το κατά πόσο ο παραγωγός έκανε σωστά τον έλεγχο συμμόρφωσης και την αξιολόγηση του κινδύνου. Δεν πρέπει και οι δύο ξεχωριστά να κάνουν τους ελέγχους. Και μόνο αν υπάρχει πρόβλημα ε, θα να γίνει αξιολόγηση του κινδύνου της μη συμμόρφωσης από την εποπτική αρχή. Εμείς θέλουμε να ελεγχιστοποιηθεί το διοικητικό άχθος ε, για τους ε, φορείς της αγοράς, τους ε, εμπορικούς παράγοντες και συμφωνώ με τον συνάδελφο της Eurocommerce. Υπάρχουν στην πρόταση κάποιες απαιτήσει που είναι υπερβολικές. Είναι εύκολο να ζητούμε περισσότερες σημάσεις και πληροφορίες και μεγαλύτερε ετικέτε, αλλά μην ξεχνάτε ότι πίσω από την απέτηση αυτή κρύβεται μια ολόκληρη διαδικασία επαχθή. και δεν είναι εύκολη η θέση εμπορία ενό προϊόντος από μια εταιρεία. Υπάρχει πολύ έργο που ε, προαπαιτείται. Επίση, το θέμα τη προέλευση του προϊόντο. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να συζητάνε οι αποπτικέ αρχέ με τον διαχειριστή μια επιχείρηση ενό εργοστασίου στο Μπαγκλαντές ή στην Κίνα. Έχουν ένα ε, πρόσωπο επαφής και νομίζω ότι πιο σημαντικός είναι ο παραγωγός. Γι' αυτό και εφαρμόζεται τώρα το ευρύτερο πακέτο για την ασφάλεια των προϊόντων. Οι καταναλωτές ε, δεν ξέραν να θα αγοράσουν ένα κινέζικο προϊόν ε, εφόσον έχει ένα ευρωπαϊκό σήμα και υπάρχει και ένα σύστημα ελέγχου πίσω από αυτό. Είναι δύσκολο άλλωστε να υπολογιστεί αυτή η ένδειξη προέλευσης για πολύ περίπλοκα προϊόντα. Γιατί μιλούμε για, για ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, ε, για ένα πλυντήριο ή για κάτι περίπλοκο που αποτελείται από ε, τμήματα που μπορεί να παράγονται σε διαφορετικά μέρη. Επίσης, απέτηση επιστοποίησης. Καταλαβαίνουμε αυτό το πειρασμό που υπάρχει, αλλά η επιστοποίηση επισης απετηση επιστοποιηση καταλαβαινουμε αυτο το πειρασμο που υπαρχει αλλα η επιστοποιηση ειναι ε, εργαλείο πριν τη θέση εμπορία, ενώ η εποπτεία είναι εργαλείο για μετά τη θέση εμπορία. Σε καμία περίπτωση η πιστοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εποπτεία της αγοράς, γιατί και η πιστοποίηση αλλά και τα σήματα μπορούν να άνετα να φαλκιδευτούν, να, να παραποιηθούν. Μπορεί να το κάνει ένα έμπορος άνετα. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ του εργαλείου της εποπτείας της αγοράς. Θεωρούμε ότι η εποπτεία της αγοράς θα βελτιώσει την εφαρμογή των ε, προτάσεων που δίνουμε και στο 678, δηλαδή τη συνεργασία των αρχών εποπτείας αγοράς, αλλά και τη συνεργασία των εποπτικών αρχών, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τα τελωνία. Θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε στο φόρουμ αυτό, ιδιαίτερα για την κατάρτιση καταθεντήριων γραμμών. Η εμπειρία αυτή ε, ήταν πολύ επιτυχής στις ομάδες εργασίας για τις διάφορες οδηγίες. Και τέλος, χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι κέριος παράγοντας. Ήδη υπάρχει πρόταση για την επιβολή τελών, συμφωνούμε με την πρόταση αυτή, και ας μην ξεχνούμε και τις κυρώσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις να είναι αποτρεπτικές και αναλογικές. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης. Δηλαδή, ε, να μην έχουμε επιχειρηματικά μοντέλα που θα στηρίζονται στα μη συμμορφω... Ε, τα προϊόντα που δεν ε, συμμορφώνονται με τους κανόνες. Θα πρέπει η κύρωση να εξαρτάται από τη σοβαρότητα της παράβασης και όχι από το μέγεθος του, της επιχείρησης. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που πολύ ξεκάθαρα μας παρουσιάσατε κάποια θέματα τα οποία μας βοηθούν. Ακριβώς γι' αυτό κάνουμε και την ακρόαση εξάλλου. Η Ανδρέα Βόιτ για πέντε λεφτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε σε αυτή την ακρόαση. Θα σας περάσω στον κόσμο της ψήξης, θέρμανσης, που είναι ένας πολύ ειδικό τομέας και επηρεάζει την καθημερινότητά μας σχεδόν σε όλους τους τομείς. Ε, εκπροσωπώ τους κατασκευαστές ε, εξοπλισμού, ψήξης, θέρμανσης και ε, κλιματισμού. Ε, η θέρμανση και η ψήξη υπάρχει καθημερινά παντού στη ζωή μας, παίζει και επηρεάζει σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας και επηρεάζεται από διάφορα νομοθετήματα πολύ έντονα. Θα τονίσω το eco-design και την νομοθεσία ε, για την ε, οικολογική ετικέτα. Θα αγγίξω και θέματα που άκουσαν συνάδελφοι, ε, γιατί ήμουν σε αυτή τη συνάντηση στην οποία αναφέρθηκε στη Μάλτα χθε και ακούσαμε και τα σχόλια των αρχών εποπτείας αγοράς που δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικά θα ήθελα να πω. Κάτι που είναι γνωστό σε όλους, αλλά που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για να επιτύχουμε τους ενεργειακούς μας στόχους στην Ευρώπη. Έχουμε πολλά διαφορετικά νομοθετήματα για να πετύχουμε αυτή την αποδοτικότητα, αλλά αν δεν εφαρμόσετε σωστά αυτή την νομοθεσία, τότε είναι άχρηστη. Και αυτό αφορά και το, την οικολογικό σχεδιασμό και την ε, ενεργειακή ετικετοθεσία, την αποδοτικότητα των κτηρίων και πάρα πολλά, πολλούς άλλους τομείς. Επίσης, συμφωνούμε και τονίζουμε ακόμα μια φορά ότι η υποπτία της αγοράς είναι πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική για να πετύχουμε τους ε, κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μειώσουμε το χάσμα για την ε, υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και βεβαίως, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, να εξασφαλίσουμε ισότιμη ε, ανταγωνιστικότητα για τη βιομηχανία και να προωθήσουμε την αγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που μας απασχολεί πάρα πολύ. Χρειάζεται όμω να γίνουν γι' αυτό περαιτέρω βελτιώσεις. Χθε, σε αυτή τη συνάντηση στη Μάλτα, υπήρχαν 17 χώρες παρούσες και αυτές οι χώρες ε, παρουσίασαν εντυπωσιακές πληροφορίες για το πώς δουλεύουν ε, και πώς προάγουν την εποπτεία της αγοράς και είναι ε, σαφές ότι αγωνίζονται να αναγνωρίσουν αμοιβαία τα δεδομένα που παίρνουν, δηλαδή μία από την άλλη. Επίση υπάρχει έλλειψη τεχνική ε, πραγματογνωμοσύνη. Δεν μπορούμε να του κατηγορήσουμε γιατί έχουν να κάνουμε πολλά διαφορετικά προϊόντα. Ε, αν εγώ ε, δο, κάνω μία δοκιμή, α πούμε, σε ένα λαμπτήρα, δεν είναι το ίδιο με τη δοκιμή που θα κάνω, α πούμε, σε ένα μηχάνημα κλιματισμού. Δεν είναι, πολλά πρέπει να βελτιωθούν. Αυτό συνδέεται και με τα εργαστήρια που κάνουν τι πιστοποίησει και τι δοκιμέ και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δοκιμές, που δεν είναι δεν είναι ο ίδιος τρόπος, ε, δεν υπάρχουν εναρμονισμένες διαδικασίες, άρα υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Και τέλος, για τις αρχές υποπτίας της αγοράς, ε, υπάρχει το πρόγραμμα ε, για την έξυπνη Ευρώπη, προγράμματα μάλλον του παρελθόντος, ε, ε όπου ασχολούνται με την νομοθεσία των ψυγείων και η επισήμανση της ενέργειας δεν ανταποκρινόταν στα όσα, ή μάλλον έλεγε και τα α πράγμα και οι κατασκευαστές θεωρούσαν άλλο πράγμα. Ε, οι κατασκευαστές δήλωναν ότι έκανε αυτό το ψυγείο και μετά τις δοκιμές βλέπαμε ότι δεν το έκανε αυτό το ψυγείο. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι είναι η δήλωση από πλευρά του κατασκευαστή, αλλά είναι πολύ περιπλοκά αυτά τα πράγματα και δεν ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει το eco επίσης άλλο, μια άλλη πρωτοβουλία, κοινή πρωτοβουλία διαφόρων κρατών μελών που συνέρχονται και προσπαθούν να βελτιώσουν την εποπτεία της αγοράς για τις, τον, τις απαιτήσει του οικολογικού σχεδιασμού. Δηλαδή, ελάχιστε απαιτήσει για την ενεργειακή αποδοτικότητα των προϊόντων ε, διαφορετική τεχνολογία. Εξετάζουν πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αν ένα προϊόν έχει την ετικέτα και αν ο κατασκευαστής ε, δηλώνει ότι το, το προϊόν του πληρεί αυτές τις ενεργειακές προϋποθέσεις, ισχύει όντω αυτό. Ε, πώς μπορούν να το εξασφαλίσουν ε, αυτό και να το πιστοποιήσουν οι αρχές ε, εποπτείας αγοράς. Θα πρέπει να το δοκιμάσουν. Πώς θα το δοκιμάσουν αυτό το προϊόν, πώς θα το τεστάρουν, πού, πού θα βρουν τα λεφτά. Άρα πολλά πρέπει να γίνουν. Επομένω, ναι, με καλωσορίζουμε αυτή την πρόταση για την ε, εποπτεία και επιτήρηση τη αγορά. Στέλνει τα σωστά μηνύματα. Με την ευρεία έννοια. Όμω δεν λέει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει μόνο η ασφάλεια, αλλά και η περιβαλλοντική νομοθεσία και κυρίω η νομοθεσία για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θέλουμε αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει να ξεκαθαρίσουν στην νομοθεσία παντού ότι πρέπει να προωθήσουμε και την ενεργειακή αποδοτικότητα στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Επίσης, ζητάμε να αναγνωριστεί η σημασία της τεχνικής, της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατον οι αρχές εποπτείας αγοράς να κάνουν αυτό που πρέπει, γιατί δεν μπορούν να τα κάνουν όλα από μόνοι Χρειάζονται υποστήριξη και η βιομηχανία πρέπει να ενθαρρυνθεί για να δώσει αυτή την πραγματογνωμοσύνη και να είναι εταίρος σε, αυτή, σε αυτό το φόρουμ εποπτείας αγοράς που πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία τέλος και σημαντικό, ζητάμε από αυτούς που αποφασίζουν να δώσουν ένα πλαίσιο για να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας αγοράς με βάση τις εμπειρίες που έχουμε και αναγνωρίζουμε την, και θα, μας αρέσουν η ιδέα των ε, πιστοποιημένων δοκιμών ε, των εργαστηρίων Συγγνώμη, πιστοποιημένων εργαστηρίων δοκιμών και τις δημιουργίες αυτής της βάσης δεδομένων η κατάρτιση, η χρηματοδότηση, η πραγματογνωμοσύνη είναι απαραίτητα στοιχεία για να καταλαβαίνουμε μονοσήμαντα τα όσα λέει η νομοθεσία. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ σαφή παρουσίαση. Τα περιβαλλοντικά, την περιβαλλοντική διάσταση είναι καλό να την έχουμε υπόψη μας. Βλέπω ότι ο Στίβεν είναι λίγο σκεπτικιστής, ίσως λόγω έλλειψης πόρων. Αλλά βλέπετε ότι έτσι παρουσιάζονται σφαιρικά όλες οι απόψεις καθένας παρουσιάζει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Για να έχουν χρόνο οι εμπειρογνώμονε τώρα, θα ήθελα ε, οι συνάδελφοι να θέτουν στοχευμένα ερωτήματα. Θα δώσω το λόγο καταρχά στου σκιώδει ε, εισηγητέ, κύριε κυρία Πετικάνα, κυρία Σαντελμόζε, η κυρία Ρούιλερ, ο κύριο Φόξ Λίπη όμω. Και ο κύριο Κούζη. Ε, ο κύριο Κούτα, που είναι ο εισηγητή ε, τη Επιτροπή Εμπορίου για αυτή την πρόταση, τον καλωσορίζουμε. Ξέχασα να τον πω πριν, συγγνώμη. Περιμένουμε να ακούσουμε τα σχόλιά σα. Η κυρία Στάιλερ και η κυρία Ρόιτοβα. Άλλο κανεί. Βασικά όλοι όσοι είναι εδώ θέλουν να μιλήσουν. Αλλά σα παρακαλώ πολύ σύντομα. Ε, παρακαλώ. Ε, θα ήθελα στις 25 ε, να αρχίσουν οι απαντήσεις για να μην καθυστερήσουμε πολύ. Κυρία Πιέτη Κρέναν, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας. Καταρχάς θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη όσο γίνεται με ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία, τις ιδέες, τις τοποθετήσεις. Ε, θα είμαι πολύ σαφής και απερίφραστη με τις ερωτήσεις που θα σας υποβάλλω για το θέμα αυτό, διότι πιστεύω ότι η ουσία της νομοθεσίας έγινε ακριβώς στην εποπτεία, την συμμόρφωση, γιατί δεν έχουμε συστήματα, γιατί δεν έχουμε πόρους. Και η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα καλό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα ακόμη, στα οποία θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Και πολλές από τις παρατηρήσεις που έχω ακούσει από ε, συνομιλητές έχουν να κάνουν με την συμμόρφωση προϊόντων που δεν προέρχονται από τις δικές μας αγορές. Πέραν αυτού, πέραν του συστήματος πιστοποίησης δηλαδή που από ό,τι μου λένε δεν λειτουργεί, ε, τίθεται το ζήτημα ότι δεν είναι αξιόπιστο, ότι δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά πέραν αυτού τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Βλέπετε άλλες δυνατότητες δράσης για α, αύξηση των κοινών δράσεων μεταξύ κρατών μελών μέσα αυτήν την προσέγγιση που στηρίζεται στην διακινδύνευση. Ένα πιο αποτελεσματικό βεβαίω νομοθετικό πλαίσιο ασφαλώ είναι πολύ χρήσιμο και απαραίτητο. Πρέπει να πω ότι ανησυχώ όχι μόνο για τον καταναλωτή, αλλά και για τον κατασκευαστή, για τον παραγωγό, είτε του, του ενό τομέα είτε του άλλου που συμμορφώνεται και παράγει καλό προϊόν με αποτέλεσμα, με τίμημα υψηλή τιμή και τελικά αυτός δέχεται κόλαφο από την νομοθεσία και η ευρωπαϊκή βιομηχανία γενικότερα δέχεται κόλαφο από αυτήν την νομοθεσία και δεν θα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Πώς λοιπόν μπορούμε να αναπτύξουμε την νομοθεσία αυτή. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε τώρα γιατί με την, υφίστα, με την υφιστάμενη νομοθεσία έχουμε πρόβλημα και είμαστε υποχρεωμένοι να την τηρήσουμε, αλλά περαιτέρω σε περίπτωση αναθεώρησης πώς βελτιώνουμε το το νομοθετικό πλέγμα με χαμηλότερο κόστος, με πιο απλούς κανόνες, αλλά και πιο, και πιο ομοιόμορφη τήρηση. Μπορούμε να βελτιώσουμε τα συστήματα ελέγχου και αντί για τα πιστοποιητικά μπορούμε να έχουμε συστήματα ιδίας εποπτείας, ποιοτικά συστήματα που μπορούν να έχουν και που έχουν το ή για τη διαχείριση της ποιότητας οι εταιρείες, οι καλές εταιρείες. Και κάποιες πιστοποιημένες ενδεχομένω αρχές όπως εργαστήρια και μετά να υπάρχει μια τρίτη ε, πλευρά, εξωτερικός έλεγχος που θα κάνει δειγματοληπτικούς και τυχαίους ελέγχους στις διαδικασίες αυτεπόπτευσης του κατασκευαστή. Μπορεί αυτό να είναι πιο οικονομικό, πιο αποτελεσματικό. Μπορεί να φέρει καλύτερη ποιότητα και μπορεί εν τέλει να επιτρέψει την διοχέτευση των διοικητικών διαδικασιών εκεί που πράγματι εντοπίζονται οι κίνδυνοι. Σε αυτό θα ήθελα τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Κύριε Σόλτ Μόζαρ. Ευχαριστώ. Πολύ σε αυτή η ιδέα, κύριε Πιτικάρη, να την αναπτύξουμε περαιτέρω μετά. Αλλά έχω πρώτα για την Business Europe μια ερώτηση. Ίσως και για την Όργαλη. σε περίπτωση που έχουμε ένα προϊόν το οποίο συμμορφούνται, λέτε θα είναι ανοησία η αρχή να το βγάλει από την αγορά γιατί ε, με, με, επιχείρημα ότι είναι μη ασφαλές. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Ίσως να μην κατάλαβα καλά τα λόγια σας, αλλά μπορείτε να τα αναπτύξετε. Τα τέλη, το κόστος δηλαδή. Είπατε ότι αν εισαχθεί ένα σύστημα με τέλη στην υποπτία της αγοράς, ε, μπορεί αυτό να σημαίνει επιπλέον ε, επιβάρυνση οικονομική της επιχείρησης ή και του καταναλωτή. Αλλά τώρα, θα σας απαντήσω εγώ, είναι ο καταναλωτής του η αλλος επιβαρημενος εν παση περιπτωσει οταν πληρωνει ο καταναλωτής επειδη αυξηθηκε η τιμη του προϊόντος, α πληρώνει γιατί με το υψηλότερο τίμημα εξασφαλίζει κάτι καλύτερο ως προς το προϊόν που θέλει να αγοράσει. Οι αρχέ δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπουν στον πειρασμό να επιβάλλουν πρόστιμα ή τέλη μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα. Όχι, αλλά περισσότερο για να εξυπηρετήσουν το στόχο της προστασίας, φαντάζομαι. Αλλά παρακαλώ, στο ερώτημα για τον ε, φορολογούμενο, παρακαλώ να δώσετε απάντηση. Για την Business Europe, νομίζω ότι με το φόρουμ των εμπλεκομένων, στο stakeholder forum, ήσασταν ικανοποιημένοι, αλλά πείτε κάτι αν θέλετε. Κάτι ακόμη. Εντοπίζω μια αντίφαση. Η Ένωση των Επιπλοποιών θέλει σήμανση της χώρας προελεύσεως και μας λέει ότι δεν κοστίζει επιπλέον για την ευθέσιμη πληροφορίες. Η Business Europe μας λέει το αντίθετο. Θα μας δώσετε πιο πολλές εξηγήσεις. Η κυρία Ρούιλε. Θα ήθελα να φερθώ σε ένα, πρώτο, σε ένα κύριο ερώτημα το οποίο κανείς από εσά δεν έθιξε γιατί έχω μιλήσει με πολλούς ε, από τους οικονομικούς φορείς στο χώρο αυτό και οι οποίοι μου καταγγέλουν ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά σύστημα. Το ECMS αφενός και το RAPEX εφετέρου. Μπορείτε να μου πείτε ποια προβλήματα βλέπετε. Επίσης, διαγνώσκω ε, αντίφαση στα όσα είπε ο κύριος Μπέρκε για την εποπτεία στην αγορά αφενός και τη σήμανση με το ευρωπαϊκό σήμα EC αφετέρου. CE μάλλον. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς ε, τι εννοείτε. Τρίτη ερώτηση. Διεύρυνση του πεδίου. Η Άνεκ καταλαβαίνω ότι έχει ανησυχίες σε περίπτωση που διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής και περιορίζονται αντίστοιχα τα κονδύλια που τη στηρίζουν. Θα είναι περιορισμένες δυνατότητε παρέμβαση από την άλλη. Τι νόημα έχει αν εισάγονται νομοθετήματα και οδηγίες χωρίς να εφαρμόζονται σωστά. Αυτό το έχουμε δει και στην ε, ενέργεια ήδη. Πολλέ οι αλλά συμμόρφωση και ε, επιβολή της συμμόρφωσης δεν υπάρχει. Και θα ήθελα να ρωτήσω, δεν συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν θα πρέπει να, παραπλανείτε ο, να παραπλανάτε ο καταναλωτής, δηλαδή να εκδίδετε μια οδηγία η οποία τελικά δεν τηρείται και ο καταναλωτής νομίζει ότι τηρείται. Όσο δεν αφορά την επιφυλοκτικότητά σας για την πιστοποίηση από τρίτες αρχές, και τη βρίσκω βέβαια πολύ ενδιαφέρουσα την παρατήρηση της κυρίας ε, Πιετικάινεν, θα ήθελα να τη συστήσουμε λίγο περισσότερο. Ε, πάλι με δεδομένη την ε, ε, στενότητα πόρων. Λέει η Επιτροπή ότι μπορεί να γίνεται έλεγχος από μία αρχή, αυτό το είδαμε και από το impact assessment, από την αξιολόγηση των εκτόσεων. Υπάρχει η απέτηση την οποία όλοι έχουμε μπροστά μας, δηλαδή την ε, καλύτερη λειτουργία της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Και στην αξιολόγηση της, ε, του κινδύνου δεν θα πρέπει κάποια προϊόντα στα οποία βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να εκτίθενται σε αυτή την έξωθεν ε, εξέταση από την τρίτη αρχή ή να εισάγεται αυτό που είπε η κυρία Πιετικάινεν, ενώ που υφίσταται δηλαδή σύστημα διαχείριση ποιότητας να λειτουργεί αυτό στο ιστορικό της επιχείρησης και να επαληθεύεται ότι πράγματι τηρήθηκε σωστά. Για τους οικονομικούς φορείς... Είπε η κυρία Πιετικέινεν ότι θα υπάρχει πρόβλημα προς την ε, τήρηση ισότιμων ε, προδιαγραφών και ότι εκείνοι οι οποίοι τηρούν τις προδιαγραφές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Η Business Europe τι έχει να προτείνει συγκεκριμένα ώστε να εμπλακούν πιο αποφασιστικά οι οικονομικοί φορείς σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Θα ήθελα να προβλέψουμε αρκετό χρόνο για τις απαντήσεις. Γι' αυτό παρακαλώ Κύριε Κούτας, χρόνου φίδου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. First of all, thank you to all of you uh, that you allow me to address. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια στους ε, εμπειρογνώμονές σας και να τους ευχαριστήσω για τις ε, πολύ κατατοπιστικές ε, ομιλίες τους. Όπως είπατε και εσείς είμαι ο συντάκτης γνωμοδότης στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς. Ε, διεθνού εμπορίου, συγγνώμη. Οπότε όλα τα συναφή με τα εμπόριο θέματα θα τα καλύψουμε στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σφετεριστώ δικέ σα αρμοδιότητε ή να μπω στα δικά σα χωράφια. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στην Επιτροπή σα. Απλώ να κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση Το της συζήτησης που έγινε στην ακρόαση. Θα ήθελα να πω ότι όλοι οι καλεσμένοι εξέφρασαν μάλλον ικανοποίηση με τον κανονισμό και ομολογώ ότι και εγώ το ίδιο ε, ευτυχής είμαι με τον κανονισμό. Θεωρώ ότι θα ε, βελτιώσει την κατάσταση για τους καταναλωτές μας. Το θέμα είναι πόσο θα τη βελτιώσει. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ στους καλεσμένους και να τους ρωτήσω. Αν επιλέξετε μία και μόνο προτεραιότητα, αν χρειαστεί να επιλέξετε μία μόνο προτεραιότητα για τον κανονισμό, ποια θα ήταν αυτή η δική σας προτίμηση. Όπως σας είπα, ως συζητητής ε, της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου θα επικεντρωθώ σε ορισμένα θέματα. Καταρχήν, θα ζητήσω καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, μεγάλων εξαγωγικών χωρών. Για παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα ε, Συμπερίληψη του σημείου αυτού στη Μελλοντική Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Και μάλιστα αναφέρθηκε και προηγουμένως κάτι τέτοιο. Απλούστευσε των, των απαιτήσεων και η παρακολούθηση και η, η απλούστευση του ΡΑΠΕΞ ε, επίσης είναι πολύ σημαντική. Ε, Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συνεργασία και των επιπτικών αρχών, των τελωνιακών αρχών και όλων των ενδιαφερομένων. Και όπως είπε η κυρία Πιετικά, είναι η συζήτηση σχετικά με την πρόταση που μας έκανε θα είναι μάλλον ενδιαφέρουσα. Συμφωνώ με τον κύριο Βαν Μπόρεν και ο συντονισμό των κυρώσεων είναι σημαντικό θέμα. Ακόμη και αυστηρά πρόστιμα προκειμένου να έχουν κυρώσει αποτρεπτικό χαρακτήρα για τους ε, ε, εμπόρους που θέλουν να... δεν, για τους ανέντιμους εμπόρους μάλλον. Τώρα το θέμα της ε, ένδειξης προέλευσης. Ε, μέχρι τον Ιανουάριο Μέχρι... είχαμε σχετικό ψήφισμα το Ιανουάριο του 2013 για το θέμα αυτό και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σεβαστεί την ηλυμένη του απόφαση. Επίσης, είμαι υπέρ της ε, πανευρωπαϊκής ε, βάσης δεδομένων ε, για τα προϊόντα και κυρίως για τα μηχανήματα, α, για τα ατυχήματα και καλό θα ήταν να, έχουμε μια απογραφή τέτοιων ατυχημάτων σε μια βάση. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο και για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές των τραυματισμών που προκαλούνται από έλλειψη ασφάλειας προϊόντων. Το, σε ό,τι αφορά το θεμητό εμπόριο, είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε στρέβλωση ανταγωνισμού και να εξασφαλίσουμε εφαρμογή των κανόνων σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλιώς θα πρέπει να βρούμε κάποια άλλη λύση. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο το ραβδί ή το μήλο, λέει ο μιλητής. Επιβράβευση, τέλο πάντων, το κίνητρο ή το φόβητρο, αλλά είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ε, εφαρμογή του κανονισμού αυτού σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και αν έχετε συστάσεις, τις περιμένουμε με ανυπομονησία, παρά το λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Good. Well, thank you very much. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, τη δεσμευσή σας και ξέρω ότι οι συγητές ήταν πολύ ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή σας. Η κυρία Στάιλερ και η κυρία Ρόιτοβα. Σύντομα παρακαλώ, γιατί θα ήθελα να δώσω στους πέντε ομιλητές μας ε, την ευκαιρία να απαντήσουν στο σύντομα. Κύριε Στάιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομη. Πρώτο σημείο. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν συνεργάζονται τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό. Αυτό προέκυψε από τις πέντε παρουσιάσεις. Πώς θα ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτήν την προσπάθεια. Και επίσης, αυτό που είπατε και το 70% των προϊόντων που έχουν ε, ετικετοθεσία για την ενέργεια η οποία δεν είναι ακριβή. Αυτό είναι σοκαριστικό. Κύριε Ρόιτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Μία σύντομη παρουσίαση για τα ψυγεία. Φυσικά υπάρχουν ανεξάρτητες δοκιμές, το detesting. Γιατί είναι το ερώτημά μου. Οι αρχές εποπτείας αγοράς δεν μπορούν να προσφύγουν σε αυτές τις ανεξάρτητες οργανώσεις ε, για να βοηθηθούν και να ανοιχνεύσουν ε, παραπλανητική διαφήμιση ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες που δίνουν οι κατασκευαστές. Ε, το βασικό είναι να είμαστε συνεπείς όταν επιβάλλουμε κυρώσεις και να επιβάλλουμε κυρώσεις όταν υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ε, τώρα, να δώσω το λόγο ε, από τον τελευταίο εμπειρογνώμονα. Ε, μπορούμε να κάνουμε μια υπέρβαση του χρονοδιαγραμματός μας, του, της προθεσμίας που έχουμε στις 12.30, κατά 5 λεφτά όχι παρα, παραπάνω όμως. Ε, ξεκινάμε την τελευταία ομιλήτρια, την κυρία Βόιτ, και θα συνεχίσουμε τους υπόλοιπους. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Ε, θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σε δύο λεφτά. Καταρχάς για την πιστοποίηση και το σήμα CE έχει νόημα μόνο αν υπάρχει πραγματική εποπτεία της αγοράς και συνεργασία μεταξύ των αρχών. Γιατί οποιοδήποτε σήμα, είτε ευρωπαϊκό είτε οποιοδήποτε άλλο, είναι άχρηστο εάν κάνετε τζεκάρι τι υπάρχει πίσω από αυτό. Δεύτερον, να σας δώσω ένα παράδειγμα από τις ΗΠΑ, από τον κλάδο δικό μας, που είναι μια, μια μεγάλη οργάνωση που κάνει τις δοκιμές και τα αποτελέσματα αυτά τα δίνει ε, στο Υπουργείο ενέργεια για την ενεργειακή ε, αποδοτικότητα και μπορεί το Υπουργείο να χρησιμοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα αν θέλει. Και αν θέλει μπορεί να κάνει επιπλέον δοκιμέ μετά, να αμφισβητήσει αυτέ τι δοκιμέ. Εν πάση περιπτώσει έχουν ένα σημείο θετηρία, έχει το Υπουργείο δηλαδή Ενέργειας, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αν υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε την κατάσταση αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το παράδειγμα και πρέπει να το κοιτάξουμε. Ίσως να υπάρχουν κάποια ζητήματα που μπορούμε να κοιτάξουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς τα πιστοποιημένα εργαστήρια δοκιμών και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που έχουν στο ιστορικό τους οι εταιρείε, θα κοιτάξουμε τον οικολογικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική χρήση ενέργειας, όλα στηρίζονται στις ε, δηλώσει, στην αυτοπιστοποίηση δηλαδή του παραγωγού. Βεβαίως μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα και να εισαγάγουμε και άλλα συστήματα ή τμήματα συστημάτων ε, ως προς την πιστοποίηση που ήδη υπάρχουν και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος. Υπάρχει ωστόσο ένα πρόγραμμα Atletin, το οποίο ήταν ε, ένα, μια πρωτοβουλία της ΣΥΣΕΤ e με αποτελέσματα διαθέσιμα δημόσια, αλλά αν θέλετε μπορεί να σας τα βρω και να σας τα στείλω. Και υπάρχει και μια δεύτερη φάση αυτού του προγράμματος του Ακλητ. Σε εξέλιξη, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που τηρήσετε και το χρόνο σας, κυρία Σλάιερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στα, ε, την περισσότερη πιστοποίηση και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Όλα αυτά προηγούνται τη θέση εμπορία. Το τι σημαίνει αργότερα από τη στιγμή που θα τεθεί ένα προϊόν στην αγορά σε εμπορία είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Γιατί και στη συνέχεια μπορεί να συμμορφωθεί. Ακόμη και στην αρχή δεν είναι συμβατό το προϊόν και αυτό το εξασφαλίζει η υποπτή της αγοράς. Η συνεργασία και η συλλογή πληροφοριών και ανταλλαγή εμπειριών είναι πολύ χρήσιμη με τα εργαλεία που μας δίνει ο κανονισμός και που ήδη βρίσκονται στο 6, 768, ε, στον κανονισμό 765, συγγνώμη. Ε, επίσης, ε, η υπάρχει ε, εξαίρεση ορισμένων προϊόντων. Ε, βέβαια, στην... η εμπειρία αυτή ήταν σχετικά επιτυχημένη στο παρελθόν. Για το RAPEX, το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων. Υπάρχει στο έγγραφο με τις θέσεις μας, δεν το αναφέραμε ρητά. Θα θέλαμε το RAPEX να είναι σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και για το σοβαρό κίνδυνο και να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο από τις αρχές εποπτής αγοράς για να μπορούν να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες και τις εμπειρίες τους. Κατά τη γνώμη μας αυτός είναι ο σκοπός ενός τέτοιου εργαλείου. Και την ένδειξη της προέλευσης. Γιατί φαντάζομαι ότι Business Europe δεν μπορεί να πει πολλά γι' αυτό. Υπάρχει όντως μια αντίφαση αυτό εξαιτία των προϊόντων που εκπροσωπεί ο κάθε κλάδο. Εμεί εκπροσωπούμε πολύ περίπλοκα προϊόντα για τα οποία είναι δύσκολο να αναφέρεται η ένδειξη προέλευση κάθε τμήματο, κάθε μέρο. Και ο λόγος που δίνεται, ε, το επιχείρημα που δίνεται για την αναφορά της προέλευσης είναι η χνηλασιμότητα, αλλά αυτό δεν, για μας ε, δεν εξασφαλίζει καμία περίπτωση, δεν συμβάλλει στην ε, χνηλασιμότητα η ένδειξη της προέλευσης. Ο κύριος Βάντεν Μπρακ. Η κυρία Σοντεμόζε είπε τι γίνεται με τα σήματα προέλευσης και γιατί είμαστε εμείς κατά. Όχι, δεν είμαστε κατά. Πολλά κράτη, ε, πολλοί συμμετέχοντες είναι κατά, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι υπέρ. Για τα τέλη. Η Business Europe είναι υπέρ των τελών. Δηλαδή, υπο, κυρώσει υπομορφή τελών. Αλλά υπό τον όρο ότι θα μας οδηγήσει στο να στο, στο εξής αποτέλεσμα. Οι φταίχτε να ε, πληρώσουν το τίμημα. Δεν θέλουμε το κόστος ε, να καταμεριθεί ισότιμα σε όλες τις επιχειρήσεις. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Θα πρέπει οι καλοί παίχτες, οι καλές επιχειρήσεις να μην τιμωρηθούν και δεν θα πρέπει να φέρουν το τμήμα του βάρους. Τώρα, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να φύγουν από την αγορά. Οι αρχές πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα αλλά θα πρέπει να είναι υλικό μη συμμορφούμενο που να, που να μετράει. Όχι για κάθε εξάρτημα. Παραδείγματο χάρη έχουμε, ε, έχουμε καλώδια τα οποία δεν είναι ασφαλή γιατί δεν υπάρχει αρκετός χαλκός. Ε, αυτά προκαλούν φωτιές και καίγονται σπίτια εξαιτία αυτού. Αυτό είναι πρόβλημα. Τώρα για τα συστήματα εξασφάλισης ποιότητας είναι ένα ε, μέτρο πριν τη θέση στην αγορά, συμφωνώ με αυτό και μπορεί να παραποιηθεί, όντως. Το πρόβλημα είναι ότι θα τεθεί ξανά, υπάρχει κίνδυνος να τεθεί ξανά ε, βάρος σε καλόπιστους παίχτες. Παραδείγματος χάρη, ένα τμήμα της ε, Philips έχει έχει ένα τμήμα των επιχειρήσεών της στην Ολλανδία και η Ολλανδία εμπιστεύεται τη Philips για αυτά που κάνει. Ε, και η χώρα όταν έχει εμπιστοσύνη σε μια εταιρεία μπορεί να την ελέγχει λιγότερο. Είναι ένα σύστημα που μπορούμε να το διερευνήσουμε αυτό. Επίσης πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τους προμηθευτές στην ε, διαδικασία. Ε, ξέρουν πολύ, πάρα πολλά το, από αυτά που συμβαίνουν στην αγορά οι προμηθευτές, αλλά συχνά ε, διστάζουν να καταγγείλουν ας πούμε, άλλους ε, στις αρχές, ε, γιατί φοβούνται ότι αυτό δεν είναι σωστό για τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ κύριε Σορμπούρεν. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλή ειδή αυτό που είπατε, διότι πολλές είναι πληροφορίες ε, που θα χρειαστούν και μόνο 0,001% θα, κάνει ε, θα τηρήσει αυτό που χρειάζεται για να έχουμε ασφαλή προϊόντα για τη ράπεξ. Και η ISIS μες μπορεί να ε, καταστραφεί από, τα, την πληθώρα των δεδομένων που θα κυκλοφορήσουν. 80% των επιθεωρήσεων τώρα, από αυτές που αναλαμβάνει η δική μου οργάνωση, είναι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μόνο 20% έχουν να κάνουν με επαλήθευση προϊόντων. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε επαλήθευση φακέλων εάν υπάρχει λόγος. Η απουσία πόρων. Η εποπτεία στα μη τρόφιμα βέβαια έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με την εποπτεία στον χώρο των τροφίμων. Πολύ μεγάλο περιθώριο υπάρχει ως εκ τούτου για εποπτεία ε, εκτός τροφίμων. Αλλά στα προϊόντα τα καταναλωτικά έχουμε από τη Γενική Διεύθυνση για το Καταναλωτή και την Δημόσια Υγεία στήριξη. Και έτσι μπορούμε να έχουμε εναρμονισμένα προϊόντα, την οποία θα μπορούσε και η Γενική Διεύθυνση για τις επιχειρήσεις να υποστηρίξει. Πρέπει λοιπόν να το συστήσουμε αυτό και με την Επιτροπή. Η αποτελεσματικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για να δούμε πώς μπορούμε να τηρήσουμε τη στρατηγική και να ενημερώσουμε, να καταρτήσουμε τους επιθεωρητές και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τη βιομηχανία και για τα εναρμονισμένα προϊόντα. Αυτά νομίζω με τα φτωχά αγγλικά μου. Ευχαριστώ. Εν τέλει ο κύριος Ράσελ. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Δεν ήθελα εγώ να παίξω το ρόλο της Κασάνδρας στην παρουσίασή μου. Βεβαίως και θέλουμε την εποπτεία της αγοράς και, τη σχετική, και το σχετικό κανονισμό, αλλά με, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Δεν τηρείται σε όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, γιατί πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Πρέπει λοιπόν και να γίνει σεβαστή η εθνική αρμοδιότητα, αλλά και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και έτσι Crystal, ναι, ε, είμαστε υπέρ του φόρουμ. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται για κοινούς ορισμούς, για κοινέ δράσεις στην κοινότητα, σε συνεταιρική σχέση με τους διαφορούς παράγοντες αγορές, της αγοράς, αλλά πρέπει να βρεθούν και οι πόροι, το πώς θα ρεμένει Δεν νομίζω ότι μπορεί μια οργάνωση καταναλωτών να δώσει απάντηση σε αυτό. Έχουμε απευθύνει κάποιες προτάσεις ε, με ιδέες για διαρθρωτικά ταμεία που, παραδείγματι, θα μπορούσαν να απελευθερωθούν για χώρες που έχουν μεγάλα, έχουν εκτεταμένα γεωγραφικά σύνορα. Ασφαλώς θα μπορούν να υπάρχουν και άλλες ε, λύσεις. Η περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά κάθε τύπου νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα βέβαια, αλλά η ασφάλεια πάνω απ' όλα. δεν με ενδιαφέρει τόσο να έχω ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ το οποίο θα είναι περιβαλλοντικά, θα είναι οικολογικό αλλά επικίνδυνο. Προτιμώ να είναι ασφαλές. Τρίτη, ε, τρίτες αρχές πιστοποίησης της ε, ασφάλειας δεν μπορεί να είναι αυτοπανάκια γιατί μόνο σε προϊόντα που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο που, ή όπου έχουν εντοπιστεί δυσκολίες στην εποπτεία μπορεί να έχουν ε, ε, χρησιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πραγματογνωμοσύνη σας. Μας έχετε βοηθήσει πολύ. Και δύο λόγια για να κλείσουμε εν συντομία για να απελευθερώσω τους διερμηνείς σε μερικά λεπτά μόνο. Κυρία Πιέτη Κάινεν και κυρία Σάλτε Μόζερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλια, πολύ επικοδομητική συζήτηση. Κλείνουμε, Μαρία. Και ως και η φαντάζομαι, θέλουμε να συνεχίσουμε την συνεργασία και αν βρούμε και άλλες μεθόδους χρήσιμες, ε, αποτελεσματικές, οικονομικές για τη βελτίωση του συστήματος. Ξέρετε, όταν κάθεται ο κόσμος να μιλήσει και να βρει κοινέ λύσει, ασφαλώ θα τα καταφέρει γι' αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Κυρία Σόλτα Μόζερ, Σα ευχαριστώ και εγώ για τι καλέ σα παρεμβάσει, για τη συμμετοχή στη συζήτηση, πολύ σημαντική για το πακέτο για την ασφάλεια των προϊόντων. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σε περισσότερε λεπτομέρειε ε, και για την ασφάλεια των προϊόντων. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπώ. Uh, uh, και εγώ, λέει ο ευχαριστώ τους πάντες και ελπίζω να μας παρακολούθησαν αρκετοί και μάλιστα από το χώρο της εποπτείας, των προδιαγραφών, ε, της στήριξης των προδιαγραφών από τις επιχειρήσεις. Με χαρά παρακολουθήσαμε ό,τι είχατε να μας πείτε σήμερα. Αυτό το νόημα άλλωστε είχε και συνεδρίαση. η δημοκρατική δηλαδή συμβολή η δική σας στην διαδικασία να Οι εισηγητέ για τα πρακτικά 11 Ιουνίου θέλουν τι τροπολογίε για μετάφραση. 8 ή 9 Ιουλίου πρώτη εξέταση. Προθεσμία 4 Σεπτεμβρίου για τι τροπολογίε, τι οποίε θα εξετάσουμε μαζί με τι συμβαστικέ για να ψηφίσουμε, το Σεπτέμβριο για να ψηφίσουμε στις 17 Οκτωβρίου. Ξέρω ότι είναι στενά τα φωνικά περιθώρια. Αλλά θα συμφωνήσετε πιστεύω και ασφαλώς συμφωνούν και οι δικοί μα ότι πρέπει οι διαπραγματεύσει με τα κράτη-μέλη να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό και πριν να ε, λήξει η θητεία του Κοινοβουλίου. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές και δεν θέλουμε να πέσει σε μια μαύρη τρύπα ανάμεσα σε, ε, στο τωρινό και το επόμενο μετά τις Ευρωεκλογέ Κοινοβούλιο. Έχουμε πολλή δουλειά, ούτω ή άλλως αυτό δεν θα είναι το τέρμα. Ε, έχουμε πάρα πολλά σημαντικά νομοθετικά ζητήματα και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, ό,τι πόρους έχουμε διαθέσιμο θα τους αφιερώσουμε σε αυτό το έργο. Σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Πέρα συνεδριάσεις προς το παρόν έως τις 3, όπου έχουμε κάποια άλλα θέματα να συζητήσουμε.